non, Possiamo allora aprire i nostri lavori. Καλημέρα, μπορούμε να αρχίσουμε τις εργασίες μας. Σας υπενθυμίζω πρώτα απ' όλα ότι ε, θα ήθελα να σας ε, συστήσω Ε, μάλλον να σας ε, πω ότι ε, η συνεδρίασή μας μεταδίδεται απευθείας από το διαδίκτυο. Δηλαδή είναι δημόσια, μας ακούν, μας βλέπουν εκτός της αίθουσας και από όλα τα γραφεία του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι δημόσια ακρόαση, άκρος σημαντική. Και θα μας επιτρέψει να συζητήσουμε για μια καλύτερη μελλοντική ε, αρχιτεκτονική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λυπούμε ε, για την ισχνή παρουσία εδώ του κοινού. Ευχαριστώ τους εισηγητές, αλλά σας υπενθυμίζω και τονίζω ότι μας παρακολουθούν και στα γραφεία του Κοινοβουλίου, αλλά και εκτός. Και θα πρέπει ε, να ξέρετε ότι για αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα θα συμπεριληφθούν στην έκθεση των εισηγητών μας και θα ζητηθούν στην Ολομέλεια. Έχετε την ευκαιρία παρόντες να κάνετε ερωτήσεις, ε, υποδείξεις, ε, προτάσεις. Η πρώτη πρωινή συνεδρίαση από τις 9 μέχρι μάλλον συγγνώμη, από τις 9 και 4 μέχρι τις 11.30 περίπου, αφορά την ευελιξία και τη διαφοροποίηση στην ενοποίηση υπό τη συνθήκη της Λισαβόνας και νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε αμέσως δίνοντας το λόγο στους εισηγητές. Ε, πρώτα, ε, στον κύριο Γκολτιέρη και στον κύριο Τσαρκόφσκι. Ποιος θέλει το λόγο πρώτος, ο κύριος Γκολτιέρη ίσως. Thank you. Κύριε κύριος Γκουαλτιέρη, σας ευχαριστώ στα αγγλικά. Ε, κυρίως τους ομιλητές ευχαριστώ. Ε, πρέπει να σας πω ότι και για μένα και για το Ράφαλ είναι τιμή όσο και ε, προνόμιο να σας έχουμε ενώπιόν μας. Σας διαβάζουμε και τώρα σας βλέπουμε και όλες και έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την εργασία μας. για το σχέδιο πρώτα έκθεσης για τα συνταγματικά στοιχεία της ε, διακυβέρνησης πολλαπλών ταχυτήτων. Δεν έχει ακόμα εκπονηθεί ούτε καν το σχέδιο έκθεσης, αλλά αυτό το σεμινάριο βεβαίως θα είναι και πάρα πολύ χρήσιμο και για τα υπόλοιπα θέματα που μας απασχολούν στο Κοινοβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουμε στο εγχείρημα αυτό ε, που ε, ξεκίνησε στο Συμβούλιο. Γνωμοδοτούμε και για την έκθεση Tyson που είναι έκθεση πρωτοβουλίας με βάση το άρθρο 50 ε, για τη γνήσια οικονομική και νομισματική ένωση και στο Κοινοβούλιο και εγώ συμμετέχουμε ως ΣΕΡΠΑ ε, στη διαβούλευση με τον κύριο Βαν Ρόμπεϊ. Η ομάδα λοιπόν των ΣΕΡΠΑ έχει ε, συντάξει ένα σύντομο έγγραφο ως πρώτη αντίδραση στο έγγραφο θέσεων που γκρίθηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων την περασμένη Τρίτη και ελπίζω να σας διανεμηθεί. Ο Ζαν Βικτόρ Λουί μας έστειλε μια περίληψη ε, για το τι είναι φυκτό βραχυπρόθεσμα και επιθυμητό μέσο πρόθεσμα θα πρέπει να βασίζεται ε, σε μια ευρύτερη θεώρηση συνταγματικής φύσεως. Ε, αυτή τη θεώρηση θα πρέπει να την ορίσουμε και το θεσμικό πλαίσιο και η ε, αιτία της κρίσης αλλά και τα διλήμματα από πλευρά συνταγματικής πρέπει να αντιμετωπιστούν για να βρεθεί μια αποτελεσματική λύση στην κρίση. Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι από το 2010 και μετά η κρίση ήρθε να ενισχύσει την ολοκλήρωση της Ένωσης και των χωρών της. Μέχρι τώρα όμως ο δρόμος που έχει επιλεγεί ε, έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι αποτελεσματικός, ενώ ε, ε, ταυτόχρονα διευρύνει και το δημοκρατικό έλλειμμα. Το μοντέλο αυτό βασίζεται κυρίως σε ένα αντάλλαγμα δημιουργείται ένας ε, μηχανισμός σταθερότητας διακυβερνητικός ε, που χρηματοδοτούν τα κράτη-μέλη και υπάρχει πολύ μεγάλη ε, ρεσιμότητα και το αντάλλαγμα είναι πιο ισχυροί δημοσιονομικοί κανόνες και πιο δεσμευτικοί. Όπως είπε και ο Μαντούρο, αυτό το σύστημα που βασίζεται στις εθνικές δημοκρατίες δεν λειτουργεί αποτελεσματικά διότι υπάρχει μια μη βιώσιμη αντιφατική ε, διάσταση, μια αντίφαση μεταξύ των εθνικών πολιτικών και της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής. Ε, στην απάντηση που δίνει το έγγραφο θέσεων προσπαθούμε να δώσουμε ένα όραμα ε, που να βασίζεται σε μια πιο σαφή διάκριση των ρόλων, ε, των λειτουργιών και των πόρων μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών που διαχειρίζονται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με μια ευρωπαϊκή ε, χρηματοδότηση αφενός και αφετέρου τους εθνικούς πόρους και τις εθνικές δημοκρατίες. αυτή η θεώρηση που είναι αμυγός ομοσπονδιακή, παρόλο που είναι περιορισμένες οι αρμοδιότητες και εξουσίες σε ομοσπονδιακό επίπεδο, απαιτεί ε, τα θεσμικά όργανα να διαχειρίζονται ε, την ΟΝΕ, ε, αλλά και τις αντίστοιχες ασυμμετρίες μεταξύ ΟΝΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίθεται και το θέμα των αρμοδιοτήτων, των εξουσιών και των διαδικασιών όπως ορίζονται από τις συνθήκες. Ε, υπό την έννοια αυτή η δική μας προσέγγιση είναι σαφής. Τι πιστεύουμε εμείς ότι πρώτον οι παρούσες συνθήκες παρέχουν όλα τα απαραίτητα εκείνα εργαλεία ε, για να καθορίσουμε το πλαίσιο αυτής της γνήσιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Και επίσης τονίζουμε και τις δυνατότητες του άρθρου 136 ενισχυμένης συνεργασίας αλλά και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τη ρήτρα ευελιξία του άρθρου 352 σε συνδυασμό με το άρθρο 136 για την ενισχυμένη συνεργασία το 20. Δηλαδή ε, να χρειάζεται ομοφωνία μόνο μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης ή εκείνων των χωρών που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία. Δεύτερον, με τις παρούσες συνθήκες όχι μόνο μπορεί να υπάρξει ένας εκ των προτέρων οικονομικός και δημοσιονομικός συντονισμός, αλλά και πάλι με το παρόν πλαίσιο των συνθήκων και βέβαια αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε, να το ψηφίσουμε, να το αποφασίσουμε γιατί δεν είναι ακόμα κοινή θέση του Κοινοβουλίου, παρόλο που κάπου εκεί ε, κινείται το έγγραφο του ΣΕΡΠΑ, να έχουμε ένα μηχανισμό για τους ιδίους πόρους και τον προϋπολογισμό πολλαπλών ταχυτήτων στο παρόν δημοσιονομικό και θεσμικό πλαίσιο. Αυτό το Ταμείο της Ευρωζώνης, ας πούμε, που συζητείτε τώρα, γνωρίζετε τη γαλλική και τη γερμανική πρόταση, δεν είναι κάτι που γράφεται εκτός του κοινοτικού προϋπολογισμού και να ε, ε, είναι κάτι το οποίο θεωρείται αυτόματο σταθεροποιητής από εθνικούς οικονομικούς πόρους. Ε, δεν είναι αυτόματο κάτι τέτοιο και πάλι θα πρέπει να το συζητήσουμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να εξετάσουμε την ανάγκη τροποποίηση των συνθηκών για να συμπληρωθεί η αρχιτεκτονική της γνήσιας ΟΝΕ. Για λόγους όμως και πολιτικούς, όχι μόνο θεσμικούς. Φρονώ προσωπικά ότι ο μόνος τρόπος να γίνει ε, δυνατή η προοπτική της αναθεώρησης είναι να μην είναι αυτή η αφετηρία αλλά να ενισχύσουμε την ΟΝΕ, να ε, αναφέρουμε την ισορροπία προς μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση χρησιμοποιώντας τα εφιστάμενα μέσα και εργαλεία και να ε, κάνουμε μια μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση. Οι επόμενε ευρωεκλογέ να είναι μια ευρωεκλογέ που να βασίζονται σε ένα ευρωπαϊκό πολιτικό χώρο και οι πολίτε να επιλέγουν ε, όχι μόνο το Ευρωβουλευτή τους, αλλά και την κυβέρνησή τους. Βλέπει Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση πολιτική συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης χρειάζεται και μια νομιμοποίηση για επόμενα βήματα εκχώρησης αρμοδιοτήτων και εξουσιών. Δεύτερον, απορρίπτουμε πλήρως και νομίζω θα χρειαστεί συζήτηση το επιχείρημα που λέγει ότι υποτίθεται ότι δεν έχει νομιμοποίηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω της ασυμμετρίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης και των υπολείπων μελών της Ένωσης. Μα αυτή η ασυμμετρία προβλέπεται και μάλιστα ρητά στις συνθήκες. Όχι μόνο μεταξύ διαφόρων ειδών νομιμοποίησης Κοινοβουλίου και Συμβουλίου αλλά και για τις διαδικασίες που ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί. Και αναφέρομαι στο άρθρο 136 σε συνδυασμό ε, με το 121.6. Είναι πολύ σημαντική η νομοθεσία που έχει βασιστεί και πολύ αποτελεσματική για τις χώρες Ευρωζώνης με μια αποφασιστική ψηφοφορία ε, στο Κοινοβούλιο Ευρωβουλευτών που δεν είναι από χώρες του Ευρώ. Και ουδής ήρθε να αμφισβητήσει ε, ας πούμε την ισχύ των ε, όσων ψηφίσαμε στη δέσμη 6 οδηγιών. Βεβαίως η δημοκρατία δεν είναι ποτέ τέλεια. Το θέμα είναι τώρα να κοιτάξουμε και να εξετάσουμε και τα προβλήματα των εναλλακτικών λύσεων. Ας πούμε, ε, για να Αναφέρω τα όσα λέει ο Ζων Κλοντ Πυρή, μια ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία εθνικών κοινοβουλίων. Δεν θεωρώ ότι είναι βιώσιμη εναλλακτική λύση. Ένα τέτοιο σώμα δεν θα είχε καμία νομοθετική εξουσία και αρμοδιότητα. Δεν θα μπορούσε, ας πούμε, ε, να δημοσιευθεί τίποτα στην επίσημη εφημερίδα. Θα ήταν απλώ μια λέσχη συζητήσεων. και δεν θα υπάρχει και αναλογική εκπροσώπηση ούτε με όρους πολιτικούς ούτε με όρους εθνικούς εκτός και αν φτιάξουμε κανένα τεράστιο ε, σώμα. Γιατί είναι πιο νομιμοποιημένο ένα όργανο που έχει ίσο αριθμό μελών από τη Γερμανία και από τη Μάλτα, ας πούμε. Ε, ενώ ε, δεν θα ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συμμετέχουν ευρωβουλευτές χωρών που δεν είναι στο ευρώ. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε συμφωνίες κυρίων. Και ήδη τις κάνουμε για τις προτεραιότητες σε θέματα του ευρώ, ε, συντονιστές, εισηγητές, ε, προς τους βουλευτές της, ε, των χωρών της Ευρωζώνης. Και αυτό μπορεί να ενισχυθεί ακόμα. Είναι να ενισχυθεί και η διάσταση των κοινοβουλευτικών πολιτικών ομάδων. Ας πούμε, οι κατάλογοι ψηφοφορία που καταρτίζονται από τις πολιτικές ομάδες δεν είναι των εθνικών αντιπροσωπιών, είναι εγκάρσει, οριζόντιε, σαν πολιτική ομάδα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια θέματα ε, που μας ενδιαφέρουν πολύ, που τα υποστηρίζουμε. Είμαστε κατά μιας ε, διακυβερνητικής συνθήκης, θέλουμε να εργαστούμε στο ε, πλαίσιο των υφισταμένων συνθήκων ε, βλέπουμε τα προβλήματα βέβαια, τις αντιφάσεις, τα διλήμματα. Να δούμε ποια θα είναι η βάση λοιπόν της έκθεσής μας και γι' αυτό το λόγο σας καλέσαμε να συζητήσετε μαζί μας, να ανταλλάξουμε απόψεις, να μας δώσετε τα φώτα σας. Εμείς είμαστε απλοί πολιτικοί. Χρειαζόμαστε ε, σοβαρή συζήτηση με τους πιο σημαντικούς ε, συνταγματολόγους και εμπειρογνώμονες. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε και θα δώσω το λόγο στον Ράφα. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Γουαλτιέρη. Κύριε Τσαρκόφσκι. I will be very brief because we will have... Θα είμαι πολύ λακωνικός γιατί θα έχουμε αρκετή ευκαιρία να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες του θέματος αυτού στη διάρκεια των συζητήσεων των πάνελ. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή ε, που σας έχουμε όλους εδώ. Έχω και μερικούς από τους καθηγητές μου στο Κολέγιο της Ευρώπης και είναι πολύ ενδιαφέρον που θα συζητήσουμε εδώ όλοι μαζί αυτό το επίκαιρο θέμα και που θα ξεκινήσουμε ε, μία συζήτηση που μερικές φορές είναι δύσκολο ιδιαίτερα για έναν Ευρωβουλευτή από μια νέα χώρα μέλος που δεν ανήκει στην Ευρωζώνη. Γιατί όταν εξετάζουμε διάφορες συνταγές ε, για το μέλλον της Ευρώπης, μερικές φορές ε, μου στερούν την ομοποίηση για τρεις ε, λόγους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσω να ε, εμείνω στο ρόλο μου. Πάντως, διαπραγματευόμαστε και το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Και μάλιστα στις συζητήσεις που έχουμε με τους ΣΕΡΠΑ, που μας ε, εκπροσωπούν στις συζητήσεις ε, με τον Βανερόν Πόη, ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά, αλλά δεν θέλουμε η συζήτηση να έχει μόνο ακαδημαϊκό χαρακτήρα, γιατί μερικές φορές η Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντιμετωπίζεται ως ε, think tank. Αλλά μας ενδιαφέρουν οι συζητήσεις με στόχο την ανέβρεση πρακτικών λύσεων. Και όταν εννοώ ότι χρειαζόμαστε μια ειλικρινή συζήτηση, όταν λέω κάτι τέτοιο το εννοώ, γιατί μερικοί θεωρούν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι πηγή νομιμοποίηση. Αν κάποιο το πιστεύει, θα πρέπει να το πει ειλικρινά και να το συζητήσουμε. Ο Ζαν Κλοντ είπε σε ένα βιβλίο του ότι μια σχετική αποτυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και μάλιστα το relative, το σχετική αποτυχία, το, ε, το πρόσθεση για λόγους πολιτικής ορθότητας. Να το συζητήσουμε λοιπόν και αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι ε, αμφισβητείται όχι μόνο ε, η νομοποίησή μας ως προς την ε, συμμετοχή στη συζήτηση, αλλά και προς τα αποτελέσματα. Ε, πάντως τουλάχιστον να έχουμε κάποια αποτελέσματα, ακόμη και αν δεν θεωρούν οι πολύ σχολαστικοί ότι δεν υπάρχει πλήρης νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν όμως προβλήματα αποτελέσματος, παραγωγής αποτελέσματος και αυτό το βλέπει και η κοινή γνώμη. Οπότε θα πρέπει να αναλύσουμε τα επιτεύγματά μας, να αναλύσουμε τις ε, απόψεις και τις διεκδικήσεις μας και να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Γιατί επικεντρωνόμαστε σε θεσμικές αλλαγές, προσπαθούμε ε, να προβάλλουμε ε, και να πείσουμε τον κόσμο για την συνθήκη της Λισαβόνας και για τη συνέχεια της, αλλά μερικές φορές φαίνεται ότι επιμένουμε στα σημεία που δεν είναι τα πιο σημαντικά, όπως α, ε, ε, μας έχουν αποδείξει οι εξελίξεις, γιατί είχαμε όντω μερικές σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μερικές από αυτές ε, όμως δημιουργήσαν προβλήματα. Αυτό διαπιστώσαμε με την εφαρμογή κάποιων διατάξεων και τη σύγκρουση αρμοδιοτήτων που απέρευσε από αυτές. Πάντως οι πραγματικά απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπίσουμε την κρίση ιδιαίτερα σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο και οικονομία δεν φαίνεται να έλαβαν χώρα. Προσπαθούμε λοιπόν να εγγύψουμε πιο διεξοδικά σε αυτά τα θέματα και το σημείο κίνησης και το δικό μου και του Ρομπέρτο αλλά και ε, η σύμφωνη γνώμη των συναδέλφων στην Επιτροπή είναι ότι θέλουμε να προσπίσουμε την μοναδικότητα του ευρωπαϊκού σχεδίου. Αντιλαμβάνομαι ότι μερικοί ε, μίλησαν για τη θεσμική ανοχή και νομίζω ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι ότι είναι προαιρετική αυτή η αποδοχή της υπαγωγής στο ευρωπαϊκό σχέδιο και αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της ε, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Βέβαια, στα χαρτιά υπάρχουν ε, πολλέ λύσει. Ο φεντεραλισμό είναι πιο συνεχή, η επαναφορά στο παρελθόν με τη δημιουργία μια ένωση εντό τη ένωση. Και να αντιμετωπίσουμε κάποια νοσταλγία τον παλιό καλό καιρό που ήμασταν πιο συνεπείς, για να σα πω την αλήθεια, εσείς ήσασταν πιο συνεπείς. Δεν πιστεύουμε όμως ότι τέτοιες λύσεις τη σήμερα ημέρα τουλάχιστον είναι δόκιμες ε, ή άμεσης ε, εφαρμογής. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπίσουμε τα μέχρι τώρα επιτεύγματά μας και πρώτα απ' όλα να προσπίσουμε την ακαιρεότητα του ευρωπαϊκού σχεδίου και των ευρωπαϊκών ε, θεσμικών οργάνων. Και το θέμα είναι πόσο ριζοσπαστικοί πρέπει να είμαστε. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή, αυτή τη σύγχυση που δημιουργείται γύρω μας. Ε, μπορούμε να το καταφέρουμε με περιορισμένες ε, αλλαγές στη συνθήκη, όπως προβληματίστηκε και ο Ρομπέρτο. Πάντως θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε να επιτεθούμε στην, να πλήξουμε την ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ή μήπως θα πρέπει να αναζητήσουμε ακόμη και από τώρα κάποιες πιο ριζοσπαστικές λύσεις όπως προτείνει ο Ζαγκλώτ Πύρης ε, στο βιβλίο του. Και στην πορεία της συζήτησης θα προσπαθήσω να καταρρύψω μερικά από τα επιχειρήματα αυτά, αλλά αυτό θα φανεί στη συζήτηση. Έχουμε αρκετά δύσκολα θέματα λοιπόν μπροστά μας. Έχουμε ολόκληρη τη μέρα στη διάθεσή μας για να επισέλθουμε σε όλα αυτά τα επιμέρους θέματα και σας ε, διαβεβαιώ ότι θα σας ακούσουμε με ιδιαίτερη προσοχή ε, δεν το συνηθίζουν αυτό οι πολιτικοί να ακούν, αλλά πραγματικά με ενδιαφέρει μια μεστή συζήτηση και τεκμηριωμένη, ώστε να καταλήξουμε σε έγγραφα που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο στο, εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και γενικώ στη συζήτηση για το μέλλον της ΟΝΕ και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ζαρκόφσκι. Και τώρα θα αρχίσουμε να ακούμε τους ειδικού μας που είναι όλοι υψηλότερο του επίπεδου και για τους οποίους ήδη ευχαρίστησα στην αρχή της συνεδρίασης. Σας ευχαριστώ για αυτή την επιλογή και για τη γραμματεία μας ε, για τη διοργάνωση αυτού του σεμιναρίου. Πριν να δώσω το λόγο θα πρέπει να διευκρινίσω ότι επειδή πρέπει να σας ακούσουμε και να δώσουμε και το λόγο στους συναδέλφους που είναι παρόντες ε, θα σας καλέσω να διατηρήσετε τις παρεμβάσεις σας εντός 15 λεπτών. Ε, δεν είναι και πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει 15 λεπτά θα πρέπει να αρκούν. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο πρώτα στον κύριο Ζαν Βικτόρ Λουίς που είναι καθηγητής του Ελευθέρου Πανεπιστημίου των Βρυξελών. Και παρακαλώ να έρθετε εδώ στο έδρανο της Προεδρίας. Ο κάθε ομιλητής μπορεί να διαλέξει αν θέλει να καθίσει στη θέση του ή να έρθει εδώ στο έδρανο της Προεδρίας. Il tema che è stato indicato è quello dei dilemmi istituzionali che l'Unione Το θέμα είναι ε, ε, αυτό, τα, τα θεσμικά διλήμματα που προκύπτουν λόγω της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Παρακαλώ, καθίστε. Mr. Αγγλικά θα μιλήσω, τουλάχιστον να προσπαθήσω. Μου ζήτησαν να σας πω ε, τι πιστεύω για τα θεσμικά διλήμματα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Μερικά από αυτά τα διλήμματα ήδη τα παρουσίασαν οι προλαλήσαντες. Οπότε μου διευκολύνουν ε, το δικό μου έργο. Όπως ήδη υπόθηκε από τον κύριο Γκολτιέρη, το θέμα του τι ε, πρέπει να γίνει στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ε, χωριστά ε, και αποκομμένο από τη γενικότερη ε, θεσμική αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Εγώ όμως ανέλαβα να μιλήσω για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και σε αυτή θα επικεντρωθώ. Επιτρέψτε μου να πω και να επαναλάβω αν χρειάζεται ότι έχει γίνει εντυπωσιακή πρόοδος από την αρχή της κρίσης στην οικονομική διακυβέρνηση. Μια πρόοδος που ήταν ε, αδιανόητη πριν την κρίση. Η δομή όμως ε, που δημιουργήθηκε και απορρέει από όλες τις πρωτοβουλίες και τα επιτεύγματα είναι συγκεχημένη, είναι θολή για να δανειστώ ε, το χαρακτηρισμό του Think Tank Bruegel. Και αυτός ο μεγάλος αριθμός αποφάσεων, διεθνών συμφωνιών και ρυθμίσεων ε, οδήγησε σε ένα ε, patchwork, σε μια κουρελού ε, μέτρων. Όπως είπε και ο Ζαν Κλοντ Πυρίς. Έχουν εγκριθεί διάφορα μέτρα που δεν είναι της ίδιας φύσεως στο καθένα και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ε, και με διαφοροποίηση είναι πραγματικά άναρχη. Ε, έχουμε κανόνες που σωρεύονται είτε νομικούς είτε πολιτικούς που έρχονται να συγχαίουν ακόμα περισσότερο τις ευθύνες. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι ένα καλό παράδειγμα παρά τους ισχυρισμούς για το στόχο του για να, για να κρατηθούν πραγματικά διαφορετικές οι διάφορες διαδικασίες. Όπως είπε και έγραψε ο Άντριου Ντάφ στο πρόσφατο βιβλίο του, Υπάρχουν πολλά όργανα, θεσμικά όργανα, Eurogroup, ECOFIN, με διαφόρους προέδρους κάθε φορά, Eurogroup, Working Group, Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή και τώρα έχουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Όλα αυτά τα πρόσωπα και οι θεσμοί ε, ασχολούνται με την ΟΝΕ. Έχουμε μια διακυβέρνηση πλέον κατακαιρματισμένη ε, και ε, έρχεται να απαντήσει στην έλλειψη της διακυβέρνησης. Ο δημοκρατικός έλεγχος ε, είναι ανεπαρκής και αυτό οφείλεται εν μέρη στην ασυμμετρία, όχι 100%. Όλα αυτά τα εντυπωσιακά μέσα δεν ε, δημιουργούν εκείνο το τείχος που θα άντεχε σε οποιαδήποτε κρίση και θα προστάτευε την Ευρωζώνη. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τις μεγάλες οικονομίες των χωρών της Ευρωζώνης. Η δομή αυτή η παρούσα είναι και ατελής και ε, ε ημιτελής και αυτά τα στις 26 Οκτωβρίου του 2011, πολύ σημαντική συνεδρίαση, ενδιαφερόμενη, ε, αφού διατράνωσαν ότι το ευρώ είναι η καρδιά του ευρωπαϊκού εγχειρήματο και θέλουν να ενισχύσουν την καρδιά αυτή, την οικονομική ένωση, για να είναι στο ίδιο ύψος με την νομισματική ένωση. Για να επιτευχθεί ένας τέτοιο φιλόδοξο όμω, στόχο. και ε, και για να βασιστούμε στα τέσσερα μπλοκ της έκθεσης Πάι χρειαζόμαστε ένα θεσμικό οικοδόμημα πιο αποτελεσματικό και πιο λειτουργικό. Ε, υπάρχουν μια σειρά ιδεών και προγραμμάτων ε, δημοσίων ή ιδιωτικών που προσπαθούν να δείξουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Με κάποια διαφοροποίηση ε, όλα για να ληφθούν υπόψη ειδικέ ανάγκες των χωρών της Ευρωζώνης και τα εμπόδια που θα μπορούσαν να ανακύψουν απουσία τέτοιας ε, διαφοροποίησης. Αλλά ε, είναι αδύνατο και μπορεί και να μην είναι και επιθυμητό να παραγνωρίσουμε πλήρως ε, την πραγματικότητα της ολοκλήρωσης των 27. Η Τραπεζική Ένωση είναι ένα καλό παράδειγμα. Αν διαβάσατε την έκθεση του ε, κ. Βάρομπάη της 25ης Ιουνίου θα είδατε ότι για να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις, της θεσμικές της ε, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ε, θα πρέπει ταυτόχρονα να διαφυλαχθεί η ε, ακαιρεότητα και η ενότητα της ενίας αγοράς. Γι' αυτό χρειάζεται και παραθέτω ε, ένα ολοκληρωμένο ε, χρηματοπιστωτικό πλαίσιο που να καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη διαφοροποίηση μεταξύ χωρών της Ευρωζώνης και χωρών εκτός της ε, Ευρωζώνης. Πολύ λεπτό όμως αυτό το εγχείρημα. Πώς γίνεται η διαφοροποίηση. Μπορεί να γίνει εντός ή εκτός των ιδρυτικών συνθήκων. Νομίζω ότι αυτό το θέμα θα καλυφθεί από άλλους ομιλητές σήμερα, αλλά επιτρέψτε μου να πω γιατί είμαι χρωμένος μερικά λόγια. Μια κεντρική ε, εποπτεία των τραπεζών μπορεί να γίνει όπως γνωρίζετε βάσει του άρθρου 127.6 της Συνθήκης ε, για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζεται Ε, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης-29ης Ιουνίου ενεστώτος έτους και στις 12 Σεπτεμβρίου με την ίδια νομική βάση έκανε πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ένα πρώτο βήμα προς την Τραπεζική Ένωση που ε, οφείλει να έχει και ένα κεντρικό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων και ένα σύστημα Καθάριση των τραπεζών για να μπορεί η εξυγίανση των τραπεζών να υπάρχει μια σύνδεση ε, των τραπεζών με ε, το ζήτημα του δημοσίου χρέους. Ε, αυτό χρειάζεται ομοφωνία στο Συμβούλιο και τυπικά διαβούλευση μόνο με το Κοινοβούλιο. Αυτή η απέτηση ομοφωνίας είναι από τις μεγαλύτερες δυσκολίες και δυναμίες της συνθήκης της Λισαβόνα. και οι πρόσφατες εξελίξεις ε, απέδειξαν, αν χρειαζόταν τέτοια απόδειξη, ότι οι δυσκολίες στην επίτευξη των στόχων μπορούν να προέρχονται όχι μόνο από τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ε, υιοθετήσει το ευρώ, που αυτό είναι σημαντικό εμπόδιο για να διαθετηθούν ε, κανόνες ειδικά για την Ευρωζώνη, αλλά μπορεί να απορρέουν αυτές οι δυσκολίες και από τις ίδιες τις χώρες της Ευρωζώνης. Για άλλα θέματα μπορούμε να φέρουμε το άρθρο 136 που έπαιξε μεγάλο ρόλο στην προηγούμενη θητεία για τη διακυβέρνηση αλλά έχει και αυτό τα όρια του. Δεν είναι ρήτρα αναθεώρηση το άρθρο 136 η ε, διαδικασία για τη γενική ενισχυμένη συνεργασία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί όπως και το άρθρο 351 ε, για να καλυφθεί το κενό στη συνθήκη, αλλά ούτε αυτό είναι πανάκια. Όλα τα βήματα αυτά δεν είναι αναγκαστικά εύκολα. Το ένα θέλει ομοφωνία. Γι' αυτό ε, μπαίνουμε στον πειρασμό να κοιτάξουμε εναλλακτικέ λύσεις και η εναλλακτική ε, λύση, πάντα με τις παρούσες συνθήκες, χωρίς αναθεώρηση, είναι το άρθρο 348 της συνθήκης, ε, χρησιμοποιήθηκε για τις συμφωνίες Σέγγεν και Πρύμ για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων. Και αυτή η διαδικασία έχει τα όρια της. Μια διεθνή συνθήκη δεν μπορεί να επεμβαίνει σε θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νομισματική πολιτική είναι αποκλειστική, ενώ η οικονομική όχι και αν εγκρίνονται όλο και περισσότεροι κανονισμοί ε, επιτόπου, θα έχουμε ένα είδος αποκλεισμού ε, λόγω της δράσης. Ε, θα πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο, μία αντιφατικό που να φτάνουμε. Έχουμε πολλούς στόχους και πολλά μέσα και εργαλεία στη συνθήκη, στο Σύμφωνο Σταθερότητας, Συντονισμού και Ανάπτυξης και Διακυβέρνησης για την Ευρωζώνη. Είναι ένα στοιχείο λοιπόν αυτό διεθνούς δικαίου παράλληλο με τη συνθήκη. Τα συμβαλόμενα μέρη δεσμεύονται εντός μιας προθεσμίας να ε, δώσουν ε, το νομικό πλαίσιο εντός ε, των συνθήκων. Αυτή η ιδέα άτυπα εκφράζεται και από την έκθεση της ομάδας Τομάσο Παντοάς Κιόπα για τη συμπλήρωση του ευρώ και τον οδικό χάρτη, το 17 και περισσότερων, και αυτό ορίζει ότι εν ευθέτω χρόνο ε, η δομή αυτή μπορεί να ενταχθεί στην παραδοσιακή νομική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει ειδικό ε, στόχος για ε, το Σύμφωνο Σταθερότητας Σύγκλησης και Διακυβέρνησης της Ευρωζώνης η συνθήκη του πρώην, ε, ε, καμιά φορά ονομάζεται και Σέγγεν θα μπορούσε να είναι ε, μια σύγκριση για μια αντίστοιχη διεθνή συμφωνία μεταξύ των κρατών μέλων. Αν κοιτάξουμε τα τέσσερα μπλοκ, τις τέσσερις ενότητες της έκθεσης Φανρόν Πάι, γίνεται μια σύνδεση ανάμεσα ε, στην πολιτική έννοια, στο πολιτικό οικοδόμημα της Ευρώπης, στα νέα βήματα που πρέπει να γίνουν προς μια πιο αποτελεσματική και δημοκρατική ε, οικονομική διακυβέρνηση. Όλα αυτά είναι πρωτοφανή ζητήματα. Ε, για πρώτη φορά αντιμετωπίζονται στην Ένωση. Στην έκθεση η Ευρώπη μας και στην έκθεση Βαν ε, Ρομπόι προς μια γνήσια οικονομική και νομισματική ένωση γίνεται λόγος για ένα πακέτο, για μια δέσμη και με ποιοτικά μέτρα που θα υλοποιούνται προοδευτικά ε, με ένα προκαθορισμένο ε, χρονοδιάγραμμα η κατάληξη είναι Τραπεζική Ένωση και η Δημοσιονομική Ένωση, η οποία πηγαίνει χέρι με χέρι με μεγαλύτερη οικονομική ένωση και συμπεριλαμβάνει και την ανάγκη και χρειάζεται ε, μεγαλύτερη πολιτική ένωση. Είναι σημαντική πρόοδος προς μία ολοκλήρωση που δεν είναι δυνατόν να γίνει με ε, τρόπο διακυβερνητικό. Σε ό,τι φορά την ομολογία του ΔΕΚ, όπως είπαμε, υπάρχουν ε, εγγενή ε, όρια σε παράλληλες διεθνείς ε, συνθήκες. Δεν είναι αποτελεσματικό ούτε ευαρκές υποκατάστατο στην αναθεώρηση των συνθήκων. Σε περίπτωση κατεπίγουσας ανάγκης θα μπορούσε κάτι τέτοιο να είναι αποδεκτό, αλλά ε, ε, χωρί να έχει εντό εισαγωγικών επαναστατικέ αλλαγές στη σχέση μεταξύ της Ένωση και των κρατών μετών, μελών, ούτε μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Επιπλέον, ε, πλεονεκτήματα για τη δημοκρατία και τη διαφάνεια θα είχε η αναθεώρηση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση δια της κανονικής οδού αναθεώρησης για τροποποίηση συνθήκης με συντακτική συνέλευση. Η επιλογή αν θα γίνουν αυτά εντός ή εκτός των συνθήκων ε, εξαρτηθούν πάρα πολύ από το δρόμο που θα πάρει το Ηνωμένο Βασίλειο στις μελλοντικές σχέσεις με την υπηρετική Ευρώπη. Χρειάζεται ε, μια ε, αποσαφήνιση και όσο γρηγορότερο τόσο καλύτερα. Την άλλη εβδομάδα οι εταίροι θα γνωρίζουν περισσότερα για τη βρετανική στάση, για τη μεταρρύθμιση. σε σχέση με το όσα αποφάσισε το Συμβούλιο 28-29 ε, Ιουνίου. Όπως και τον περασμένο Δεκέμβριο, οι Βρετανοί ε, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν αυτό που αποκάλεσε ο Νταφ μία άκομψη βρετανική ε, πρωτοβουλία και θα πρέπει να απαντήσουν. Βεβαίως υπάρχει και το Εθνικό Σύνταγμα ε, κάθε φορά και τα συνταγματικά δικαστήρια πέρα από τα ευρωπαϊκά. Θα παίξουν ένα ρόλο αυτά τα δικαστήρια ε, και κυρίως το ε, Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο συγκέντρωσε την προσοχή και κίνησε τη συζήτηση. Δεν χρειάζεται νομίζω να επιμείνω εγώ σε αυτό το στοιχείο αυτή τη στιγμή. Τα γνωρίζουμε πολύ καλά από τα πρώτα μέτρα που ελήφθησαν για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Ε, από την απόφαση του για το Μάστριχ το 1993 ε, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας ε, χαράσει το πλαίσιο για τη δημοκρατία και τη σταθερότητα. Γνωρίζουμε ότι η Γερμανική Βουλή θα πρέπει να παραμείνει κύριος και κυρίαρχος των αποφάσεών τους. Αυτή η ιδιαίτερη σημασία της αρχής αυτής γίνεται όλο και πιο σαφής μετά από μια σειρά αποφάσεων. Η δημοσιονομική πειθαρχία λοιπόν δεν είναι ε, κάτι που βρίσκει αντίθετο το συνταγματικό δικαστήριο. Βλέπετε την απόφαση για τη Λισαβόνα, αλλά εδώ βλέπουμε πώς περιορίζεται ε, η ισχύ των εθνικών κοινοβουλίων, ε, αλλά χρειάζεται και κάποια νομιμότητα ο θεσμός που τα επιβάλλει. Ε, η ομάδα Βέστερβέλε και κάποιων ε, Υπουργών Εξωτερικών ε, έδειξε ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να αποφασίζουν για τον προπολογισμό. Αυτά είναι κάποια ανυπέρβλητα όρια. Ε, βλέπω ότι τελειώνει ο χρόνος μου και το τρίτο θέμα που θέλω να αναφέρω είναι ο δημοκρατικός έλεγχος και η διακυβέρνηση. το είπαν και οι προλαλήσαντες και το τόνισαν. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος θα πρέπει να ενισχυθεί και στις χώρες της ΟΝΕ. Πώς θα οργανωθεί αυτός. Αναφερθήκατε στην θέση που λέγει ότι θα πρέπει να δούμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μήπως χρειαστεί να αναλάβουν κάποιο ρόλο για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ας πούμε, στο άρθρο 13 της ε, Συνθήκης για τη Διακυβέρνηση του Ευρώ θα πρέπει να δούμε ποια ε, είναι ε, τα πλαίσια εξουσίες, αμυγός συμβουλευτικές ή όχι, τα Εθνικά Κοινοβούλια και όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι οι συλλογικοί ε, ελεγκτές, οι κανονικοί ελεγκτές αυτού του συστήματος. Τι μας διδάσκει η μέχρι τώρα εμπειρία από τη Συνθήκη της Λισαβόνα, από τα Εθνικά Κοινοβούλια για τον έλεγχο της επικουρικότητας και τι εξουσίες που τους έχει δώσει. Σας παραπέμπω στην ανάλυση που έχω κάνει σχετικά τα θέματα τα δημοσιονομικά θα τα συζητούν οι οικονομικές επιτροπές των Εθνικών Κοινοβουλίων και ε, θα, ε, τα κάνουν κτήμα τους τα κράτη αυτά τα ζητήματα τα ευρωπαϊκά και ποια λογοδοσία θα χρειαστεί στις νέες πολιτικές αντίστοιχες ε, με τις σημερινές του οικονομικού και νομισματικού διαλόγου ή θα είναι πιο συγκεχημένες. Τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη λογοδοσία της και όταν δρά και ως κεντρικός τραπεζίτης για τα νομισματικά αλλά και για την προληπτική εποπτεία. Πώς θα ενημερώνει το Κοινοβούλιο σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 21 του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό ε, Σώμα ε, Συστημικού Κινδύνου. Ε, ας πούμε τι κατεύθυνση θα ληφθεί σε σχέση με τα όσα ε, λέγει η έκθεση Humboldt του αντιστοιχού ε, Πανεπιστημίου του Βερολίνου που σας έχει παρουσιαστεί για τα δικαιώματα μειοψηφία και για το να έχει την τελική απόφαση για τα ελλείμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Όλα αυτά είναι ζητήματα πάρα πολύ ε, ενδιαφέροντα σε ό,τι αφορά τις κυβερνήσεις και τη διακυβέρνηση. Δεν μπορώ να επεκταθώ γιατί τελειώνει ο χρόνος μου. Ε, τι ρόλο θα έχει ο Υπουργό Οικονομικών. Ε, ε, θα είναι ένα Υπουργείο Οικονομικό Ευρωπαϊκό, αυτά λέγει η έκθεση Φαν Ρομπάι, που στο μέλλον θα παραμείνει ένα όργανο ελέγχου ταξί ομοτήμων. Αλλά αυτό έχει δείξει αδυναμίες και, και ότι δεν είναι βιώσιμο. Όταν υπάρχει υπερβολικό έλλειμμα ή μακροοικονομικές ανισορροπίες, πώς θα δρά αυτό. Η έκθεση Ευρώπη μα Notre Europe, επιμένει στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι το υποκείμενο τη πολιτική αυτή. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Υπουργό Οικονομικών με τον τρόπο που προτείνεται, όχι μόνο στην παρούσα έκθεση, αλλά και από τον Jean-Claude Trisset, λέγει ότι Ε, τα θέματα της ε, κυριαρχίας πλέον συνδέονται με τη φερεγγιότητα και ε, έχουμε μια ομοσπονδία, ένα φεντεραλισμό ή μια, μια ομοσπονδία κατ' εξέρεξη. Δηλαδή, αν μια χώρα διαρκώς παραβιάζει τους κανόνες, χάνει τη δημοσιονομική του κυριαρχία. Αυτό ε, υπόθηκε το περασμένο Ιούλιο. Μα τέτοια εξουσία έκτακτη πώς εκχωρείται. Η πιο προληπτική δράση δεν είναι πιο αποτελεσματική όπως αναγνωρίζει η δέσμη των έξι οδηγιών. Και τι ε, ε, νομιμοποίηση έχει ένας τέτοιος υπουργό Οικονομικών. Θα ήθελα να πω και δύο λόγια τώρα, ολοκληρώνοντας για την Ευρωζώνη στην παγκόσμια σκηνή. Πιστεύω ότι έχει έρθει ο χρόνος ε, η Ευρώπη να έχει εκπροσώπηση για το ευρώ παγκοσμίω και διεθνώς και στο σύστημα Bretton Woods αλλά και κατά την άποψή μου σε όλους αυτούς τους ε, φορείς ε, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ε, ή προτύπων ε, η πολύ ισχυρή και σκληρή Επιτροπή της Βασιλείας για την εποπτεία των τραπεζών και γίνεται παγκόσμια αναφορά για βέλτιστες πρακτικές στα λογιστικά των τραπεζών και έχει σημαντικό ρόλο, για να μην πω αποφασιστικό, και στις αντίστοιχες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει έρθει η ώρα, πιστεύω, λοιπόν, το άρθρο 138 να εφαρμοστεί σε τέτοιες περιστάσεις ε, σε οργανισμούς ε, προτύπων. Ξέρω ότι εμείς δεν εγκρίνουμε τραπεζικούς κανόνες. Ε, θα πρέπει να συγκεράσουμε την προστασία του γενικού οικονομικού συμφέροντος της Ευρωζώνης με την εμπειρία και τις δεξιότητες εθνικών θεσμών. Για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μία από τις λύσεις θα μπορούσε να είναι να υπάρχει μια περιφέρεια για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Το θέμα είναι ποιος θα προεδρεύει εκεί. Ε, υπάρχουν διάφορες απόψεις που κυκλοφορούν, αλλά από ό,τι φαίνεται η λύση θα εξαρτηθεί από τη μεταρρύθμιση την ίδια του ε, δούλου του, γιατί το εκτελεστικό συμβούλιο δεν θα είναι πλέον και το διοικητικό συμβούλιο. Ε, το γνωρίζουμε προς το παρόν είναι, αλλά μπορεί να γίνει ένα ε, όργανο απλώς εποπτείας και ε, το προσωπικό θα έχει μεγαλύτερο ρόλο. Εν πάση περιπτώσει αυτά είναι θέματα που είναι προς συζήτηση. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Άρχισα με ε, την ανάγκη να έχουμε αποτελεσματική διακυβέρνηση για την Ευρωζώνη χρειάζεται να προβληματιστούμε στη συζήτηση και τελειώνω επιμένοντας για μια πιο λογική και αποτελεσματική εκπροσώπηση διεθνώς ε, ανάλογη με τη σημασία της Ευρωζώνης. Είναι ιστορικός ο ρόλος, η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει παγκόσμιος πρωταγωνιστής. Αυτό το λέει και ενδιάμεση έκθεση ε, των Προέδρων των Υπουργών Εξωτερικών για το μέλλον της Ευρώπης 15 Ιουλίου 2012. Σας ευχαριστώ. E Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Και τώρα ο καθηγητής Γιάννης Εμμανουηλίδης που που προέρχεται από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής των Βρυξελών, σύμβουλος των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και διαφόρων μη κυβερνητικών οργανισμών, συγγραφέας διαφόρων έργων για τις εξελίξεις της θεσμικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια είμαι υποχρεωμένος να ζητήσω από τους ομιλητές μας να ελέγξουν ε, το ε, χρονικό τους όριο γιατί πρέπει όλους να τους ακούσουμε. Λοιπόν, αν αυτό ελεγχθείτε θα είναι καλύτερα. Λοιπόν, κύριε Εμμανουηλίδη. Thank Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα ευγενικά σας λόγια και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση για τη συζήτηση αυτού του πολύ επικαιρού θέματος. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που είμαι εδώ. Όταν ε, μου ζήτησα να σκεφτώ το θέμα της συζήτησης, ε, αναρωτήθηκα ποια είναι τα διδάγματα της ε, διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης και η παρούσα χρήση της διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης. Βέβαια, είναι σχεδόν αδύνατο να καλύψει κανείς όλο αυτό το προβληματισμό, γιατί μάθαμε πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες ουσιαστικά, μερικά τα περιέλαβα στο εγγραφό μου. Έχουμε τόσα πολλά διδάγματα που θα μου είναι δύσκολο να επικεντρωθώ σε ένα τέταρτο μόνο. Θα προσπαθήσω όμως ε, να εστιαστώ σε έξι βασικά διδάγματα και να τα συνδέσω με το παρελθόν, με τα διδάγματα της διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης και ε, να τα συνδέσω με το προβληματισμό για την περαιτέρω ευάθυνση της ολοκλήρωσης σε οικονομικά και δημοσιονομικά ζητήματα, κάτι που θεωρούμε όλοι αναπόφευκτο για τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο μέσα σε ένα τέταρτο να αναλύσω όλα αυτά τα θέματα. Μερικές φορές θα είμαι κάπως πιο επιγραμματικός, άλλες φορές ε, υπεραπλουστευμένο θα τα παρουσιάσω. Έχω δυόμιση λεπτά για το καθένα ουσιαστικά. Καταρχήν, το πρώτο θέμα μπορεί να παραφαίνεται γενικό, αλλά είδαμε από μια σφοδρή και φλογερή συζήτηση τα τελευταία δύο-τρία χρόνια ότι η διαφοροποιημένη ολοκληρώση έδωσε μια στρατηγική ευκαιρία για μια μεγαλύτερη και πιο ετερόκλητη όλο και περισσότερο Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ήταν ένα, αυτό ήταν ένα δίδαγμα του, δίδαγμα του παρελθόντος και μερικές φορές η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση ήταν καταλήτης για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αν όμως ακολουθήσουμε τη συζήτηση για διευθυντήρια, τριανδρίες, ομάδες πρωτοπόρες, ε, κέντρα βαρύτητα, πυρήνε κτλ. Βλέπουμε ότι έχουμε υπεραπλουστεύσει, απειλέ, φόβου, σημασιολογικέ και ενιολογικέ παρεξηγήσει. Και αν αυτά τα χρησιμοποιήσουμε ως δίδαγμα του παρελθόντος, στο μέλλον θα πρέπει να αποδραματικοποιήσουμε τη συζήτηση. Και σημείο κίνησης είναι ότι η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση Όπω την ξέρουμε και η Ευρώπη πολλών ταχυτήτων είναι ήδη μια πραγματικότητα. Οπότε το κεντρικό ζήτημα τώρα είναι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια διαφοροποίηση. όχι αν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια διαφοροποιημένη ολοκλήρωση, αλλά τι είδου ε, τέτοια ολοκλήρωση χρειαζόμαστε. Σε ό,τι αφορά την εμβάθυνση τη οικονομική και διαμεσονομικής ολοκλήρωση, εκεί η διαφοροποίηση μα δίνει μια στρατηγική ευκαιρία και ω τέτοια θα πρέπει να την ε, αντιληφθούμε. Αλλά δεν είναι ούτε μαγικό φίλτρο, ούτε πανάκια, ούτε αυτό. σκοπό είναι ένα μέσο μόνο για να κρατήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως ε, την Ευρωζώνη ε, λειτουργική. Δεύτερο δίδαγμα. Αν δούμε λίγο το ιστορικό της διαφοροποίησης και διάφορα παραδείγματα διαφοροποίησης, διαπιστώνουμε ότι η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση ποτέ δεν ήταν η συνέχεια ενός ε, συγκεκριμένου στόχου, δεν επιδίωξε ένα συγκεκριμένο στόχο, αλλά ουσιαστικά ήταν ε, μια προοδευτική, σταδιακή, λειτουργική, ρεαλιστική διαφοροποίηση προκειμένου να υπερκεραστούν κάποιες, κάποια διέξοδα. Ήταν ουσιαστικά μηχανισμός έσχατης ανάγκης και το ίστατο επιχείρημα, ultima ratio. Οπότε δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον ε, διαφοροποιημένη ολοκλήρωση και τη γενική αυτή συζήτηση για να υλοποιήσουμε ένα συγκεκριμένο στόχο. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αντιπαραγωγικό. Είναι πολύ πιο χρήσιμο να χρησιμοποιήσουμε μια λειτουργική προσέγγιση και να χρησιμοποιήσουμε τη διαφοροποιημένη ολοκληρώση για να ξεπεράσουμε συγκεκριμένε προκλήσει. Και έχουμε μια συγκεκριμένη πρόκληση, την κρίση στην Ευρωζώνη. Θα πρέπει να δούμε πώ θα την ξεπεράσουμε με ρεαλιστικό τρόπο. Μην με παρεξηγήσετε. Δεν εννοώ ότι δεν θα πρέπει να έχουμε κατά νου ένα στόχο ε, ή μπορούμε να αναλύσουμε το γιατί θα πρέπει να κάνουμε ορισμένα πράγματα και να χρησιμοποιήσουμε την διαφοροποιημένη ολοκληρώση χωρίς να έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο, αλλά κάποια, κάποιους πιο γενικούς στρατηγικούς σκοπούς. Δεύτερο δίδαγμα είναι ότι η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση, όπως ε, φαίνεται και στα γραπτά των συναδέλφων, δεν οδήγησε σε, μια θεσμοποιημένη, ε, σε ένα θεσμοποιημένο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε ένα πιο συνεκτικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να έχουν δημιουργήσει μια πρωτοπόρα ομάδα που έχει διαχωριστεί από τις υπόλοιπες. Βλέπουμε την επισκόπηση του κυρίου Βέσελ στη σελίδα 28 που μας δείχνει πόσο περίπλοκη είναι όλη αυτή η δομή. Αλλά δεν υπάρχει μία ομάδα σκληρού πυρήνα ή εμπροστοφυλακής ή πρωτοπορίας. Υπάρχουν διάφορες μορφές ε, διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης με διαφορετικά κράτη-μέλη κάθε φορά. Και το δίδαγμα για το μέλλον είναι ότι θα πρέπει να αποφύγουμε μία Ευρώπη δύο ταχυτήτων ή μία ένωση εντός της ένωσης, όπως είπε προηγουμένω, αν δεν κάνω λάθο, ο κύριος Λουί. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη και φυσικά χρησιμοποιώντας και τα διδάγματα του παρελθόντος. Καταρχήν, δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ανυπέρβλητα εμπόδια για τους pre-ins ή τους outs. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ε, ε, μόνιμους, παράλληλους ε, μηχανισμούς και θεσμούς. Όχι ξεχωριστό κοινοβούλιο της ε, Ευρωζώνης, όχι η Ειδική Επιτροπή της Ευρωζώνης, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος του κατακαιρματισμού. Επίσης, να μην γίνει διαφοροποίηση μεταξύ της χώρες Ευρωζώνης και της χώρες πέραν της Ευρωζώνης ή της εκπροσώπησής τους στην Επιτροπή ή το Δικαστήριο. Γιατί είχαμε κάποιε ενδείξει προ αυτή την κατεύθυνση. Κατά τη γνώμη μου είναι εσφαλμένη αυτή η κατεύθυνση και σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Γιατί κάτι τέτοιο θα υπονομεύσει τους υπερεθνικούς χαρακτήρες αυτοθεσμικών οργάνων και την εκπροσώπηση των χωρών εκτό τη Ευρωζώνη σε συγκεκριμένου τομεί και θα διαρρήξει το δεσμό μεταξύ τους, ε, των pre-ins, των ins και των outs και θα δημιουργήσει μεγάλη δυσπιστία. Οπότε τα βασικά θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως είπε και ο προλαλής είναι το πώς θα ε, ενισχύσουμε την δημοκρατική νομιμοποίηση σε μια όλο και πιο διαφοροποιημένη Ευρώπη. Εδώ υπάρχουν δύο βασικά θέματα. Το θέμα είναι πώς θα γίνει η διάκριση μεταξύ των ε, ευρωβουλευτών από τις χώρες Ευρωζώνης και τις χώρες εκτός Ευρωζώνης και μετά πώς θα αναμίξουμε και τα εθνικά κοινοβούλια. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες στο θέμα αυτό, γιατί θα μας απασχολήσει λίγο αργότερα αλλά αν σκεφτούμε πώς ε, ε, θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε τη διαφοροποίηση με την νόμιμοποίηση, ε, πιστεύω ότι είναι δύσκολο να δώσουμε μια απάντηση αν δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, προκειμένου να φτάσουμε, μια πιο, να φτάσουμε πιο κοντά σε μια Οικονομική και Δημοσιονομική Ένωση που θα εμπεριέχει και κάποια στοιχεία πολιτικής ένωσης. Θα πρέπει να έχουμε επίγνωση των συγκεκριμένων μέτρων και γι' αυτό χρειαζόμαστε προηγουμένως μια συμφωνία για τα συγκεκριμένα μέτρα. Και στη συνέχεια θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε τι θα σημάνει κάτι τέτοιο υπό το πρίσμα της δημοκρατικής νομοποίησης. Ε, πρέπει να ξέρουμε αν θα υπάρχει ένας κοινωτικός προϋπολογισμός ή ένας προϋπολογισμός πολλών ταχυτήτων, αν θα έχουμε μια δημοσιονομική αρχή ή έναν ε, Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομικών. Ε, και έναν ε, μηχανισμό που δεν θα είναι μόνο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα, αλλά Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταθερότητα. Τι θα σημάνουν όλα αυτά. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τι λεπτομέρειε για να δούμε ε, πώ θα γίνει η διαφοροποίηση μεταξύ Ευρωβουλευτών Ευρωζώνη και Ευρωβουλευτών από χώρε εκτό Ευρωζώνη και πώ θα αναμειχθούν τα εθνικά κοινοβούλια στην όλη διαδικασία. Υπάρχει ένα κίνδυνο, ίσω ε, περιπλέξει κάπως το σύστημα, αλλά είναι μια εύλογη ανησυχία πριν ο κύριος Λουί μας ανέφερε το, την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου. Θα πρέπει όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη. Τέταρτο δίδαγμα. Ε, έχουμε πολλές θεσμικές και πολιτικές προκλήσεις που σχετίζονται με την ολοκλήρωση. Και ε, αυτό σχετίζεται και με την οργάνωση του ευρωπαϊκού πλαισίου έχουμε ένα τέτοιο δίδαγμα από το παρελθόν. Αν ε, έχουμε μια οργάνωση της διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης εντός του ε, νομικού πλαισίου της ε, συνθήκης, στα πλαίσια των συνθήκων, αποφεύγουμε μια άναρχη διαφοροποίηση. Σεβόμαστε το θεσμικό πλαίσιο και περιορίζουμε τον άναρχο και ανεξέλεκτο τρόπο χρήσης της διαφοροποίησης και βελτιώνουμε τον τρόπο υπολογισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όσους δεν συμμετέχουν σε κάποιες μορφές της διαφοροποίησης, γιατί έχουμε σαφείς κανόνες σε σχέση με την αρχή, την λειτουργία και τη διεύρυνση της διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης και έτσι έχουμε ένα μεγάλο άνοιγμα, μια μεγάλη διαφάνεια. Βέβαια, τα διδάγματα του παρελθόντος ε, μας ε, έχουν ε, διδάξει ότι μερικές φορές δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Νομικού Πλαισίου, αλλά θα πρέπει να προβλέψουμε κάποιους τρόπους διαφοροποίησης εκτός, όπως σύμβαση του Σέγγεν ή σύμβαση Προύμ σημαντικά παραδείγματα. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τη διαφοροποιημένη ολοκλήρωση εντό του νομικού πλαισίου τη συνθήκη ή δυνατόν. Αν όμω κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο ή μερικέ φορέ τουλάχιστον όταν είναι κάτι τέτοιο αδύνατο, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και έρχομαι στο πέμπτο ε, δίδαγμα διακυβερνητική συνεργασία εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι τέτοιο ενέχει πολλού κινδύνους. Και ο βασικό κίνδυνο είναι ο κατακαιρματισμό, η ρήξη, η διαίρεση μεταξύ αυτών που συμμετέχουν σε κάποιε μορφέ ε, ολοκλήρωση Στην περίπτωσή μα ε, Ευρωζώνη, χώρε Ευρωζώνη και χώρε εκτό Ευρωζώνη. Υπάρχει ένα γενικό κίνδυνο, αλλά υπάρχει και ένα ειδικό κίνδυνο. Αν δούμε τη συζήτηση για την Τραπεζική Ένωση. Είδατε στην Πολωνία, για παράδειγμα, πώ διεξήχθη η συζήτηση και εκεί υπάρχουν συγκεκριμένε ανησυχίε, όχι μόνο γενικέ, αλλά και διαφοροποίηση ω προ την Τραπεζική Ένωση. Πέραν των κινδύνων αυτών πάντως, η διαφοροποίηση, η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση ε, ήταν ε, ε, εποφελής και στο παρελθόν και πιστεύω ότι μπορεί να είναι χρήσιμη και στο μέλλον. Ε, θα μπορούσαμε να έχουμε μια διακυβερνητική πρωτοπορία, για παράδειγμα, με τρει προποθέσει όμω. Καταρχήν, ανάμειξη ε, και μερικέ φορέ και ενίσχυση του ρόλου των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, στο μέτρο του δυνατού υπάρχουν φυσικά και όρια σε αυτό. Δεύτερον, η διακυβερνητική εμπροστοφυλακή αυτή η πρωτοπορία να είναι ανοιχτή προ όλε τι χώρε που θέλουν να συμμετέχουν και τρίτη προϋπόθεση να υπάρχει συγκεκριμένο στόχο, ιδιαίτερα των ε, βασικών χωρών μελών που προώθησαν την συνεργασία εκτός της, του πλαισίου της συνθήκης να συμπεριλάβουν αυτή την εξωτερική διαφοροποιημένη ολοκλήρωση να τη συμπεριλάβουν στο πλαίσιο το νομικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συνθήκης το συντομότερο δυνατόν. Για παράδειγμα, έχουμε την, ε, την, ε, ε, τη συνθήκη για το μηχανισμό σταθερότητας αλλά και τη συνθήκη σταθερότητας σύγκλησης και διακυβέρνηση Ευρωσόνη. Αν δείτε το σύμφωνο Ευρώπη-ΣΥΝ, σε όλε αυτέ τι περιπτώσει είχαμε μία απόπειρα παρά τι ε, συγκεκριμένε πιέσει του χρόνου και τη κρίση να εμείνουμε σε αυτέ τι αρχέ ε, και τι προποθέσει που σα προανέφερα. Δεν ε, δημιουργήθηκαν νέε παράλληλε θεσμικέ δομέ με εξαίρεση το Euro Summit, αλλά υπάρχουν σαφεί δεσμοί και στενεί δεσμοί μεταξύ των χωρών τη Ευρωζώνη και των χωρών εκτό τη Ευρωζώνη και υπάρχει μάλιστα ανάμειξη των κοινοτικών θεσμικών οργάνων στην ε, στον τρόπο δανεισμού, για παράδειγμα. Και ε, το είδαμε και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΕΚ στη, στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο, Fiscal Compact Treaty Επίσης, ε, είδαμε την ανάμιξη κάποιων υπερεθνικών θεσμικών οργάνων και το είδαμε αυτό στη διάρκεια της κρίσης, αλλά πιστεύω ότι θα δούμε κάτι τέτοιο πολύ πιο έντονο και μετά την κρίση και διεύρυνση βασικών θεσμών της Ένωσης, ε, ε, γιατί αν ε, δούμε τι συνέβη στο 2010 και το καλοκαίρι του 2011, είδαμε ότι υπήρξε μια όθηση για, την, για τον τονισμό υπερεθνικών θεσμών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μερικές χώρες, όπως η Γερμανία, η πατρίδα μου για παράδειγμα, διαπίστωσαν ότι έχει νόημα να ασκηθεί πίεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς τα κράτη-μέλη και όχι μόνο από μία χώρα προς τις υπόλοιπες χώρες. Αυτό τώρα σε ό,τι αφορά την διευρυμένη σταθερότητα και το σύμφωνο ανάπτυξη. Έχουμε σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, αλλά και στην ε, διαδικασία των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Εκεί θα πρέπει να δούμε αν λειτουργούν όλα αυτά. Πάντω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα αυτά τα θέματα έχει αναλάβει πολύ θεμελιώδη ρόλο. Επίση για τα προγράμματα διάσωση έχει σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια και συμμετέχει στην Τρόικα. Βέβαια, δεν είμαι αφελή. Διαπιστώνω ότι υπάρχουν κίνδυνοι στην ε, διακυβερνητική μέθοδο. Βέβαια, είναι ρευστή χρήση των όρων, γιατί ε, με την ε, Λισαβόνα είναι πια ρευστά τα μεταξύ διακυβερνητική και υπερεθνική διάσταση. Βέβαια, ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ε, θεμελιώδη το εξαπλό πακέτο, το διπλό πακέτο, τα θέματα και τη συζήτηση για τα ευρωομόλογα, την κοινή ανάληψη του χρέους κτλ. Και διαπιστώνουμε ότι έχουμε μια, έναν αποκλεισμό της, ε, του ελέγχου των ομοτήμων. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένα άνοιγμα για τι ε, διακυβερνικέ ρυθμίσει μεταξύ όλων των χώρων μελών. Είχαμε το τις έξι χώρε που είναι εκτό τη που συμμετέχουν στην ε, ε, συνθήκη για τη σταθερότητα, σύγκληση και διακυβέρνηση. Οχτώ μάλιστα χώρε εκτό τη Ευρωζώνης συμμετέχουν. Και βέβαια θα πρέπει να είμαστε ειλικρινοί. Οι χώρε τη, ε, ε, εκτός Ευρωζώνης μερικές φορές παραγωνίστηκαν, αλλά ήταν θετικές οι επικρίσεις που άσκησαν και επίση ήταν πολύ θετική συμμετοχή του στην υπέρβαση τη κρίση, γιατί δημιουργήθηκε μια εμπιστοσύνη για το γεγονό ότι οι χώρε εκτό Ευρωζώνη άσκησαν τέτοια πίεση στις χώρες Ευρωζώνη, λέγοντα ότι ε, για το ευρώ ενδιαφερόμαστε και εμεί. Και η τρίτη προπόθεση είναι η στόχος συμπερίληψη των κανόνων που ε, λύθησαν εκτό ε, του νομικού πλαισίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση στου κανόνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπως, είναι, όπως συμβαίνει και με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Βέβαια, με δύο τρόπους μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί κανείς να είναι ε, υπέρ ε, μιας ε, μεγάλης εμβέλειας αναθεώρησης της συνθήκης, προκειμένου να συμπεριληφθούν και τα νέα στοιχεία. Υπάρχουν κάποια κίνδυνοι εδώ βέβαια. Και η δεύτερη πιο συντηρητική προσέγγιση, με βάση την εμπειρία και του παρελθόντος. Και υπάρχει και η πρόταση για επιπλέον διακυβερνητικές συνθήκες. Νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις διάφορες μεθόδους. Δηλαδή στην επόμενη φάση μετά το Δεκέμβριο να έχουμε ε, πολύ περισσότερες προσπάθειες με ένα δίκτυ ασφαλείας, γιατί χρειάζεται δίκτυ ασφαλείας, παρόλο που έχει χαλαρώσει λίγο η κρίση, δεν έχει εξαλειφθεί. Και μπορούμε ίσως να χρησιμοποιήσουμε και τα δύο. Οπότε το δίδαγμα του παρελθόντος λέει να χρησιμοποιήσουμε τις αντικυβερνητικές ρυθμίσεις και να τις επαναφέρουμε στο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το συντομότερο δυνατό, γιατί όσο περισσότερο μένουν εκτός, τόσο πιο πολλοί κίνδυνοι δημιουργούνται. Επίσης, ήθελα να πω ότι τελευταία διετία η κρίση του ευρώ δημιούργησε μια νέα ποιότητα και μια νέα συζήτηση, μερικές φορές αντιπαραγωγική, για τις πιθανές προοπτικές και τις συνέπειες της αρνητικής ολοκλήρωσης, όπως είπαμε. Έγινε η συζήτηση αυτή σε σχέση με την Ελλάδα, σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και όπως είπα πολλές φορές ήταν αντιπαραγωγική ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Και έχουμε δύο πιθανούς ε, τύπους ε, μη ολοκλήρωση. Για παράδειγμα, απομάκρυση κάποιων χωρών από κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές και δεύτερον, μια πιο ριζοσπαστική αρνητική μορφή διαφοροποίηση, έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ξεκινήσουμε με το δεύτερο, την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, εδώ δεν έχουμε διδάγματα από το παρελθόν, δεν έχουμε τέτοιε εμπειρίε. Το άρθρο 50 μα δίνει κάποιου προσανατολισμού. Αν κάτι τέτοιο ε, λάβει χώρα, θα πρέπει να βρεθεί μια συμφωνία για νέο είδου σχέσει μεταξύ τη χώρα που έχει εξέλθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και των υπολείπων. Εδώ ίσω θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια σύνδεση ή ενισχυμένη σύνδεση. Κάτι παρόμοιο έχουμε με την Τουρκία στην Τελωνιακή Ένωση. Ή να δημιουργήσουμε κάτι ακόμη πιο ισχυρό, ε, ένα είδο μερική συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε η αποχωρούσα χώρα να συμμετέχει σε κάποιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και να ψηφίζει και να έχουμε ένα είδο πιο ενισχυμένη σύνδεση, δηλαδή. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι είναι μάλλον απίθανο ε, να εξέλθει μια χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ερχόμαστε στη δεύτερη μορφή αρνητικής διαφοροποίησης ε, της αποχώρηση από ορισμένε πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένοντα όμω μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε και αυτό είναι ευκταίο σενάριο, αλλά είναι πιθανό. Ακούσαμε να μιλάνε κάποιοι για περιορισμένη συμμετοχή, για συμμετοχή μείωνη, συνδεδεμένη συμμετοχή, όπω είπα ο Άντριο Νταφ. Ε, το θέμα είναι ότι η χώρα που θέλει να αποσυνδεθεί από κάποιες πολιτικές να παραμένει παρόλα αυτά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι μια πιθανότητα που θα μπορούσαμε να την ε, μελετήσουμε. Αν κάτι τέτοιο όμως υλοποιηθεί, θα έχουμε, δύο διαφορετικές, ε, θα έχουμε διαφορετικές μορφές συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έννοια αυτή δεν είναι καινούρια, αλλά με την συζήτηση αυτή δημιουργούνται νέες προπτικές και ίσως και νέοι Νέε ευκαιρίες για χώρες που θέλουν να έρθουν κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν είναι σε θέση ή μερικές φορές δεν επιθυμούν ε, πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, υπάρχει ένα είδος διαφορετικής συμμετοχής. Αυτή είναι η νέα συζήτηση. Ε, δυστυχώς δεν επιθυμουν πληρη ενταξη στην ευρωπαικη ενωση ναι υπαρχει ενα είδο διαφορετική συμμετοχης αυτη ειναι η νεα συζητηση δυστυχως δεν τηρησα το χρόνο μου πιστά, αλλά ελπίζω ότι μερικές τουλάχιστον από τι παρατηρήσει μου να δώσουν τροφή για σκέψη. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, τα σημειώνουμε όλα αυτά που είπατε και τα όσα θα πούνε και οι υπόλοιποι. Και τώρα δίνω το λόγο στον καθηγητή Μπρούνο Ντεβίτε, που είναι καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μάστριχτ, επίση διδάσκει στο Ινστιτούτο της Φλωρεντίας και ενδιαφέρεται για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το διεθνές ε, δίκαιο. Παρακαλώ κύριε καθηγητά να πάρετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα μιλήσω στα αγγλικά. Το θέμα που μου ανετέθη είναι αρκετά συγκεκριμένο. Πρόκειται για ένα νομικό ζήτημα. Το κατά πόσο δηλαδή η οθέτηση από πλευρά των κρατών μελών διαφόρων διεθνών συνθήκων, όπω η ΕΣΕΜΑ για τον Μηχανισμό Σταθερότητα και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, εκτό δηλαδή του πλαισίου των συνθήκων, και κατά πόσο αυτό οδηγεί σε ασυνέπειε σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το συμπέρασμά μου, το οποίο μπορώ να σας πω από τώρα, μπορεί να βοηθήσει να χαλαρώσει κάπως η συζήτηση, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, γιατί πιστεύω πως ο, εν γέννη δεν υπάρχουν από νομικής άποψης τόσες πολλές ασυνέπειες. Καταρχήν θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το φαινόμενο το ίδιο της σύναψης μιας συμφωνίας των κρατών μελών ε, εκτός των συνθήκων υπάρχει ανέκαθεν εξ αρχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή για να το πω κάπως αλλιώς οι Ευρωπαϊκές ε, Κοινότητες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν ήταν αποκλειστικό πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Πολλές λοιπόν από αυτές τις συνθήκες δεν είναι και τόσο σημαντικές και δεν επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της Ένωσης, αλλά είχαμε επίσης Ραδείγματα όπως αυτά που αναφέρθηκαν, τη συνθήκη του Σέγγεν, η σύμβαση του Σέγγεν και συμφωνία, η Προύμ, η συμφωνία Προύμ, που σχετίζονταν στενά με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, αλλά που εν γέννη συνέβαλαν στην ολοκλήρωση και δεν την απείλησαν. Τώρα βεβαίω έχουμε αυτές τις δύο νέες συνθήκες που και οι δύο υπογράφηκαν νωρίτερα φέτος και που συνδέονται με τις ε, κεντρικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλοί είπαν πως αυτό είναι πρόβλημα όχι μόνο από πολιτική και θεσμική πτυχή αλλά και από νομική άποψη. Ε, βέβαια είναι αλήθεια ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να συνάπτουν ό,τι συνθήκη θέλουν, όποτε το θέλουν και για οποιοδήποτε θέμα. Ε, πρέπει να λειτουργούν εντός των πλαισίων που απορρέουν από τις ε, ε, υποχρεώσεις τους με βάση το κοινοτική νομοθεσία. Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο έχει μια ρήτα στο άρθρο που αναγνωρίζει την προτεραιότητα του ευρωπαϊκού δικαίου ήταν μια ρήτρα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέμεινε να μπει μέσα στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο, ενώ το, η συνθήκη περί του στο μηχανισμού σταθερότητα δεν περιλαμβάνει τέτοια ρήτρα, αλλά ο ίδιος κανόνας ισχύει. Οι διεθνείς συνθήκες, ακόμα και ανάμεσα στα κρατη ποτέ δεν μπορούν να περιλαμβάνουν κανένα κανονισμό, καν, καμιά διάταξη που να είναι σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο εκκίνησης. Θα δούμε λοιπόν τέσσερα συγκεκριμένα ζητήματα σύντομα και να σας πω ότι Φυσικά αυτό που σας λέω εδώ είναι δική μου προσωπική άποψη, αλλά φαντάζομαι ότι για ορισμένα από αυτά τα ζητήματα θα υπάρξει ούτως ή άλλως απόφαση από το ε, δικαστήριο, από το ΔΕΚ, γιατί η υπόθεση Pringle που προέρχεται από το ε, Ιρλανδικό Ανώτατο Δικαστήριο και θίγει κάποια από αυτά τα ε, θέματα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την απόφαση πριν το τέλος του χρόνου, αλλά δεν είναι βέβαιο. Έχουμε λοιπόν εδώ τέσσερα ζητήματα. Το πρώτο αφορά ε, το γεγονός ότι οι συμφωνίες ανάμεσα σε κάποια, αλλά όχι όλα τα κάποια μελη σε, δεν επιτρέπονται σε θέματα που εμπίπτουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Ένωσης. Η νομισματική πολιτική είναι σε σχέση με τις ε, χώρες του ευρώ αποκλειστική αρμοδιότητα. Από το, αυτό προκύπτει από το άρθρο 3. Και επίσης στην υπόθεση Pringle η συνθήκη φαίνεται, μάλλον γνωρίζουμε, ότι η συνθήκη για το μηχανισμό σταθερότητας αφορά την νομισματική <coughs> πολιτική και άρα τα κρατημέλη δεν έχουν δικαίωμα να συνάψουν τη συνθήκη αυτή. Ωστόσο, αν δούμε το τίτλο της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, θα δείτε ότι το θέμα της οικονομικής βοήθειας προς τα κράτη-μέλη τοποθετείται όχι στο κεφάλαιο της νομισματικής πολιτικής, αλλά στο κεφάλαιο της οικονομικής πολιτικής. Η οικονομική πολιτική είναι κοινή αρμοδιότητα, δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα όπως γνωρίζουμε. Και εφόσον είναι κοινή αρμοδιότητα, τότε τα κρατημέλη έχουν το δικαίωμα να ασκούν τις δικές τους πολιτικές παράλληλα με τις ε, κοινοτικές πολιτικές. Δηλαδή μπορούν να τις ασκούν ε, μεμονωμένα ή και από κοινού, δηλαδή συνάπτοντας μια διεθνή συμφωνία όπως έπραξαν εδώ. Δεύτερο σημείο, δεύτερη επίκριση νομικού τύπου επίσης και σε σχέση με τη συνθήκη για τον μηχανισμό σταθερότητα έχει λεχθεί ότι παραβιάζει τον κανόνα περί μη διάσωσης, no bailout, το άρθρο 125 δηλαδή. Και ότι δηλαδή τα κράτη-μέλη δεν είναι υπεύθυνα για τις οικονομικές υποχρεώσεις άλλων κρατών μελών. Και γι' αυτό ακριβώς και ο μηχανισμός σταθερότητας δημιουργήθηκε, ώστε τα άλλα κράτη-μέλη να είναι το καθένα υπεύθυνο για τα χρέη του άλλου. Εμέσως και στο βαθμό της, κάθε, της συνεισφοράς του κάθε κράτους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι δύσκολο να πούμε ότι δεν θα υπάρχει διάσωση μέσα στο πλαίσιο του μηχανισμού σταθερότητα. Αφού αυτό είναι ο στόχος του, γι' αυτό φτιάχτηκε. Εδώ υπάρχει λοιπόν μια, μια α, σύγκρουση. Το νέο άρθρο 136 όμως, το οποίο θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου, θα άρει αυτή την, ε, την αντίφαση γιατί αυτό το άρθρο επιτρέπει ρητά τη δημιουργία ενός μηχανισμού συλλογικής οικονομικής στήριξης ως εξαίρεση από το γενικό κανόνα περί διάσωσης. Βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο δε πρωτογενούς δικαίου και θα αποτελεί μια εξαίρεση ε, για τον μηχανισμό σταθερότητα. Υπάρχει όμως ένα μικρό πρόβλημα προθεσμιών εδώ, γιατί ξέρουμε ότι η συνθήκη για το μηχανισμό σταθερότητα άρχισε να ισχύει πριν από λίγε μέρε, δηλαδή πριν να αρχίσει να ισχύει η προσαρμογή τη συνθήκη. Αν όμω είναι προπόθεση η τροποποίηση τη συνθήκη για να λειτουργήσει ο μηχανισμό σταθερότητα, θα πρέπει εδώ να προσέξουμε πάρα πολύ και θα ήταν σοφό τα νέα όργανα του Μηχανισμού Σταθερότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο κτλ. να περιμένουν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι ότου υιοθετήσουν το πρώτο τους πρόγραμμα στήριξης οποιασδήποτε χώρα γιατί μπορεί να υπάρχει πρόβλημα ασυνέπειας στο κοινοτικό δίκαιο. Τρίτο νομικό ζήτημα είναι τώρα σε σχέση με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο όπου ε, λέχθη ότι οι διατάξεις που αφορούν τη δημοσιονομική πειθαρχία και ισορροπία στα κάτι μέλη είναι στην ουσία επικαλυπτόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις πρωτογενούς ή δευτερογενούς ευρωπαϊκού δικαίου σε σχέση με τα ελλείμματα του προπολογισμού. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι η συνθήκη ορίζει το maximum deficit στο 3%, ενώ το Δημοσιονομικό Σύμφωνο το μειώνει στο 0,5% ή στο 1%, ανάλογα με τη χώρα. Ωστόσο, αν το σκεφτεί κανεί, είναι ότι ε, ε, ε, βλέπει ότι αυτές, αυτά, αυτά τα στοιχεία είναι διαφορετικά, αλλά όχι ασύμβατα. Δεν υπάρχει σύγκρουση γιατί η Ευρωπαϊκή Συνθήκη επιτρέπει στα κατημέλη ελεύθερα να κατέβουν και κάτω από το 3%. Μπορούν να φτιάξουν κανόνες ε, διατάξεις όπως η Γερμανία και η Ισπανία που ορίζουν χαμηλότερα το έλλειμμα. Και αυτό εδώ τους επιτρέπει να το κάνουν αυτό συλλογικά, μέσω του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Δηλαδή μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους να ορίσουν το μάξιμο με επίπεδο ελλείμματος χαμηλότερα από ό,τι στην συνθήκη. Υπάρχει εδώ λοιπόν διαφορά, αλλά όχι ασυμβατότητα. Τέλος, το επόμενο επίμαχο θέμα και ίσως και το πιο δύσκολο είναι αυτό το θέμα της ανάμεξης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο και στη Συνθήκη περί σταθερο... Μηχανισμού Σταθερότητας, όπως αυτό που ανέφερε ο Γιάννης προηγουμένως, δηλαδή ο δανεισμός των ε, ευρωπαϊκών θεσμών. Από πολιτικής άποψη είναι καλό, αλλά από νομικής μπορεί να είναι προβληματικό, γιατί καταρχήν οι αρμοδιότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ορίζονται από τις συνθήκες. Υπάρχει μάλιστα το άρθρο 30 που λέει ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λειτουργούν υπό το περιορισμό των αρμοδιοτήτων που τους ε, αποδίδονται από τις συνθήκες. για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να γίνει τώρα μια διάκριση ανάμεσα στη συμμετοχή του ΔΕΚ και τη συμμετοχή των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων. Για το ΔΕΚ ευτυχώς το, το πρόβλημα δεν είναι τόσο δύσκολο γιατί έχουμε ένα σύντομο άρθρο στη συνθήκη εξ αρχή από τη συνθήκη της Ρώμης που επιτρέπει στα κρατημέλη ε, υπό ειδική συμφωνία ανάμεσα στα μέρη να υποβάλουν οποιαδήποτε διαφορά έχουν στο ΔΕΚ. Και ακριβώς αυτό συμβαίνει τόσο με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο όσο και με τη συνθήκη για τον ε, Μηχανισμό Σταθερότητας. Πρόκειται για ειδικέ συμφωνίες ανάμεσα σε κάποια κρατημέλη που συμφωνούν μεταξύ τους να λύσουν τις διαφορές τους ανάμεσα τους το καλύπτεται νομίζω από το δίκαιο, το ευρωπαϊκό. Το θέμα είναι τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίω, που έχει σημαντικό ρόλο να παίξει κυρίω στο μηχανισμό σταθερότητα, όπου οι ιδέε τη Κομισιόν είναι να εφαρμοστούν τα προγράμματα οικονομικής στήριξης, δημοσιονομικής στήριξης. Πώς το κατανοούμε λοιπόν αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι αν κανείς εξετάσει προσεκτικά το, τις διατάξεις της που ανέφερε το, το 30, λέει ότι θα, 13 με συγχωρείτε, λέει ότι θα πρέπει να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Εκτελεστική Επιτροπή υπό, ε, στα όρια μάλλον των αρμοδιοτήτων της όπως ορίζονται από τις συνθήκες. Πρέπει να διαχωρίσουμε λοιπόν ανάμεσα στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα. Είναι δυνατόν να ανατεθούν νέα καθήκοντα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με άλλα μέσα. Για παράδειγμα μέσω μιας δευτερόνωσης συμφωνίας από τη στιγμή που αυτά συμβαδίζουν με τις ε, αρμοδιότητες αυτών. Στην περίπτωση της Κομισιόν, για παράδειγμα, η εφαρμογή μηχανισμού δημοσιονομικής στήριξης υπάρχει ίδιος ε, καθήκον και γνωρίζουμε ότι υπό τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας που φτιάχτηκε από τον κανονισμό του Συμβουλίου του 2010, που είναι μέσω δηλαδή του Ευρωπαϊκού Δικαίου, η Κομισιόν ανέλαβε, μάλλον τη ανετέθη, ε, ο ίδιος πάλι ρόλος το κάνει ήδη με την Ελλάδα, όπου ήδη ε, εφαρμόζει έναν μηχανισμό δημοσιονομικής στήριξης το να της ανατεθεί άλλη μια φορά αυτό το καθήκον, με το, μέσω δηλαδή της συνθήκης μηχανισμού σταθερότητας, είναι απόλυτα συμβατό και άρα και νομικά ως αποδεκτό και επιτρεπτό. Συμπέρασμά μου λοιπόν και μετά από αυτή τη σύντομη ανάλυση και με την προπόθεση ότι αυτό θα εγκριθεί από το 10, θα επικυρωθεί από το 10, είναι ότι Ούτε το δημοσιονομικό σύμφωνο, ούτε ο μηχανισμός σταθερότητας δεν, είναι, δεν παραβαίνουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τουλάχιστον, όπως είπα, από την, αρχή, από την ημερομηνία ισχύω του άρθρου 36 από την 1η δηλαδή του 2013. Αν θα ήθελα να προσθέσω δύο ε, συμπεράσματα. Η νομική εκτίμηση την οποία εγώ σας υποβάλλω δεν σημαίνει ότι η επιλογή που έκαναν τα κρατημέλη να συνάψουν αυτές τις χωριστές ε, διεθνείς συμφωνίες ήταν η καλύτερη επιλογή που είχαν. Υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην νομική ανάλυση που πρέπει να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, ότι δηλαδή τα κράτη-μέλη έχουν την αρμοδιότητα, την εξουσία να συνάπτουν διεθνεί συμφωνίε μεταξύ του, και την πολιτική εκτίμηση του κατά πόσο είναι αυτό ο σοφό δρόμο, να βγει κανεί δηλαδή από την ευρωπαϊκή νομική τάξη, ένομη ε, τάξη και να. Αυτό είναι όμω άλλο θέμα. Το επόμενο όμως συμπέρασμα είναι ότι το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και το Μηχανισμό Σταθερότητας δεν ε, είναι απόλυτες, απόλυτη ε, θα εξαρτηθεί από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και πώ αυτή θα εξελιχθεί στο μέλλον. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, από τη στιγμή που τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα υιοθετήσουν νέα μέτρα, τα οποία θα έρθουν σε αντίφαση με το περιεχόμενο του δημοσιονομικού συμφέρονου ή του μηχανισμού σταθερότητα, θα αντικαταστήσουν αυτόματα τούτε εδώ τι συνθήκε. Γιατί αυτέ ε, ω χωριστέ διεθνεί συμφωνίε δεν θα είναι πια ε, συμβατές με, την με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αυτή η ρήτρια λοιπόν περί συμβατότητας είναι μια κινητή ρήτρα και αυτό είναι και ένα δίδαγμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ίσως δεν πρέπει να δαπανά την ενέργειά του καταπολεμώντας αυτές τις συνθήκες της τεχνής αλλά αντιθέτως ίσως να προσπαθήσει να τις αντικαταστήσει σε ένα μεγάλο βαθμό. Να το επαναπατρίσει το περιεχόμενο δηλαδή μέσα στην νομικό πλαίσιο της Ένωσης μέσω της υιοθέτησης ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ώστε αυτά να θεωρηθούν πλέον ε, ασύμβατα. Οι νομικές προϋποθέσεις για να συνάπτονται ξεχωριστές διεθνείς συμφωνίες επίσης ισχύουν για οποιαδήποτε μελλοντική προσπάθεια για πιο φιλόδοξες δηλαδή διεθνείς ε, ε, συμφωνίες όπως αυτές που συζητήθηκαν σήμερα το πρωί και που πιστεύω θα τις αναφέρει και ο Ζαν Κλοντ Πυρίς. Πρέπει να δούμε λοιπόν αν υπάρχουν σχέδια για σύναψη ε, τέτοιων χώρων συμφωνιών μεταξύ των κρατομελών και κατά πόσο είναι, αυτά είναι συμβατά με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτή είναι μια απόλυτη νομική προϋπόθεση και όρος και ε, πρέπει να εγκριθεί και από το ΔΕΚ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ καθηγητά Ντεβίτε και για την τήρηση του χρόνου σας. Και θα δώσω το λόγο στον καθηγητή Jean-Claude Piri, που είναι επίτιμος ε, καθηγητής του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που θα ολοκληρώσει αυτή την πρώτη σύνοδο με τη δική του παρέμβαση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά επιτρέψτε μου να πω πόσο με τιμά η παρουσία μου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω την ευκαιρία να ομιλώ ενώπιον της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων με την οποία είχα κάποιες επαφές ε, σε προηγούμενη ιδιότητά μου επί σειρά ετών. Θα ήθελα κυρίως να συγχαρώ την Επιτροπή σας, Εγκάρδια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους βουλευτές που ενδιαφέρθηκαν για αυτά τα θέματα και ασχολήθηκαν με τη διοργάνωση διότι θεωρώ ότι είναι εξαιρετική πρωτοβουλία και άκρος επίκαιρη ε, για να συζητήσουμε σήμερα για αυτά τα θέματα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Το θέμα που μου ανατέθηκε έχει ως εξής ποιες θεσμικές λύσεις θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί για να διαχειριστούμε ε, τη διακυβέρνηση πολλαπλών ταχυτήτων χωρίς να αλλάξει το παρόν θεσμικό πλαίσιο των βασικών συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα βασιστώ σε μια διπλή αφετηρία αν θέλετε. Αφενός, είναι νομίζω γενική αποδοχή, αναδυόμενη μεν, πλην όμως όλο και πιο ισχυρή για τον τρόπο με τον οποίο ε, μπορεί να λυθεί με βιώσιμο τρόπο η σημερινή κρίση του ευρώ. Ανεξάρτητα από την ανάγκη διασώσεων, τυχών ή συγκεκριμένων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, στη ε, γραμμή της απόφασης που έλαβε 6 Σεπτεμβρίου το Συμβούλιο ε, των διοικητών. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να ισχυροποιηθεί η Ευρωζώνη και να γίνει γνήσια ο ναι. Ε, το νομισματικό σκέλος είναι δεδομένο, το οικονομικό δεν υπάρχει, χωλαίνει η υπόθεση και θα πρέπει αυτό να αναταχθεί. Και στις 28-29 Ιουνίου το Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά. Αυτή είναι η πρώτη μου αφετηρία, δεύτερη αφετηρία. Για να φτάσουμε λοιπόν σε αυτή την ονέ ναι της Ευρωζώνης, φαίνεται πολιτικά αδύνατο σήμερα, έτσι πιστεύω, μπορώ να το πω, να τροποποιηθεί η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν θα υπάρξει ομοφωνία των 27 απλούστατα. Αυτή τουλάχιστον είναι προσωπική μου γνώμη. Αντίθετα, οι 17 της Ευρωζώνης θα μπορούσαν κάλλιστα να προχωρήσουν χωρίς τροποποίηση των βασικών συνθήκων της Ένωσης, υπό τον όρον βεβαίως ότι αυτό θα γίνει με τρόπο συμβατό με τις συνθήκες. Εάν λοιπόν αυτή η διπλή αφετηρία ως παραδοχή ισχύει, ε, μπορούμε να σκεφτούμε δύο είδους λύσεις. Δύο, δάμε, συγγνώμη. Είτε οι 17 θα ε, ενοποιηθούν περισσότερο, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες ενισχυμένης συνεργασίας που παρέχει το σημερινό πλαίσιο των συνθήκων, χωρίς να χρειαστεί να συναυθεί οποιαδήποτε νέα συνθήκη, νομίζω αυτό είπε ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη προηγουμένως, είτε η δεύτερη δυνατότητα να συμπληρωθεί αυτό το πλαίσιο από ένα νέο είδος συνθήκης που δεν είναι τροποποίηση, γιατί φρονώ ότι πολιτικά αυτό είναι αδύνατο, αλλά να είναι μια πρόσθετη συνθήκη, λεγόμενη διακυβερνητική, για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Επιτρέψτε μου να κάνω εδώ μια μικρή παρένθεση για την ορολογία. Διακυβερνητική είναι ο όρος που χρησιμοποιείται προς μια κατεύθυνση ή προς άλλη, ανάλογα με την περίσταση. Εδώ απλώς πρόκειται για μια συνθήκη που δεν έρχεται να τροποποιήσει τις βασικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα χρησιμοποιεί διακυβερνητικές κλασικές μεθόδους, είτε λήψης αποφάσεων, που είναι πάντα η ομοφωνία ή η νέα συμφωνία, είτε για να ελέγχει και να εποπτεύει ε, την εφαρμογή από τις χώρες που συμμετέχουν. Και αυτό μπορεί να ανατεθεί σε ένα δικαστήριο ή στο ΔΕΚ με δύο λόγια θα ήθελα να σας περιγράψω τις δύο αυτές δυνατότητες. Δυνατότητα πρώτη, τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη διαδικασία ενισχυμένη συνεργασίας που ε, παρέχουν σήμερα οι συνθήκες. Το είπαν και πολλοί προαλήσαντες, Η βάση ε, ουσιαστικά είναι το άρθρο 136 και ε, ενδεχομένω και το 138 για τις συνθήκες για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό τον όρο να συμμετάσχουν και οι 17 και στα πλαίσια ε, του πεδίου εφαρμογή αυτών των συνθήκων να είναι καλύτερη νομική βάση για να δρουν εδώ τα κράτη. Και όπως είπαν και πολλοί ομιλητές, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γενικές διατάξεις των συνθήκων για την ενισχυμένη συνεργασία με τον όρο να συμμετέχουν κάθε φορά τουλάχιστον 9 κράτη-μέλη και μετά να συμπληρώνονται τα δύο άρθρα που σας ε, προανέφερα για να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία. Αυτή ε, η επιλογή, και επιτρέψτε μου να περιγράψω λίγο τα υπέρ και τα κατά της, αυτή η επιλογή προφανώς ε, έχει πολλά εκτίματα. Και μάλιστα προφανή ε, είναι αμέσου εφαρμογής. Καμία νέα συνθήκη δεν χρειάζεται να συναυθεί, να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις γνωστές δυσκολίες για να καταλήξει κανείς και να κυρώσει και σε 17 κράτη-μέλη. Από την άλλη, ε, οι θεσμικές διατάξεις των συνθήκων βρίσκουν άμεση και πλήρη εφαρμογή. Όλα τα θεσμικά όργανα παίζουν το ρόλο τους με την πλήρη του σύνθεση χωρίς να αλλάξουν τίποτα. Και στο Συμβούλιο ε, μόνο οι εκπρόσωποι των κρατών ε, μελών ε, συμμετέχουν και ψηφίζουν, άρθρο 136 με τη γνωστή διαδικασία. Αντίθετα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχουν και αποφασίζουν και σέβονται όλη τις διαδικασίες, οι οποίες υφίστανται τον κανονικό έλεγχο της Κομισιόν και του ΔΕΚ. Ωστόσο, πιστεύω ότι υπάρχει σε αυτή την επιλογή και μειονέκτημα ή μειονεκτήματα. Επί της ουσίας θα πρέπει να δούμε ότι σέβεται το σημερινό πρωτογενές δίκαιο. Δηλαδή δεν υπάρχει νομική δέσμευση των κρατών αυτών να ε, ολοκληρώσουν την οικονομική ένωση. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν αναγκαστικά σύγκληση των δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών, αλλά ε, νέα εκχώρηση αρμοδιοτήτων, τις οποίες θα μοιράζονται τα κράτη-μέλη, με το Ευρωπαϊκό Κέντρο. Αυτή η εκχώρηση όμως αρμοδιοτήτων δεν προβλέπεται από τις συνθήκες. Και επίσης δεν πιστεύω ότι είναι αρκετό αυτό ούτε πολιτικά για να πιστούν οι λαοί, οι πληθυσμοί και οι χρηματαγορές που χρειάζονται να πιστούν, ούτε οικονομικά για να επιτύχει, γιατί δεν υπάρχει νομική δέσμευση με την ε, απειλή κυρώσεων. Από την άλλη, στο θεσμικό πλαίσιο, τα κράτη που συμμετέχουν ενδεχομένω να έχουν πολιτικές δυσκολίε να δεχθούν ότι οι αποφάσεις που τους αφορούν αποκλειστικά θα λαμβάνονται, αφού θα προτείνονται από μια Κομισιόν και ένα Κοινοβούλιο που συντίθενται από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαρτίζονται και έχουν αρμοδιότητες και εξουσίες που αυτή τη στιγμή είναι εθνικές και όχι κοινοτικές ή ενωσιακές. Έρχομαι τώρα στη δεύτερη επιλογή. Τα κράτη της Ευρωζώνης ε, συνάπτουν επιπλέον διακυβερνητική ε, συνθήκη επιπλέον των βασικών συνθήκων για να έχουν μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Αυτή η επιλογή θα επέτρεπε στα συμμετέχοντα κράτη να ενέχονται νομικά, να δεσμεύονται, να δημιουργήσουν μια πραγματική οικονομική ένωση. Επιπλέον συνθήκη βεβαίω θα χρειαζόταν πολύ χρόνο για τη διαπραγμάτευση, την έγκριση, την κύρωση από τα 17 κράτη-μέλη και την εφαρμογή στη συνέχεια. Πολλό δε μάλλον που για την κύρωση θα μπορούσε, ανάλογο με το περιεχόμενό της, να επιφέρει τροποποιήσεις ε, κάποιων συνταγμάτων στα κράτη-μέλη, που πράγμα επίσης ε, χρειαζόταν ενδεχομένως και δημοψηφίσματα, εκτός από την έγκριση των Εθνικών Κοινοβουλίων. Βραχυπρόθεσμα όμως μια απόφαση αρχής ε, να ακολουθηθεί αυτή η κατεύθυνση, ενδεχομένως αν ήταν αρκετά σαφής, θα μπορούσε να πείσει και τους λαούς και τις χρηματαγορές ότι έχουμε εδώ μια λύση που μπορεί να είναι και βιώσιμη και εφικτή, αλλά και ε, που επίκειται. Και αυτό θα επέτρεπε την κατάσταση να καταπραϊνθεί λίγο μέχρι να ληφθεί απόφαση. Τώρα, αν ευσταθεί νομικά αυτό, στο μέτρο που όπως πολύ ωραία εξήγησε ο Μπρίνο Ντεβίτε η επιπλέον συνθήκη θα ήταν συμβατή με τις υφιστάμενες ε, συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα επιβεβαίωνε την υπεροχή τους και την ε, κυριαρχία τους δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Η βασική δυσκολία βεβαίως είναι εδώ πολιτική και μίζων μάλιστα. Δηλαδή θα χρειαζόταν υποστήριξη των πληθυσμών, των λαών και των εθνικών κοινοβουλίων σε ένα πολιτικό πλαίσιο άκρος δυσχερές. Επίσης, ταυτόχρονα θα έπρεπε, και μάλιστα όχι ταυτόχρονα, προηγουμένως θα έπρεπε να συμφωνηθεί το θεσμικό πλαίσιο. Και εδώ, ε, κυρίως θέλω να σταθώ. Υπό την έννοια αυτή θα ήταν βεβαίως ε, προτιμητέο ε, η νέα συνθήκη να μην δημιουργήσει κανένα νέο θεσμικό όργανο. Αρκετά περίπλοκη είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και αρκετά δυσνόητη λειτουργία της για τους πολίτες. Σε ό,τι αφορά τώρα κάποιου θεσμού, ε, θεσμικά όργανα, το ελεγκτικό συνέδριο, το ΔΕΚ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, νομίζω ότι αυτά τα θεσμικά όργανα θα μπορούσαν με τη σύμφωνη γνώμη και των 27 να συμμετέχουν στην εφαρμογή ε, μια επιπλέον συνθήκη χωρί να αλλάξει τίποτα, ούτε στο καθεστατικό του, ούτε στη σύνθεσή του. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο και πάλι δεν βλέπω δυσκολία. Ήδη συνεδριάζουν ε, de facto, όπω το γνωρίζετε, σε επίπεδο Ευρωζώνη και αρχηγή κρατών και κυβερνήσεων, αλλά και οι Υπουργοί Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας. Εκεί που δυσκολεύουν τα πράγματα είναι στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά, και το θυμίζω, τα ζητήματα που σήμερα είναι αρμοδιότητες των κρατών μελών. Για λόγους νομικούς, και έρχομαι στην κριτική του κυρίου Γουαλτιέρη προηγουμένως, άρθρο 10, παράγραφος 2, άρθρο 10 παράγραφος 4 για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα επεκταθώ. Αλλά και για πολιτικούς λόγους φαίνεται δύσκολο κατά την άποψή μου, συμφωνώ δηλαδή εδώ με τον κύριο Γουαλτιέρη, να εκχωρηθεί ο δημοκρατικός έλεγχος μόνο στους ευρωβουλευτές που εκλέγονται στα κράτη της Ευρωζώνης. Αυτό ορισμένοι το σκέφτονται. Ε, θα μπορούσαν επίσης οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών να μην θέλουν έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του. Η λεγόμενη έκθεση Βέστερβέλε που είναι έκθεση 11 υπουργών εξωτερικών, 11 κρατών μελών, εκ των οποίων 9 συμμετέχουν στην Ευρωζώνη και έχει τη σημασία του αυτό. Η έκθεση για το μέλλον της Ευρώπης που δημοσιεύθηκε μέσα Σεπτεμβρίου από την πλευρά τους τα ίδια τα εθνικά κοινοβούλια θα μπορούσαν να απαιτήσουν ως αντάλλαγμα της συμφωνίας τους εκχώρησης ορισμένων εξουσιών τους και μάλιστα των πιο ουσιαστικών και των πιο ευαίσθητων που είναι η οικονομική και δημοσιονομική πολιτική. Λοιπόν, αν εκχωρήσουν ορισμένες από αυτές τις εξουσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα εθνικά κοινοβούλια θα μπορούσαν να απαιτήσουν ως αντάλλαγμα να έχουν με τον τρόπο που θα συμφωνηθεί ε, τη δυνατότητα ελέγχου των αποφάσεων που θα λαμβάνονται στο μέλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πιο ουσιαστικά ακόμα θα μπορούσαν να στηρίξουν την εξή θέση λέγοντας ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχουν αρκετή εξουσία γιατί δεν ψηφίζουν φόρους. Και από την άλλη υπάρχει και το νομικό επιχείρημα που λέγει ότι είναι αρμοδιότητες αυτές και εξουσίες ε, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά των κρατών μελών. Είναι εθνικές εξουσίες και αρμοδιότητες των κρατών μελών ενώ που συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία. Και δεν ε, δημιουργείται νέα ευρωπαϊκή αρμοδιότητα με τη νέα συνθήκη. Στο βιβλιαράκι στο οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως αναφέρω ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια αντιπροσωπεία ε, των κρατών που συμμετέχουν και ε, των μελών ας πούμε της Επιτροπής Προϋπολογισμού της κάθε χώρας και για να μην έχουμε διπλές ευρωεκλογές που θα ήταν και γελίο, άλλωστε και ο κόσμος δεν θα καταλάβαινε, ε, αυτές οι αντιπροσωπείες θα μπορούσαν να αναλάβουν με βάση την επιπλέον συνθήκη σημαντικές εξουσίες συν απόφαση σύμφωνης γνώμης, δεν ξέρω πώς θα ονομαστεί αυτό, μπορούμε να το συμφωνήσουμε, για τις σημαντικές αποφάσεις που θα λαμβάνονται στους νέους πλέον τομείς που θα καλύπτονται από αυτή τη συνεργασία και ε, που έχουν να κάνουν σήμερα με εθνικές αρμοδιότητες. Ε, μια άλλη πρόταση στην έκθεση Παντό Όπα, κάποιο μίλησε προηγουμένως γι' αυτό, για την Ευρώπη μας. Ε, συμμετείχα κι εγώ στην ε, σύνταξη αυτή της έκθεσης και πρόσφατα δημοσιεύτηκε. Εκεί λοιπόν προτείνεται να δημιουργηθεί ένα όργανο που να απαρτίζεται από 17 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εντάξει, δεν κατονομάζεται ε, η καταγωγή τους και από 34 εθνικούς βουλευτές. Βλέπε εδώ συνεργασία εθνικών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό το προβλέπει τόσο η συνθήκη της Λισαβόνας, το άρθρο 9 για τον πρωτόκολλο, για το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά και στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο προβλέπεται αυτό. Στο άρθρο 13 ε, της ε, Δευτέρας Μαρτίου 2012. Πρόεδρε, είναι σαφές ότι η συζήτηση εδώ θα γίνει με πολύ πάθος, αλλά είναι και πάρα πολύ ουσιαστική. Όπως είπε πολύ πρόσφατα όλοι η ΡΕΝ Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η βαθύτερη ολοκλήρωση θα πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρή δημοκρατική νομιμότητα. Βέβαια, απομένει να δούμε ποιο τρόπο. Και έρχομαι τώρα στη δυσκολία που αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εγώ διερωτώ με αν οι κυβερνήσεις των 17 χωρών θα μπορούσαν να δεχτούν να διαδραματίσει τον πλήρη ρόλο τους και για τις 17. Δεν είναι βέβαιο, μπορεί. Ε, ενδεχομένως κάποιες χώρες να εμφανίσουν ε, δισταγμούς και επιφυλάξεις. Από 27 και για 27 ε, απαρτίζεται αυτό το θεσμικό όργανο και μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με απλή θυμίζω πλειοψηφία σε τόσο λεπτά θέματα. Τούτου λεχθέντος είναι προφανές ότι αποκλείεται απολύτως και δεν το συζητάω καν να δημιουργηθεί ένα νέο θεσμικό όργανο σαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παράλληλα με ό,τι σημαίνει αυτό για οικονομικούς, ανθρώπινους πόρους κτλ. Θα μπορούσε από την άλλη να δημιουργηθεί μια μικρή δομή πολιτικοδιοικητική, περισσότερο πολιτική κατά τη γνώμη μου παρά διοικητική, που θα μπορούσε να ονομαστεί Υπουργό Οικονομικών της Ευρωζώνης, όπως αναφέρουν ορισμένοι και θα ήταν επιφορτισμένο αυτό το όργανο με τον έλεγχο της εφαρμογής των αποφάσεων και την προσφυγή ενδεχομένως στο ΔΕΚ σε περίπτωση παραβίασης. Αυτό το όργανο, αυτή η αρχή ε, θα απαγορευόταν να δημιουργήσει μια νέα γραφειοκρατική δομή. Άρα, κατά ανάγκη θα πρέπει να αναθέτει την προετοιμασία ε, των αποφάσεων σε άλλα θεσμικά όργανα. Και να σας κάνω εδώ μια μικρή πρόταση, αν μου επιτρέπετε. Θα μπορούσε να αναθέτει αυτή τη λειτουργία, αυτή την προετοιμασία ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπό την προπόθεση βεβαίως ότι θα τη δεχτούν 27, αλλά την Επιτροπή όπως έχει σήμερα. Αυτό το σύστημα ε, θα ήταν πολύ κοντά στο θεσμικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, σας υποσχέθηκα να είμαι σύντομος, δεν θα επιμείνω, μια επιπλέον συνθήκη των 17 θα έπρεπε οπωσδήποτε και το υπογραμμίζω οπωσδήποτε να περιλαμβάνει ε, κατάλληλες διατάξεις για να προστατεύονται αποτελεσματικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των υπολείπων κρατών μελών που δεν συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν ακόμα στην Ευρωζώνη ή υπό τον έλεγχο του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Και για να υπάρχει και ένα ε, καθεστώς ε, ενεργού παρατηρητή ε, μεταξύ των κρατών εκείνων που δεν συμμετέχουν αλλά θέλουν το συντομότερο να μπουν στο ευρώ. Επίσης και τέλος, αυτή η συνθήκη θα πρέπει να περιλαμβάνει και αντίστοιχε πρόνοιε για να διαφυλάσει και τις εξουσίες αλλά και την ενότητα, την ένωση, τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ακαιρεότητά της. Η Ευρωζώνη δεν θα είναι μια αυτόνομη διακριτή οργάνωση θα εξακολουθεί να είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, σας ευχαριστώ, καθηγητά Πυρίς. Ξέρω πως εσείς πρέπει να μας αφήσετε σύντομα, οπότε θα σας ε, συμβούλευα να μείνετε εδώ στα έδρανα αυτά για να απαντήσετε σε ερωτήσεις ή προτάσεις των συναδέλφων, ξεκινώντας με τους δύο εισηγητές που ζήτησαν ε, το λόγο ο συνάδελφος ε, τα Τσασκόφσκι και ο κύριος ε, Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ. Διάβασα τα βιβλία σας ε, για την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων και έχω την αίσθηση ότι την έκθεση την έγραψε ο Γιώστος Λίψιους και την ομιλία την έκανε ο Ζαν Κλωτ Πυρίς. Στο βιβλίο σας ήσασταν πολύ πιο ριζοσπαστικός από ό,τι στην παρουσίαση που μας κάνατε εδώ. Γιατί. Μήπως γιατί έχει μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα και στο μεταξύ το ξανασκεφτήκατε ή προσπαθήσατε σήμερα εδώ να είστε λιγότερο α, κατηγορηματικός. Γιατί είπαμε στην αρχή ότι ίσως δεν είναι καλή ιδέα να δημιουργήσουμε νέα θεσμικά όργανα και νέους θεσμούς γιατί θα επιτείνουμε τη σύγχυση. Ε, στο βιβλίο σας το σημείο αφετηρία, δεν θέλω βέβαια να το συζητήσουμε εδώ, δεν έχουμε χρόνο για κάτι τέτοιο, είναι ότι το σημείο αφετηρία στο βιβλίο είναι ότι τα περισσότερα προβλήματα απορρέουν από τη διεύρυνση και από την υπερβολική ποικιλομορφία και διαφορετικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαφοροποίηση. Και επίσης ε, κάνετε και συγκεκριμένες κριτικές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ίσως να επανέλθουμε στην παρουσίαση του Γιάννη Εμμανουλίδη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε εντός ε, του συνταγματικού και του θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο μέτρο του δυνατού. Και ακόμη και όταν ε, ε, διαπραγματευόμαστε, εντάξει παρά είναι βαρύγδουπη αυτή η διατύπωση, όταν συμμετέχουμε στη διαδικασία διαπραγματεύσεων για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, Προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε το δημοσιονομικό σύμφωνο με τρόπο ώστε να μπορεί να συμπεριληφθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη. Ακριβώ για να αποφύγουμε τη δημιουργία νέων θεσμικών οργάνων, νέων θεσμών και νέων συνθηκών που θα είναι τελείω εκτό του νομικού πλαισίου και τη Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη, τη Ένωμη Τάξη των Συνθηκών. Παρόλο που μερικοί επιθυμούσαν τη δημιουργία νέων θεσμών, εμεί το αποτρέψαμε, προσπαθήσαμε να το περιορίσουμε και μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσπαθήσαμε να, διασ... να διασφαλίσουμε την ακαιρεότητα του συστήματος και επίσης ε, ε, η sunset clause ε, που επιτρέπει στη συνθήκη να αποτελέσει τη με της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τάξης είναι σημαντική προσπαθούμε να εφαρμόσουμε κοινοτικέ μεθόδους ε, στην εφαρμογή της συνθήκης και αν οι μελλοντικέ εξελίξεις ε, μας επιτρέψουν να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο που κατά τη γνώμη είναι ο καλύτερος, ε, πιστεύω ότι ακόμη και αν εφαρμόσουμε την α, διευρυμένη συνεργασία δεν θα πρέπει να παραβιάσουμε τη συνθήκη για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, για τα δικαιώματα και τι υποχρεώσει αυτών που είναι εντός και εκτός ευρωζώνη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κατά πόσο είναι εφικτό να δημιουργήσουμε παράλληλου θεσμούς. Μιλούμε για την νομοποίηση, μιλούμε για το πώς αντιμετωπίζει η κοινή γνώμη οι πολίτες στο θέμα αυτό και πώς ε, μας βλέπουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αν ε, ακολουθήσουμε μια κατεύθυνση ε, και δημιουργούμε όλο και περισσότερα θεσμικά όργανα και νέους θεσμούς, ε, τότε είναι που θα απομακρυνθεί τελείω από εμά ο κόσμο. Δεν θα καταλαβαίνει τι κάνουμε. Είδατε τι συνέβη με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Στι διαπραγματεύσει για τη συνθήκη τη Λισαβόνα προσπαθήσαμε να παρακάμψουμε τα προβλήματα αρμοδιοτήτων και θεσμών ε, που δεν ήταν και πολύ σαφείς. Αλλά παρόλα αυτά δημιουργήσαμε νέα προβλήματα. Και το θέμα των νέων θεσμών και το θέμα της ένταξής τους ε, ή της μη ένταξής τους στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα αποφύγουμε τις συγκρούσεις. Είδαμε το σχέδιο Φουσέ, η προσπάθεια να δημιουργηθεί κάτι τελείως καινούριο, μια νέα γραμματεία, νέοι θεσμοί ε, εκτός της, ενο... Ε, εκτός ευρωπαϊκής κοινότητας τότε, ακριβώς επειδή τα κράτη-μέλη, μερικά κράτη-μέλη ήταν δυσαρεστημένα με την κατάσταση. Ή το θέμα της ανάμειξης των εθνικών βουλευτών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για κάτι τέτοιο. Πριν τη συνθήκη του Μάστριχτ, οι εθνικοί βουλευτές ε, ε, συμμετείχαν άτυπα στη διαδικασία και τους προσκαλούσαμε στις συζητήσεις ε, για τον προϋπολογισμό. Για παράδειγμα, στην Πολωνική Προεδρία είχαμε συζητήσεις τακτικές μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Έχουμε τρόπους να αναμίξουμε ήδη τα Εθνικά Κοινοβούλια. Τώρα να δημιουργήσουμε νέα θεσμικά όργανα, νέους θεσμούς και να ε, ε, διασπάσουμε την ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δημιουργήσουμε μια νέα γραμματεία, θα δημιουργήσει τεράστια νέα προβλήματα για τις σχέσεις μεταξύ των νέων θεσμικών αυτών οργάνων. Και όχι μόνο θα γίνει ακόμη πιο σαφέ το έργο μας, αλλά θα είναι αδύνατο πια να το εξηγήσουμε και στου ευρωπαίου πολίτε. αλλά και η συνολική λειτουργία του συστήματος όχι μόνο θα επιδεινωθεί, αλλά θα καταστεί τελείω ανέφικτη. Βέβαια, μιλήσατε στο βιβλίο σας ότι θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και προσπαθούμε να μην δραματοποιούμε τα πράγματα. Πώς όμως ε, θα εξασφαλίσουμε ε, την αποφυγή αυτού του κατακαιρματισμού της ακεράτας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και τώρα έχουμε προβλήματα με τη διευρυμένη συνεργασία, την ενισχυμένη συνεργασία. Δεν θέλουμε η ενισχυμένη συνεργασία να παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο. Αν δημιουργήσουμε όμως ακόμη ένα νέο, ε, νέους ε, θεσμούς, θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση. πιστεύετε ότι θα πρέπει να εθετήσουμε την πιο ριζοσπαστική μέθοδο μεταξύ των δύο συστημάτων ή πώς μπορούμε, κατά τη γνώμη σας, συμφιλιώσουμε τα, τα διάφορα θεσμικά όργανα, αυτά που είναι εκτός του νομικού πλαισίου και αυτά που βρίσκονται εντός του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Γουαλτιέρη. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω κάποια σχόλια αρχικά του Μπρούνο Δεβίτε. το, πρόβλημα, το, κοινοβούλιο δεν έχει πρόβλημα, δεν, δεν είναι το πρόβλημά του να επιτεθεί κατά των διακυβερνητικών συνθήκων. Το θέμα είναι να δούμε αν κάτι τέτοιο θα είναι καλή επιλογή για το μέλλον. Και βλέπω εδώ ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι Πώ δεν είναι νόμιμε οι συνθήκε. Το με τα επιχειρήματά σα. Είναι όμως αποτελεσματικές λύσεις. Και εδώ είναι σκόπιμο να δούμε τη συνθήκη για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Είναι πραγματικά δεσμευτική αυτή η συνθήκη. Για να μην αναφερθώ στο γύρο Plus, γιατί όλοι συμφωνούν ότι δεν είναι δεσμευτική, δεν δίνει καμία προστιθέμενη αξία. Όμως το Δημοσιονομικό Σύμφωνο να δω τη δική σας παρατήρηση ξεκινώντας. Πρόκειται για τη μόνη νομική αντίφαση λόγω των κυρώσεων. Είναι δεσμευτική εφόσον υπάρχουν κυρώσεις. Έχουμε το άρθρο 8, όπως σωστά είπατε, το 273 που προβλέπουν το 10. Το πρόβλημα όμως δεν είναι το 8.1 της συνθήκης, είναι το 8.2. Διότι το 8.2 Ε, εμπλέκει και το άρθρο 260 της συνθήκης που λέει ότι αν σύμφωνα με το 7.3 τα κράτη δεν συμμορφούνται προς την απόφαση του ΔΕΚ, τότε μπαίνει σε ισχύ το 2.60 και τότε ε, μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις. Μπορείτε να μου πείτε αν είναι αυτό νόμιμο. Είναι παράνομο βεβαίως, γιατί αν διαβάσουμε το 2.60 λέει για θέματα που σχετίζονται με τις συνθήκες. Αυτό είναι ο πυλώνα του δημοσιονομικού συμφώνου. Εφόσον δεν υπάρχουν ακυρώσει, ποια είναι η αξία αυτού του συμφώνου. Καμιά. Εγώ δεν νομίζω πω είναι επικίνδυνο. Είναι απλώ άχρηστο. Είναι κάτι το οποίο δεν προσθέτει απολύτω τίποτα. Είναι μια δέσμευση ότι θα τηρήσουμε, λέει, το νόμο, ότι το δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το οποίο είναι πολύ πιο δεσμευτικό από τη διακυβερνητική συνθήκη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι ότι είναι παράνομο. Επίση, θα ήθελα να συζητήσουμε αυτό που είπατε ότι Υπάρχει μια αντίφαση στο θέμα. Υπεροχή λοιπόν του ευρωπαϊκού δικαίου. Από τη μια πλευρά λέμε μπορούμε να, έχουμε, ε, να αναλάβουμε επιπλέον δέσμευση υπό τη διακυβερνητική συνθήκη. Προσθέτουμε 0,5. Είναι επιπλέον του 1% του εξαπλού πακέτου που λέει ότι αυτό ισχύει μόνο για χώρες που είναι κάτω από το 60% στο χρέος. Δηλαδή είναι θέμα το πώς θα ερμηνεύσουμε το πολύ κάτω, το significantly below. Τι είναι αυτό το 0,1%, τι είναι, για ποιους. Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί το Δημοσιονομικό Σύμφωνο λέει κάτι που δεν είναι δυνατό να μετρηθεί. Για χώρες λέει που είναι πολύ κάτω από το 7% ε, ε, ε, και τα λοιπά. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο ούτε γλωσσικά ούτε γλωσσικά ούτε νομικά. Αν το ευρωπαϊκό δίκαιο περάσει από το 0,5 στο, 2, στο 1% ή στο 1% ή στο 2%, το θέμα είναι πώς ερμηνεύουμε το θέμα. Ε, όσο πιο χαμηλά τόσο καλύτερα. Αν θεωρούμε πως η δημοσιονομική πολιτική είναι μια πολιτική που προσφέρει διάφορες επιλογές, τότε το επιχείρημα του να προχωρήσουμε περαιτέρω δεν, είναι, δεν προχωράει πραγματικά περαιτέρω, απλώς είναι αντιφατικό. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι και το σημαντικό γιατί δεν είναι δεσμευτικό, γιατί δεν μπορεί να επιβληθεί καμιά κύρωση. Δεύτερη παρατήρηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ διάβασα προσεκτικά το βιβλίο σας, άκουσα τις ομιλίες σας. Έχω λοιπόν μια ερώτηση. Για πώς πάρουμε το παράδειγμα του γράφου Νότρε Europe. Λέμε για δύο χώρες της Ευρωζώνης όπου το Εθνικό Κοινοβούλιο και θα επιλεγεί ανάμεσα σε άλλα και εδώ βλέπω προβλήματα ανάμεσα στους εθνικούς βουλευτές γιατί υπάρχει, γίνεται διάκριση ανάμεσά τους. Και λέει 17 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρει από το Λουξεμβούργο, τρει από την Ολλανδία κτλ. Και εδώ θα, αυτό το σώμα θα έχει λέει αρμοδιότητες. Τι είδου αρμοδιότητε θα ψηφίζουνε και θα λαμβάνουν επιφάσεις, αποφάσεις δεσμευτικές και η, ψήφος του, η ψηφοφορία θα είναι τρεις από τη Μάλτα, τρεις από τη Γερμανία και τρεις από την Ολλανδία και αυτό είναι πιο νόμιμο, πιο νομιμοποιημένο, πιο θεμητό από ότι η ψήφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το διπλό πακέτο που μπορούμε με πλειοψηφία να τροποποιήσουμε το διπλό πακέτο ενώ το Συμβούλιο μιλούσε για τους 17. Αναγνωρίζω ότι δεν είναι η τέλεια λύση η ασυμμετρική ψήφος για το, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν καταλαβαίνω και δεν βλέπω άλλη καλύτερη λύση μέχρι ότου αλλάξει η συνθήκη. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πολύ καλά πώς αυτή η διάσκεψη, ακριβώς επειδή δεν θέλουμε να φτιάξουμε ακόμα ένα μεγάλο κοινοβούλιο. Ποτέ δεν μπορούσε να σεβαστεί οποιαδήποτε λογικότητα, τόσο όσον αφορά την εθνικότητα αλλά και τις πολιτικές οικογένειες. Κάτι τέτοιο λοιπόν θα κατέληγε να είναι πιο θεμητό από το, ένα πραγμα... από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τι αρμοδιότητες θα δοθούν. Τι είναι η διάσκεψη, η διάσκεψη για να συζητήσουμε. Εντάξει, γι' αυτό είμαι υπέρ και να υπογραμμίσω ότι το δικάστρο 13 του Δημοσιονομικού Συμφώνου δεν προβλέπει πως μόνο τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου των συνυπογραφουσών χωρών θα συμμετέχουν, γιατί ακριβώς το 13 αναφέρεται στο άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου 1. Και βλέπουμε το στόχο βεβαίως. Είναι μια διεθνή συνθήκη όπου συμμετέχουν όλο, ολόκληρο το κοινοβούλιο. Αυτό το προηγούμενο λοιπόν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και συμφωνώ εν γέννη πως αυτή η συζήτηση δεν είναι πολύ χρήσιμη εκτός και αν συμφωνήσουμε στο τι σημαίνει περαιτέρω ολοκλήρωση, περαιτέρω αρμοδιότητες, τι είδους αρμοδιότητες λέμε εδώ πέρα, τι είδους ε, σημαντικότερο ρόλο της Ένωσης θέλουμε. Και εδώ επανέρχομαι στα όσα είπα στην αρχή, ότι δηλαδή αυτό το μεικτό μοντέλο που θεωρούμε την ολοκλήρωση ε, περισσότερη και εντονότερη ανάμειξη των, των εθνικών αρμοδιοτήτων μέσω από ένα θεσμό για σκοπούς διεθνούς συνεργασίας είναι το σωστό μοντέλο ή μήπως θα πρέπει να, το κάνουμε, να κάνουμε πιο απλή χρήση και διάκριση των ισχυουσών αρμοδιοτήτων. δίνοντας ε, πόρους από το μηχανισμό ιδίων πόρων που θα μπορούσε να προκύψει από την ε, προηγμένη ε, συνεργασία, για παράδειγμα, που θεωρείται τώρα υποχω... πια ως ένα αντίστοιχο του, των πόρων του GNI που θα είναι του, του ΑΕΠ που θα είναι δηλαδή αντικατάσταση ε, των ε, ιδίων πόρων και κάτι τέτοιο θα εμπόδιζε το ανάγκη. Μάλλον δεν, δεν θα υπήρχε έτσι ανάγκη να υπάρχει και ο μηχανισμό σταθερότητα κτλ. Δίκαιη κατανομή των πόρων ανάμεσα στα κράτη πολιτικά, κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή είναι. μη ρεαλιστικό γιατί βλέπουμε τις διαπραγματεύσεις για το σε πλαίσιο. Πάντως, να έχουμε ένα συντονισμό που να μην είναι δεσμευτικός, πολύ περιοριστικός σε εθνικό επίπεδο και την αντίφαση του, ότι εθνικά χρήματα χρησιμοποιούνται για ευρωπαϊκούς σκοπούς αλλά τα διαχειρίζονται τα εθνικά κοινοβούλια. Δεν αρκεί να λέμε περαιτέρω ολοκλήρωση. Πρέπει να συζητήσουμε για ποιο είδος ε, ε, ολοκλήρωση χρειαζόμαστε. Και τελευταία παρατήρηση. Δεν περιορίζομαι τώρα στον, την αναζήτηση της περαιτέρω συνεργασίας, της διευρυμένης συνεργασίας. Ε, θέλω να σας ρωτήσω το άρθρο 352 και όχι το 351 σε συνδυασμό με την ενισχυμένη συνεργασία του 136. Τίποτα στη συνθήκη δεν εμποδίζει να χρησιμοποιήσει κανείς τη ρήτρα ευελιξίας που σημαίνει νέες, αρμοδιο... Ε, νέες εξουσίες στα θεσμικά όργανα σε συνδυασμό με αυτά τα άρθρα. Δηλαδή η ομοφωνία θα είναι ομοφωνία ανάμεσα στους 17 ή ανάμεσα στους 20 για παράδειγμα αν είναι αυτό το πρότυπο της ενισχυμένης συνεργασίας σε πάντα με σεβασμό στις αρμοδιότητες και τις νομικές αρχές που είναι αναγνωρισμένες. Αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε ως μια ενδιάμεση λύση ανάμεσα στην αλλαγή της συνθήκης και την απλή χρήση της ενισχυμένης συνεργασίας του 136 για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε είναι, ποια είναι η ενίσχυση των ε, κατευθυντηρίων γραμμών, η ενίσχυση της εποπτείας κτλ. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι, ποια είναι η δική σας γνώμη για την νομική και για την πολιτική σκοπιμότητα. Πρόεδρος, έχω το πρόβλημα. Έχω πρόβλημα με το χρόνο. Και να βάλω σε τάξη τη συζήτηση. Ήδη έχουμε βγει εκτός του χρόνου. Έχω ακόμα τον συνάδελφο τάβ Λάινεν και Μπρόνς. Είπα προηγουμένως ε, στον ε, καθηγητή Πυρής ε, και που να κάτσει εδώ για να μπορέσει να απαντήσει. Αν πρέπει να φύγετε, καλύτερα να μας πείτε μια σύντομη απάντηση, γιατί ούτως ή άλλως ο προβληματισμός αυτός θα συνεχιστεί και θα πρέπει να αφήσουμε για το απόγευμα τη συζήτηση για το δεύτερο πάνελ, γιατί ήδη είμαστε στα όρια. Καθηγητά Πυρής, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια Σα ε, σας ζητώ συγγνώμη, ε, ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Μπροκ και τους άλλους ε, ευρωβουλευτέ που ζήτησαν τον λόγο. είμαι σε δύσκολη θέση γιατί πρέπει να πάρω το τρένο και να μεταβώ σε άλλη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω ελάχιστο δυστυχώ χρόνο και δυστυχώ δεν θα μπορέσω να παραμείνω στη συνέχεια τη συζήτηση. Σω πρέπει να οργανώσετε και νέα συζήτηση. Να απαντήσω λοιπόν εντάχει. Ναι, είναι αλήθεια ότι η σημερινή μου θέση και αυτό που υποστηρίζω σήμερα, όχι μόνο εδώ, αλλά και σε άρθρα που κάνω και σε διαλέξεις, ε, έχει ε, προχωρήσει, εξελιχθεί σε σχέση με αυτή τη θέση που είχα υποστηρίξει στο βιβλίο μου πριν 1,5-2 χρόνια. Γιατί στο μεταξύ έλαβαν χώρα κάποιες εξελίξει, είχα και πολλές επαφές και έκανα και εγώ κάποιο δρόμο και τροποποίησε τη θέση μου. Η σημερινή μου θέση είναι πραγματικά η προσωπική μου γνώμη όπως έχει εξελιχθεί μετά το βιβλίο που έγραψα. Θα ήθελα να πω ότι ε, αυτό που προτείνω εγώ είναι μια φεδεραλιστικη μέθοδος που προβλέπει μια σημαντική εκχώρηση αρμοδιοτήτων και αφορά τους πιο ευαίσθητους τομείς που βρίσκονται στο, στην καρδιά της κυριαρχίας πρόκειται για την υιοθέτηση του εθνικού προϋπολογισμού, πρόκειται για την ε, έγκριση της οικονομικής πολιτικής. Αυτό βρίσκεται στην καρδιά της κυριαρχίας ε, και γι' αυτό σας μίλησα. Φυσικά θα πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Και αν ισχύσει κάτι τέτοιο, αν δηλαδή ε, βλέπετε στην έκθεση «Νότχο Ευρώπη, η Ευρώπη μας υπάρχει ένα θέμα για τη διαχείριση του χρέους και την απώλεια της κυριαρχίας που είναι αντίστοιχη από τα χρήματα που χρειάζεται για την αποπληρωμή του χρέους σε σχέση με το ποσοστό του ΕΠ και όσο πιο μεγάλη είναι η αναλογικότητα τόσο χάνεται την κυριαρχία σας. Οπότε σταδιακά χάνετε όλη την κυριαρχία σας για την έγκριση του προϋπολογισμού σας μια και θα χρειάζεται πια το πράσινο φως από τον οργανισμό ή από τον Υπουργό Οικονομικών Βέβαια, δεν μπορεί να σας υποχρεώσει κανείς για κάτι τέτοιο, γιατί κάτι τέτοιο θα ανέτρεπε τα θεσμικά όργανα. Δεν θα είχατε όμως ε, βοήθεια αν δεν ε, υπακούετε στις εντολές. Οπότε, de facto, καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Οπότε αυτό το πέρασμα, στη... αυτή η μεταβίβαση κυριαρχία είναι ένα βήμα φεντεραλιστικό. Και Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφαιρεθούν σημαντικές αρμοδιότητες από τα Εθνικά Κοινοβούλια. είμαστε ρεαλιστές αγαπητοί κύριοι Ευρωβουλευτέ. Πιστεύετε ότι οι ομόλογοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια θα δεχτούν απώλεια, σημαντική, σημαντική απώλεια των εξουσιών τους χωρίς να έχουν πια λόγο, κανένα λόγο στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ε, φυσικά και δεν πρόκειται να δεχτούν κάτι τέτοιο. Η απόφαση όμως από εκείνους εξαρτάται. Θα πρέπει να δώσουν τη συμφωνία τους, ε, την ε, έγκρισή τους, παρόλο που μερικές χώρες προβλέπουν δημοψήφισμα για κάτι τέτοιο. Και αυτή είναι η βασική μας διαφορά. Πιστεύω ότι ε, για να είμαστε ρεαλιστές θα πρέπει να χρειαστούμε τη συμφωνία των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και εγώ προσωπικά, αυτό είναι προσωπική μου γνώμη όμως, πιστεύω ότι το θέμα, η συμβολή τη ε, δημοκρατική νομιμοποίηση που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αρκεί για τα ζητήματα αυτά. Δεν αρκεί μόνο η νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για πολλού και διάφορου λόγου. Δεν θα ψηφίσετε εσεί, δεν θα ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, τα φορολογικά μέτρα στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ή στη Γαλλία, για ευνόητου λόγου. Πιστεύω λοιπόν ότι για του δύο αυτού λόγου ε, είναι σημαντικό να προβλέψουμε κάτι διαφορετικό. Υπάρχει και η πρόταση του εγγράφου Νότου Ευρώπη, Ευρώπη μα. Δεν είναι δική μου προσωπική πρόταση. Ήταν μια συμβαστική λύση που καταλήξαμε στους, ε, με τους συντάκτες. Με ένα συνδυασμό των 17 και των 34. Επίσης, ε, ε, μια λύση που απορρέει από τα Εθνικά Κοινοβούλια ή από τις Επιτροπές Προϋπολογισμού. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις και λύσεις. Το βασικό είναι πάντως τα εθνικά κοινοβούλια να έχουν και αυτά το λόγο του στην όλη διαδικασία. Και επίσης για να αποφευθεί ο κατακαιρματισμός και η προσβολή της ακαιρεότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι ε, θεμελιώδη σημείο, δεν το είχα επισημάνει δεόντως στο βιβλίο μου, υπάρχουν πολλές λύσεις. Να ε, να αποφασίσουμε ξεχωριστή νομική ύπαρξη της ε, Ευρωζώνης ε, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, πολιτικών ελευθεριών, εμπορικής πολιτικής, όλα αυτά που απορρέουν από τη συνθήκη και που σε μια συμπληρωματική συνθήκη θα πρέπει να υπάγονται στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που στο οποίο θα μπορεί να προσφεύγεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οποιαδήποτε από τις 27 χώρες, όχι μόνο μία από τις 17 χώρες. Αυτά και σας ζητώ συγγνώμη, αλλά δυστυχώς πρέπει να φύγω. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Σίγουρα η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί και σε άλλη ευκαιρία. Τώρα θα πρέπει να συνεχίσουμε. θα δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας για να απαντήσουν. Αφού όμως ακούσουμε τους συναδέλφους πρώτα, τον κύριο Ντάφ. Πρόεδρε, καταρχάς επιτρέψτε μου να καλωσορίσω και εγώ τους ε, εξαιρετικούς ε, εμπειρογνώμονες καθηγητές μας και πρώην υπάλληλου που μας δίνουν τροφή για σκέψη σε αυτή τη τόσο σημαντική στιγμή. Ιστορική θα τη χαρακτήριζα και τη στιγμή και το δίλημα ε, που αντιμετωπίζουμε τη στιγμή που ομοσπονδιοποιούμαστε. Υπάρχουν δύο τεράστια προβλήματα. Το πρώτο είναι η έλλειψη κυβέρνησης. Δεν υπάρχει λόγος, δεν έχει νόημα να συζητούμε εδώ με ακαδημαϊκούς τρόπους ή με εφημισμούς για ε, διακυβέρνηση πολλαπλών ταχυτήτων ε, ή μια Ευρώπη πολλαπλών ταχυτήτων. Ενώ στο κέντρο του προβλήματος μας είναι ότι δεν υφίσταται ισχυρή, ε, όρημη, διακριτή ε, ε, δημοκρατική κυβέρνηση. Ιδιαίτερα για την πολιτική οικονομία. Έχουμε μια διάχυση τώρα αρχών, οργανισμών, υπηρεσιών, ε, θεσμικών οργάνων που προσπαθούν να συνεννοούνται μεταξύ τους, αλλά συχνά ανταγωνίζονται, αλλά και συγκρούονται μεταξύ τους είναι όλοι ενεχόμενοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ε, η Σύνοδος Κορυφής των χωρών της Ευρωζώνης, το Eurogroup, το Euroworking Group που προετοιμάζει το Eurogroup, το ECOFIN και το Διοικητικό Συμβούλιο του Μηχανισμού Σταθερότητας. Κατά την άποψή μου, την οποία ανέλησα στο σύντομο, ελπίζω εύληπτο βιβλίο μου, που αυτή τη στιγμή, σε αυτόν τον καιρό κυκλοφορεί, αναλύω ότι και θα ήμουν ευγνώμων να ακούσω τις δικές σας αντιδράσεις, ε, των εμπειρογνωμόνων δηλαδή. Αναλύω λοιπόν ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να εντάξουμε αυτούς τους ενεχομένους ε, στην υπηρεσία και υπό ένα ισχυρό Υπουργό Οικονομικών της Ένωσης. Επίσης, άλλο πρόβλημα είναι η έλλειψη η αλληλεγγύης. Η παλιά βεβαιότης ότι η συνοχή της αποστολής και του μηνύματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξαφανιστεί. Νομίζω ότι υποθέτω ότι ισχύει ακόμα ότι όλα τα κράτη-μέλη ε, στερνίζονται το άρθρο 2 της συνθήκης για τις αρχές και τις αξίες μας, αλλά δεν είναι καθόλου προφανές ότι εστερνίζονται όλοι το άρθρο 3 που ορίζει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και η πραγματική ε, έννοια ε, του συμφώνου, του δημοσιονομικού συμφώνου, ιστορικά είναι η στιγμή που οι εταίροι της Βρετανίας ε, δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν πλέον, δεν είναι διατεθειμένοι να ανέχονται τις αντιρρήσεις που προέβαλε η Μεγάλη Βρετανία διαχρονικά και τώρα με μεγαλύτερη ισχύ από ό,τι στο παρελθόν για την ε, επίτευξη των στόχων της Ένωσης όπως ορίζονται στη συνθήκη. Και υπάρχει και ένα τρίτο μέγα πρόβλημα ότι δεν γίνεται μια δημόσια συζήτηση σχετικά. Βεβαίως εδώ το συζητούμε και είναι εξαιρετική η συζήτηση αλλά κοιτάξτε πόσοι συμμετέχουν ευρωβουλευτές. Πόσοι παρευρίσκονται καν. Τα εθνικά κοινοβούλια, κατά την άποψή μου, είναι απρόθυμα ή και ανίκανα να συνεννοηθούν με τα εθνικά πολιτικά κόμματα και να ε, διατηρήσουν την δημοκρατική και αποτελεσματική ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση για μια σειρά λόγους πρακτικούς. Ας πούμε, εκλογέ για τη Γερμανική Βουλή το 2013, ευρωεκλογέ το 2014. Ε, η ανάγκη να δημιουργηθεί μια νέα και αν μου επιτρέπετε να πω καλύτερη επιτροπή το 2014, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα συνταγματικά θέματα στην ουσία τους μέχρι την άνοιξη του 2015, των νωρίτερων. Στο μεταξύ, από τώρα και μέχρι την αρχή του 2015, έχουμε να κάνουμε πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολύ σημαντική, για να εδραιώσουμε τη Δημοσιονομική Ένωση. Και ε, θα σας παρακαλούσα επίσης να μου απαντήσετε για το πώς βλέπετε εσείς αυτή τη μετάβαση και αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα από το που βρισκόμαστε μέχρι που θέλουμε να πάμε. Πρόεδρε, σταματώ εδώ, αλλά μπορεί να ξαναζητήσω το λόγο αργότερα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, για να επανέλθω. Ευχαριστούμε. Για αλλαγή δεν θα μιλήσω αγγλικά, θα μιλήσω άλλη γλώσσα. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις, εξαιρετικές όλες ε, ε, στον τομέα τους. Είναι δύσκολη η κατάσταση και ε, τις αναλύεται πολύ ωραία. Ο Ζαν Βικτόρ Λουί ενέφερθηκε σε μια άναρχη κατάσταση, αν δεν απατώμε, με τις τόσο διαφορετικές διαδικασίες. Και όντω τούτη εδώ η κρίση, όσο καμία ε, στο παρελθόν, έδειξε πόσο εκρηκτική είναι για τη συνοχή την ίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η υπόθεση, δεν ξέρουμε αν έχει λυθεί το θέμα ή ε, αν ε, τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας, αλλά διαφαίνονται κάποιες μεγάλες και δύσκολες συγκρούσεις. Ο Άντρου Ντάφ υπερασπίζει το βιβλίο του «Διακυβέρνηση της Ευρώπης» Governing Europe. Για να δούμε τι θα κάνει η Μεγάλη Βρετανία όμως. Θα συνεχίσει να συμμετέχει. Θα ανέχεται να προχωρούν άλλοι παραπάνω ή ε, θα θελήσει να αποχωρήσει. Και έχω μια ερώτηση. Το είπε ο Γιάννης Αμανουηλίδης προηγουμένως. Με νέους τρόπους, νέες μορφές συμμετοχής, ιδιότητας μέλους. Η ιδέα λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν μια κοινότητα αλληλεγγύης να είναι. Και κανονικά θα πρέπει να αντιταχθούμε να υπάρξει επιλεκτική συμμετοχή. Να διαλέγει κάθε χώρα, α, εγώ αυτή την πολιτική δεν την κάνω, άλλη πολιτική όπου την πονάει την κάθε μια να μην συμμετέχει ή δεν της αρέσει. Α, τότε είναι Ευρώπη à la carte. Αυτό ανέκαθεν θέλαμε να το αποτρέψουμε εμείς. Εγώ θα έκανα μια διάκριση εδώ μεταξύ κρατών μελών που τώρα θέλουν να ε, τα βγάλουν πέρα ε, και να επανέλθουν τα οικονομικά. Αυτό είναι τα κράτη-μέλη και τα υποψήφια κράτη που μπορεί να είναι η Τουρκία ή η Ουκρανία που να είναι ε, συνδεδεμένες χώρες. Αλλά τα υφιστάμενα κράτη-μέλη δεν γίνεται να έχουν άλλη τη γιατί είναι και ένα θέμα ε, στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Δηλαδή, δημοσιονομικό σύμφωνο, οι μεν έχουν πολύ ωραία εσωτερική αγορά και οι άλλοι ε, που χειρίζονται τα θέματα ε, της ε, αλληλεγγύης και τα δημοσιονομικά. Βλέπω πόσα δισεκατομμύρια εκταμιεύουν οι χώρες ευρώ και οι άλλοι κάθονται απ' έξω με σταυρωμένα τα χέρια και λένε «Μπράβο παιδιά, ωραία δίνετε τα λεφτά». Κάπου έχει και όρια αυτή η κατάσταση. Έφυγε ο Ζαν Κλοντ Γνωρίζουμε ε, αυτό που ήθελε η Γαλλία, μια κρυφή επιθυμία μεικτού σώματος. Κογκρέντε Πέπλο, το έλεγε ο Ζισκάρ αυτό, ένα κογκρέσο των λαών. Η γαλλική γερουσία ανέκαθεν ναι, ήθελε να έχουμε ένα μεικτό κοινοβουλευτικό σώμα. Ε, Εμεί δεν το θεωρούμε σκόπιμο, ούτε καλή ιδέα εδώ, διότι όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και πρακτικά δεν θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Να πω μόνο ότι το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο σε αυτή την περίπτωση ζήτησε να αποφασίζει το σύνολο της ολομέλειας ε, ε, της Bundestag, όχι ένα όργανο ή υπόργανο. Δηλαδή, τρία μέλη του Bundestag που θα ερχόντουσαν σε ένα μεικτό σώμα δεν θα μπορούσαν να αποφασίσουν. Γιατί υπάρχει αυτή η απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου ότι αποφασίζει η ολομέλεια της Bundestag. Και είπε και ο Γιάννης Εμμανουηλίδης ότι ε, θα εξαρτηθεί από το πώς θα διαμορφωθεί η Δημοσιονομική Ένωση. Ωραία. Δηλαδή, θα έχουμε συντονισμό ακόμα εθνικών θεμάτων ή εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών και στο δημοσιονομικό δίκαιο σε κοινοτικό επίπεδο. Και εκεί είναι σαφές ποιος ασκεί το δημοκρατικό έλεγχο. Αυτό είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ονομάζεται. Ακρόαση είναι εδώ, δεν είναι διαπραγμάτευση. Ούτε πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις σήμερα. Ανάλογα με το πώς θα γίνει η χώριση αρμοδιοτήτων και εξουσιών θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν είναι σπουδαία πράγματα και μεγάλα, ετίθεται το ερώτημα ε, μήπως θα πρέπει να συμμετέχουν οι ευρωβουλευτές των εν χωρών και όχι των υπολείπων που δεν έχουν συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια. Και θα μπορούσα να φανταστώ την Ολομέλεια στο Στρασβούργο Δευτέρα Τετάρτη να συνεδριάζουν 27 και Πέμπτη να συνεδριάζουν οι 17 συν ευρωβουλευτές ε, από αυτές τις χώρες. Θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε και ιδέες προς την κατεύθυνση αυτή, αλλιώς τον βλέπω, τον κίνδυνο να έρχεται και τον ακούω. Γίνεται μια απόπειρα να φτιαχτεί ένα Ευρωκοινοβούλιο από εθνικούς βουλευτές ή μια μεικτή μορφή που, εν πάση περιπτώσει, και τα δύο για μένα δεν είναι αποτελεσματικά ούτε σκόπιμα. Ευχαριστώ, κύριος Μπρόνς. <coughs> Ε, σας ευχαριστώ. Ο καθηγητής Λουίς άρχισε λέγοντας, και ελπίζω να μην κατάλαβα καλά, ότι έχει γίνει εντυπωσιακή πρόοδος από την κρίση που δεν θα μπορούσε κανείς να την έχει σκεφτεί πριν την κρίση. Μάλλον αναφερόταν στις κινήσεις προς την ε, Δημοσιονομική Ένωση και την ε, προεποπτεία και τις διάφορες διασώσεις. Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτή η δήλωση και καθώς και κάποιες άλλες από άλλους ανθρώπους θα πρότειναν ότι η κρίση, η ύφεση όπως λέγεται δεν θα θεωρείται τόσο ως πρόβλημα όσο ως ευκαιρία και μια δικαιολογία για να προχωρήσει η διαδικασία της ολοκλήρωσης. Είναι σαν η ολοκλήρωση να είναι δικό τους θέμα στα οικονομικά, μάλλον να έχουν συμφέρον για τα οικονομικά προβλήματα και την φτώχεια και την ταλαιπωρία που προκαλούν. Ε, τώρα από οποιοδήποτε μπορούσε να δει από την αρχή τη Ευρωζώνης ότι θα ήταν πολύ απίθανο αυτή η εξωτερική αξία ε, ε, θα παρέμενε κατάλληλη για διάφορες διαφορετικές οικονομίες και φαίνεται ότι όποιο και αν είναι το κόστος αυτής της φτώχειας διευκολύνει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τώρα, για να προχωρήσω στον καθηγητή Ντεβίτ και εδώ νομίζω πως σωστά το έγραψε αυτό που είπε, ότι δηλαδή ο μηχανισμός σταθερότητας κατέστη δυνατός μέσω της αλλαγής της συνθήκης, της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ότι προηγήθηκε αυτής της αλλαγής. Δεν την ακολούθησε. Η ερώτηση που έχω εγώ είναι μάλλον απλή. Λειτουργούν αναδρομικά οι αλλαγές των συνθήκων. Εάν όχι, τότε κάποια σκιά πέφτει στην νομιμότητα του μηχανισμού σταθερότητας. Τώρα αν προχωρήσουμε στις διακυβερνητικές συμφωνίες που είναι ένας εφημισμός για μια ιδιωτική και άτυπη συμφωνία λέει λοιπόν ότι η συμφωνία αυτή μπορεί να, το ΔΕΚ μπορεί να ε, κρίνει τις διεθνείς αυτές διακυβερνητικές συμφωνίες. Αλλά εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, μόνο τα κρατημέλη και όχι οι κομισιόν μπορούν να παραπέμψουν ε, τέτοιες διακυβερνητικές συμφωνίες ε, στη ΟΔΕΚ. Μάλιστα, ο καθηγητής Πύρη που βέβαια τώρα έχει φύγει έλεγε ότι η Κομισιόν έχει να παίξει εδώ ρόλο και νομίζω είναι κάπως αμφίβολο ότι θα παίξει ρόλο η Κομισιόν αν δεν μπορεί να παραπέμψει τις ε, παραβιάσεις αυτών των συμφωνιών στο ΔΕΚ. Έπειτα είπε μια εναλλακτική λύση ότι ίσως ένα νέο μικρό σώμα θα μπορούσε να φέρνει τα θέματα αυτά στο 10 και πάλι χωρίς αλλαγές στη συνθήκη κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Αυτά έχω να πω για να είμαι σύντομος. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπρόντς. Πριν δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονές μας, να πάρει το λόγο ο συνάδελφος Μπρόκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ποτέ δεν άκουσα Βρετανό συνάδελφο να λέει ότι η Βουλή των Κοινοτήτων έλαβε ε, παράνομη απόφαση και το ESM το κύρωσε, το Μηχανισμό Σταθερότητας. Για να κάνουμε μια εξέταση εκεί μήπως παρανόμησε η Βουλή των Κοινοτήτων να το ψάξουμε. Λοιπόν, σοβαρεύομαι τώρα. Ε, δεν συμφωνώ απολύτως με τον συνάδελφο Λάινεν. Και για τις διαπραγματεύσεις που κάνουμε σήμερα στις 3 για το έγγραφο έχουμε μια θέση του Κοινοβουλίου που λέγει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διχοτομείται, δεν επιτρέπεται. Η Νομισματική Ένωση είναι μια πολιτική του συνόλου της κοινότητας και θα πρέπει να ασκείται με όρους κοινοτικής πολιτικής και με την κοινοτική μέθοδο. Υπάρχει μια διαφορά. Δύο χώρες έχουν opt-out, αλλά είναι κοινή πολιτική, δεν είναι διακυβερνητική η Νομισματική Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ, συνεπώς. Αυτή είναι η αφετηρία μας και αυτή είναι και η σημερινή κατάσταση. Ε, εμείς θεωρούμε ότι χωρίς αλλαγή της συνθήκης, με όλα τα μέτρα που λαμβάνονται τώρα και προτείνονται, τα θεσμικά όργανα και τα κοινοβούλια ε, έχουν το ρόλο τους, όπως αναγράφεται στη συνθήκη της Σαμβώνας και τα συντάγματά τους αλλά δεν μπορεί να αλλάξει ε, η χώριση των αρμοδιοτήτων. Και συνεχίζει αυτό. Και επειδή το ευρώ λοιπόν είναι κοινοτική υπόθεση, είναι αδιέρετες ε, και οι δομές και τα θεσμικά όργανα εκτός από την Ένωση. Και υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε, δεν μπορούν να υπάρχουν μικτές λύσεις. Δεν προβλέπονται στη σημερινή κείμενη νομοθεσία και οι μικτές λύσεις έχουν και προβλήματα νομιμοποίησης. Γιατί κάθε κοινοβούλιο εκλέγεται με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικό εκλογικό νόμο και με διαφορετική αναλογική μέθοδο. Δεν αναμειγνύονται αυτά γιατί θα έχουμε προβλήματα. Και κατά τα άλλα, πολιτικά κάτι τέτοιο θα ήταν άκρο επικίνδυνο. Και η κατάσταση που το ευρώ είναι ένα μέτρο ε, ε, πρωτοποριακό και θα συμμετάσχουν. 25-26 χώρες έχουν δηλώσει ότι το επιθυμούν και θα ήταν λάθος και πολιτικά να δημιουργηθούν τώρα νέα θεσμικά όργανα. Εγώ ως Γερμανός πολιτικός, για παράδειγμα, δεν μπορώ να δεχτώ να χτίσουμε ένα νέο τείχος απέναντι στο γείτονά μας την Πολωνία. Την Πολωνία που θέλει να μπει στο ευρώ όταν τη τα κριτήρια. Έτσι το λέω εμπαρόδο. Δεν μπορούμε να υψώνουμε νέα τείχη, νέα θεσμικά όργανα. Θα το θεωρούσα πάρα πολύ προβληματικό. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο δρόμος, ακόμα και αν έχει επιλεγεί διακυβερνητικά, γιατί μια χώρα μπλόκαρε την αλλαγή της συνθήκης, που λέγεται δημοσιονομικό σύμφωνο, δεν είναι η υπόθεση των 17, αλλά των 25. Αυτή είναι η πολιτική σωστή οδός και μέτρο προβλέπεται στο κείμενο της συνθήκης, στο σύμφωνο αυτό, ότι αυτό το διακυβερνητικό οικοδόμημα μετά από πέντε χρόνια θα ενσωματωθεί στη συνθήκη. Και ε, έτσι εκφράζεται και η κοινή βούληση των 25 για την κοινωνική μέθοδο, κοινοτική μέθοδο. Ότι σε πέντε χρόνια όλα αυτά θα ενσωματωθούν στη συνθήκη. Και αυτή είναι η σωστή και λογική αφετηρία για να εκκινήσουμε. Και κάτι άλλο. αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει ε, με ξεχωριστές δομές στη λήψη αποφάσεων και στην νομοθεσία, θα πρέπει οπωσδήποτε να χωριστεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, σε ένα θέμα να αποφασίζει με 17 επιτρόπους και σε άλλα θέματα με 27. Δηλαδή, έτσι το θεσμικό οικοδόμημα αναγνωρίζει ε, ιδιότητα μέλους διαφορετικής ποιότητας. Εγώ όμως δεν μπορώ να αναγνωρίσω. Ούτε το δέχομαι ότι έχουν διαφορετική ποιότητα ευρωβουλευτέ. Ακόμα και Βρετανοί. Δεν του αναγνωρίζω ότι είναι διαφορετικής ποιότητα. Ε, αυτή είναι η δύσκολη αφετηρία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ξαναπούμε το εξή. Κάθε κοινοβούλιο αποφασίζει για τι αρμοδιότητέ του. Και βάσει του άρθρου 9 του πρωτοκόλλου παριθμών 1 για στη συνθήκη που τώρα έχει μπει στο άρθρο 13 του Δημοσιονομικού Συμφώνου, θα πρέπει να βρούμε δυνατότητες διαβούλευσης βάσης συνένεσης μεταξύ των διαφόρων ε, επιτροπών των Εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή θα είναι η θέση που ε, θα υιοθετήσει και με την οποία μπαίνει σήμερα στις διαπραγματεύσεις στο Κοινοβούλιο. Τώρα, πώς θα λειτουργήσει το εσωτερικό του, ποια θα είναι η εργασία του Κοινοβουλίου και τελικά μπορεί να υπάρχουν σχηματισμοί που είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια και αυτορύθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν μπορώ να προεξοφλήσω ποια θα είναι αυτή. Αλλά μπορώ να προτείνω να το σκεφτούμε. Αλλά αυτό πώς εκφράζεται και ρητά μόνο στον τομέα του ελέγχου. Παράδειγμα, πρέπει να πούμε ότι αν η τραπεζική εποπτεία ε, έρθει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι για αυτή η εποπτεία δεν θα εγγράφεται στον τίτλο ανεξαρτησία που είναι η συνήθις τακτική της ΕΚΤ, αλλά ε, έχουν λόγο τα κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για θέματα δικαστηρίου, για θέματα ελεκτικού συνεδρίου, για θέματα διορισμών. Ε, η προστασία της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας δεν μπορεί σε αυτή την περίπτωση της εποπτείας να ισχύει ίσως εκεί να υπάρχει μια αντίστοιχη επιτροπή που να συνεργάζεται με τα εθνικά κοινοβούλια, να κάνουμε τις ακροάσεις για τους διορισμούς. Και αυτό είναι ένα θέμα αυτορύθμισης του Κοινοβουλίου και δεν σημαίνει ότι ε, υφίστανται διακριτική ε, μεταχείριση ή ε, υπονομεύονται κάποιοι βουλευτές. Αυτά τα θέματα με 17 και 27 δεν συμφωνώ. Ε, θα έχουμε δυσκολίες για την εφαρμογή τους και παρακαλώ να μας εξηγήσουν οι εμπορογνώμονες, να μας συμβουλέψουν. Γιατί όλο και περισσότερο ακούμε διάφορες φωνές ή ανισορροπίες να μην λυθούν ε, μέσω των ευρωμολόγων, αλλά μέσω νέου προϋπολογισμού στα πλαίσια από το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, από τους ιδίους πόρους και ο προπολογισμό αυτό να αφιερώνεται στι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει που είναι απαραίτητε στι χώρε και έτσι να αρθούν οι ανισορροπίε, όχι μέσω ομολόγων, έργων κτλ. Αν αυτό δεν βρίσκει εφαρμογή και για τα 27 κράτη-μέλη, τότε πώ λαμβάνεται η απόφαση για τον προπολογισμό. Πρέπει να ομολογήσω ότι απάντηση δεν έχω ακόμα, αλλά είναι ε, κομβικό αυτό το θέμα που καλούμαστε να απαντήσουμε και θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω ε, ποια νομική δομή μπορεί να εφευρεθεί εκεί έτσι ώστε ε, αυτό το ζήτημα να μπορεί να λυθεί με βάση τις συνθήκες και να μην έχουμε ένα νέο παράλληλο διακυβερνητικό προϋπολογισμό που να εκφεύγει του ε, κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σα ευχαριστώ. Εγώ θα σα προτείνω να αλλάξουμε τα ωράρια για τις εργασίες μα με, τον εξή τρόπο, ώστε να μπορέσουν τώρα να απαντήσουν οι καθηγητέ που παρενέβησαν σήμερα το πρωί. Δεν μπορώ να δώσω περισσότερο παρά 5 λεπτά έκαστος, ε, ε, ώστε να μπορέσουν να παρέμβουν και οι άλλοι δύο εμπειρογνώμονε που έχουν προβλεφθεί για σήμερα το πρωί και το απόγευμα να ακούσουμε αμέσω του άλλου τρει καθηγητέ που ήδη προβλέπονται και η συζήτηση με τους συναδέλφους να γίνει για τις πέντε εκθέσεις αμέσως μετά από τούτη την πρώτη φάση του, στο απόγευμα. Παρακαλώ λοιπόν να πάρετε το λόγο να απαντήσετε στις προτάσεις και τα ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί μέχρι τώρα. Ποιος θέλει να πάρει πρώτος. Ο Λουίς. Ο κύριος Λουίς. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν έχει νόημα να δώσουμε απαντήσεις, αν ο στόχος ήταν να δοθούν απαντήσεις. Τουλάχιστον εγώ είχα σκεφτεί να θέσω εγώ ερωτήσεις ε, και να περιμένω κάποιες απαντήσεις. Διαπιστώνω πάντως ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο την τελευταία διετία σε θέματα οικονομικής διακυβέρνησης. Και αυτή ήταν μία διαπίστωση. Δεν είναι ότι ε, αξιοποιήσαμε την κρίση, αλλά προσπαθήσαμε με ό,τι μέσα είχαμε να την αντιμετωπίσουμε μερικές φορές και με αυτοσχεδιασμούς. Για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το είχε προτείνει το 2002, απέσυρε την πρόταση το 2004, χρειάστηκε να περιμένουμε μέχρι το 2010 για να επαναπροσανατολιστούμε προς αυτή τη μέθοδο, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που χρήζει φυσικά κάποιες βελτίωσεις από άποψη ασφάλειας δικαίου και ίσως και εκδημοκρατισμού της όλης διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τώρα, πιο γενικά, σε ό,τι αφορά την ανάγκη να λάβουμε υπόψη την ανάγκη ολοκλήρωσης σε επίπεδο 27 χωρών και ε, να λάβουμε υπόψη ότι η Ευρωζώνη θα πρέπει να σεβαστεί την ακαιρεότητα ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 27. Αυτό είναι διαφυσβήτητο, αλλά αυτό που με εκπλήσει είναι αυτό που είπε ο κύριος Μπρόκ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η ΟΝΕ είναι ένα κοινό σχέδιο. Τώρα διαπιστώνουμε ότι αυτοί που θέλουν περισσότερη ολοκλήρωση σε νομισματικά θέματα το κάνουν φυσικά ανάλογα με τις ανάγκες αυτής της ολοκλήρωσης ε, και ζητούν και περισσότερη μάλλον οικονομική ε, ολοκλήρωση είναι αυτοί που καταφεύγουν σε έκτακτους μηχανισμούς και μάλιστα το, η συνθήκη της Λισαβόνας ε, ενθαρρύνει αυτή την τάση γιατί το άρθρο 136 προβλέπει τη δυνατότητα λήψης εκτάκτων μέτρων, αλλά η εξαίρεση δεν είναι μόνο οικονομική ή νομισματική ένωση, είναι οικονομική και νομισματική ένωση. Και τώρα ε, έχουμε μερικέ χώρε που για πολιτικού λόγου θα μπορούσαν να ενταχθούν στην Ευρωζώνη, αλλά για πολιτικού λόγου δεν θέλουν. Αλλά και ακόμη και χώρε που έχουν αυτοεξαίρεση. Όταν είχαμε τη, τη συνθήκη του Μάστρικ, δεν φανταζόμασταν ότι με την αυτοεξαίρεση θα έβγαιναν άπαξ και διαπαντό εκτό ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, ε, θεωρούσαμε ότι κάποια στιγμή θα έμπαιναν και χώρες αυτές στην ΟΝΕ, γιατί είχαν συμβάλει στην εκπόνηση της συνθήκης του Μάστριχτ και του Νομισματικού Ινστιτούτου και στην διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ναι, λοιπόν, θα πρέπει να τηρήσουμε τις αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εσωτερική αγορά και τα βήματα προς μια Οικονομική και Νομισματική Ένωση ουσιαστικά αποτελούν τη φυσική συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν στα πλαίσια της συνθήκης του Μάστριχτ. Ευχαριστώ. Τώρα ο καθηγητής ο κ. Εμμανουηλίδης. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε τρία θέματα. Δεν θεωρώ ότι μπορώ να δώσω απαντήσεις βέβαια. Δύο θέματα που ανέφερε ο κύριος Λάινεν και με ρώτησε προσωπικά το νέο είδος ιδιότητας μέλους. New forms of belonging, το είπα στα αγγλικά. Νέοι τρόποι του ανήκειν σε μια κοινότητα. Θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στα κράτη-μέλη ε, που είναι μέλη της Ένωσης και κάποια άλλη ε, κράτη που είναι εκτός και επιδιώκουν τη σύνδεσή τους, είναι υποψήφια κτλ. Αυτή η συζήτηση δεν είναι καινούρια, την έχουμε κάνει εδώ και καιρό. Ε, στα έγγραφα που είχαμε για σήμερα αναφερόταν αυτό, γι' αυτό και εγώ ε, στάθηκα λίγο. Αλλά το θέμα ε, και το ερώτημα τι κάνουμε με χώρες που είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και τι κάνουμε κυρίως με το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχετε δίκιο. Θα πρέπει να αντισταθούμε στην επιλεκτική συμμετοχή σε πολιτικές, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Δηλαδή, να αναρωτηθούμε τι θα κάνουμε σε περίπτωση που φτάσουμε μέχρι ε, εκεί και τι θεθεί το ερώτημα τι κάνεις με μια χώρα που δεν είναι διατεθειμένη να ακολουθήσει κάποιους δρόμους αλλά ταυτόχρονα χρειάζεσαι τη συμφωνία του για να προχωρήσεις αυτού του κράτους μέλους. Τα λέω τόσο ασαφώς γιατί δεν ξέρουμε περί τίνος συζητούμε περισσότερη δημοσιονομική και οικονομική ενοποίηση και ολοκλήρωση χωρίς να ξέρουμε στις λεπτομέρειες τι σημαίνει. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί δεν ξέρουμε τα επόμενα χρόνια, ένα, δύο, τρία χρόνια, τι πίεση θα ασκήσει η κρίση σε μας. Και η εμπειρία μας λέει ότι η πίεση της κρίσης ήταν εκείνη που όθησε τα κράτη-μέλη σε επίπεδο 17-27 να κάνουν ή να μην κάνουν ορισμένα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από το πώς εμφανίζεται η κατάσταση, θα έρθει μια στιγμή ε, που θα τεθεί το ερώτημα. Και θα πρέπει να απαντήσουμε και μπορεί να έχει έρθει τώρα, ήδη. Τι κάνεις με μια χώρα η οποία έχει πρόβλημα με μια περαιτέρω διεύρυνση. Γι' αυτό ε, μίλησα εγώ για περιορισμένη ιδιότητα μέλους ή συνδεδεμένο μέλος. Limited ή member ότι δεν είναι βέβαια εναλλακτική. Μπορούμε να το συζητήσουμε και να πούμε ότι αποκλείεται ως εναλλακτική λύση ή να πούμε μπορούμε πάρα πολύ περιορισμένα να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά τη συζήτηση να την κάνουμε. Για τις λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζουμε επίσης και το θέμα της θεσμικής σύνδεσης των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα πρέπει να καταλάβουμε μεγαλύτερη σαφήνεια, να όταν μιλάμε για περισσότερη διαφοροποίηση και συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, θα πρέπει να ξέρουμε τι εννοούμε. Δεν έχουμε ακόμα τις απαντήσεις. Κρίμα που έφυγε ο κύριος Πύρης. Εγώ έχω την εντύπωση ότι συχνά στη συζήτηση αρχίζουμε από το τέλος. Δηλαδή, πρώτα αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε τα εθνικά κοινοβούλια και μετά κάνουμε την ερώτηση για ποιο σκοπό. Άρα ο στόχος περισσότερο είναι να συμμετέχουν τα εθνικά κοινοβούλια και όχι οι λύσεις που πρέπει να ε, βρεθούν με τα υφιστάμενα εργαλεία ή όσα πρέπει να δημιουργηθούν. Έρχομαι ξανά στα αγγλικά, πάρα πολύ σύντομα, το θέμα που έθιξε ο κύριος Δαφ. Με έχει προβληματίσει πολύ και απάντηση δεν έχω το θέμα της δημόσιας συζήτησης για την παράθεση. Δεν γίνεται τέτοια συζήτηση. Τούτη δε η ακρόαση είναι εξαίρεση. Ευτυχώς, και αυτό το είδαμε τα δύο-τρία τελευταία χρόνια σε κάποια κράτη-μέλη, έχει αρχίσει και γίνεται αυτή η συζήτηση. Σε μία από τις δύο χώρες που γνωρίζω καλύτερα, στη Γερμανία, γίνεται η συζήτηση. Τι σημαίνει το να θες να έχεις περισσότερη Ευρώπη και τι μπορεί αυτό να σημαίνει. Έχει αρχίσει αυτή η συζήτηση. Και νομίζω είναι και ευκαιρία. Γιατί σε άλλα κράτη-μέλη μπορεί να μην γίνεται η συζήτηση για το τι σημαίνει περισσότερη Ευρώπη εντό εισαγωγικών, που είναι πάρα πολύ ασαφή όρο γενικά, αλλά τουλάχιστον βλέπει τι ειδήσει στην τηλεόραση, διαβάζει τα άρθρα και είναι θέμα που πρωταγωνιστεί. Με πολύ διαφορετικού όρου γίνεται η συζήτηση, όπω πολλοί από εμά όταν συζητούμε με τον κόσμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την αίσθηση ότι είναι σαν να ζω σε άλλο πλανήτη βλέπουν το ίδιο θέμα από τελείω διαφορετική προοπτική και το θέμα είναι πώς θα έρθουν αυτοί σε συζήτηση. Χρειάζεται να εξευρωπαϊστεί η εθνική συζήτηση και να γίνει διεθνής. Αυτό δεν είναι καινούριο. Εχθέ, Μάλλον αυτό είναι μια συζήτηση που κάνουμε εδώ και χρόνια και δεκαετίες, αλλά τούτη εδώ η κρίση πραγματικά είναι ευκαιρία που δεν είχαμε στο παρελθόν. Το γιατί το θέμα δεν είναι τώρα να δημιουργηθεί ε, κάτι, ένα ωραίο φυλάδιο πολυτελές και γυαλιστερό κενό περιεχομένου. Το θέμα είναι να συζητήσουμε τα πραγματικά θέματα. Είναι επικίνδυνο, επικίνδυνο είναι βεβαίως και ρηψοκίνδυνο είναι. Γιατί είναι μεγάλες οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κρατών μελών, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε τώρα αμέσως να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Και μάλιστα έμεσα και όχι ευθέως, όχι άμεσα. Ε, ε, ε, συγγνώμη, άμεσα και όχι έμεσα. Και για το 2015 που είπατε δεν ξέρω. Νομίζω οι ευρωεκλογέ είναι πραγματικά ε, κομβική συγκυρία και θα πρέπει να δούμε αν χρειαζόμαστε ομάδα προβληματισμού, ομάδα περισυλλογή, ίσως και με μεγαλύτερη καινοτομία να σκεφτούμε τίποτα καινούριο. αλλά εγώ τη μαγική λύση δεν την έχω. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση για αυτή την πρώτη φάση. Ο καθηγητής Ντεβίτε. Παρακαλώ. Θα απαντήσω σε τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις που έγιναν προς εμένα. Δύο από τον Ρομπέρτο Γουαλτιέρη. Καταρχήν, με ρώτησε αν υπάρχει αντίφαση του Δημοσιονομικού Συμφώνου με την κοινοτική νομοθεσία, δεδομένου ότι προβλέπει κάποιες δημοσιονομικέ κυρώσει που αναφέρονται στο άρθρο 260 τη Συνθήκη Λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια διαδικασία δηλαδή με βάση την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το ΔΕΚ να επιβάλλει κυρώσει για τη μη τήρηση του κοινοτικού δικαίου, για, για τίποτα άλλο όμω. Και αν δούμε τη διατύπωση, το άρθρο 8.2 του Δημοσιονομικού Συμφώνου δεν παραπέμπει σε εφαρμογή το άρθρο 260 της συνθήκη Λειτουργίας Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάει για ένα ξεχωριστό σύστημα οικονομικών κυρώσεων στα πλαίσια του δημοσιονομικού κριτηρίου. Το θέμα είναι πώς θα υπολογίσουμε το ύψος των κυρώσεων ή πώς θα υπολογίσουμε το ποσό που ζητούν τα κράτη-μέλη. Αυτό θα γίνεται σε αντιστοιχεία με αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του άρθρου 260. Δηλαδή, η μνήα της ε, συνθήκης, ε, της, ε, του άρθρου της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάπως ατυχής. Γιατί δεν λέει ποιο σύστημα θα εφαρμοστεί, αλλά παραπέμπει σε ένα μοντέλο αντίστοιχο με αυτό που θα χρησιμοποιήσει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Δεν υπάρχει νομικό κόλλημα, ούτε αντίφαση. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι είναι αναποτελεσματικό ο μηχανισμός. Γιατί αν δούμε τι πραγματεύονται οι δημοσιονομικές κυρώσεις, βλέπουμε ότι ισχύουν σε περίπτωση αποτυχίας ε, των χωρών του δημοσιονομικού συμφώνου να ε, εισαγάγουν ε, τον χρυσό κανόνα στην εθνική τους ένωμη τάξη. Βέβαια, όταν λέμε εθνική ένωμη τάξη δεν εννοούμε σαν και καλά το Σύνταγμα. Οπότε μπορεί οποιοδήποτε χώρα το κάνει, άσχετα με το Σύνταγμα, και πληρεί αυτή την υποχρέωση. Βέβαια, ένας μη ισορροπημένος ε, ε, προϋπολογισμός που δεν τηρεί τις εθνικές διατάξεις δεν υπάγεται στις κυρώσεις του, ΕΚ, του ΔΕΚ. Οπότε συμφωνώ ότι δεν είναι και πολύ αποτελεσματικό το δημοσιονομικό σύμφωνο. Δεν ήταν και πολύ καλή ιδέα ούτως ή άλλως από την αρχή. Τώρα, για τη δεύτερη σας ερώτηση, κύριε Γουαλτιέρη. Ρωτήσατε αν μπορεί το δημοσιονομικό σύμφωνο να βάζει τον ισορροπημένο προπολογισμό στο 0,5 με 1% αν είναι πιο φιλόδοξο από την κοινοτική νομοθεσία ή είναι αντιφατικό με αυτήν. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα αυτός ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός. Από νομική άποψη πιστεύω ότι είναι πιο φιλόδοξο από τη συνθήκη, γιατί η συνθήκη λέει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν δημοσιονομικό έλλειμμα το πολύ 3%. Οπότε μπορούν από μόνο τους να αποφασίσουν ένα χαμηλότερο έλλειμμα και μπορούν κάτι τέτοιο να το κάνουν και στο δημοσιονομικό σύμφωνο. Από νομική άποψη είναι πιο φιλόδοξο, αλλά δεν είναι αντιφατικό νομικά. Από πολιτική άποψη και οικονομική άποψη πιστεύω ότι έχει πάρει λίγο στραβό δρόμο το δημοσιονομικό σύμφωνο. Μία ερώτηση μου έθεσε και ο κύριος Μπρόγκς. Τι σημαίνει το ότι ο μηχανισμός σταθερότητας έχει ήδη τεθεί σε ισχύ ενώ η έγκριση για κάτι τέτοιο μέσω τροπολογία ε, τη συνθήκη λειτουργία ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τεθεί σε ισχύ, αλλά θα τεθεί την 1η Πρώτου Ιανουαρίου. Είπατε, ε, θα ισχύσει αναδρομικά η αλλαγή τη συνθήκη. Όχι. Η απάντηση είναι κατηγορηματική όχι, γιατί οι αλλαγέ τη συνθήκε δεν μπορούν να ισχύσουν αναδρομικά. Μπορούν να ισχύσουν μόνο για το μέλλον. Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά την, τι συμβαίνει. Η ρήτρα απο, απαγόρευσης διάσωσης ε, προβλέπει τη δυνατότητα χρηματοοικονομικής υποστήριξης μιας χώρας προς άλλες. Η no bailout clause δεν απαγορεύει τη δημιουργία ενός μηχανισμού που στο μέλλον μπορεί να παράσχει ε, οικονομική στήριξη σε κάποια κράτη-μέλη. Κατά τη γνώμη μου αυτό συνέβη. Δηλαδή θεσπίστηκε ένα σύστημα μέσω της συνθήκης για το μηχανισμό σταθερότητας. Τα όργανα, το όργανο αυτό, ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί από την περασμένη εβδομάδα, οπότε μπορεί να ξεκινήσει να ε, λειτουργεί, αλλά δεν μπορεί να ξεκινήσει τη χορήγηση οικονομικής ε, ενίσχυσης πριν την 1η Ιανουαρίου, δηλαδή πριν την τροποποίηση της συνθήκης για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει δηλαδή νομική αντίφαση στο μέτρο που το Διοικητικό Συμβούλιο τη συνθήκη του Μηχανισμού Σταθερότητα δεν έχει λάβει απόφαση για την οικονομική στήριξη μια χώρα. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο μετά την πρώτη πρώτου από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ και η σχετική αλλαγή τη συνθήκη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά την, το σχέδιο Μπύρης, οι πιο μετριοπαθή πρόταση που μας έκανε σήμερα ο Ζανκλοντ Πυρίς, που αναμειγνύει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από νομική άποψη είναι προβληματική. Γιατί η ιδέα μια ισχυρότερη οικονομική και νομισματική ένωση θα σήμαινε κατά ανάγκη εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Δεν σημαίνει ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χωρί όμω αναθεώρηση των συνθηκών κάτι τέτοιο θα ήταν παράνομο κατά όλους η πιο μετριοπαθής ε, λύση του κυρίου Πυρής είναι πολύ πιο νομικός αμφίβολη από τη πιο ριζοσπαστική του λύση κάτι ε, ε, νέο εκτός του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από πολιτική άποψη όμως είναι απαράδεκτο, ενώ από νομική είναι πιο νόμιμο. Αυτά ως προς τις ε, προτινόμενες λύσεις του κυρίου Ζαν-Κλοντ Πυρής. Ευχαριστώ. Έτσι κλείνουμε την πρώτη σύνοδο εδώ και ξεκινάμε αμέσω στη δεύτερη που έχει ως θέμα τα ευρωπαϊκά και εθνικά θεσμικά όργανα στο πλαίσιο της πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Ένα θέμα το οποίο έχει βέβαια ήδη ε, αναφερθεί αλλά χρειάζεται βάθυνση. Καταρχήν για ένα τέταρτο θα ακούσουμε τον καθηγητή Ρενό Ντεούς που είναι καθηγητής ε, του κέντρου Ζαν Μονέ ε, στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών όπου διευθύνει το μάστερ ευρωπαϊκών και διατλαντικών υποθέσεων. Οι εργασίες του έχουν ανέκαθεν επικεντρωθεί στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στα πολιτικά συστήματα. Νομίζω πως έχει ήδη έρθει εδώ στην Προεδρία και μπορεί να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επειδή ο χρόνος είναι λίγος και είναι και χρήμα σήμερα, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για το κατά πόσο είναι σκόπιμη η κοινοτική μέθοδος ε, μάλλον το, τώρα. Να σα πω ποιο είναι ο ορισμό της κοινοτική μεθόδου. Είναι ένα γνωστό ορισμό εδώ και γι' αυτό θα μπω αμέσω στην ουσία των επιχειρημάτων μου, που είναι ε, η εξής. Καταρχήν, Γνωρίζουμε βασικά πόσο σημαντικό, ε, σημαντική είναι η κοινοτική μέθοδος, το θύμισε μόλις και ο κύριος Μπρόκο, για την οικοδόμηση της Ευρώπης. Αυτό που θεωρώ πως είναι σημαντικό όμως να, να τονίσουμε είναι όχι το, η προσωπική κρίση, αλλά είναι το θέμα της πολιτικής ε, και λειτουργικής αξιολόγησης. Το γεγονός ότι έχει αποδείξει ότι είναι μια, ένα σχετικά σταθερό μοντέλο από την αρχή της οικοδόμησης της Ευρώπης, σταθερή με την έννοια ότι έχει μπορέσει να ανταποκριθεί σε διάφορες πολύ ουσιαστικές αλλαγές, όπως ε, για παράδειγμα την ανάδυση ενός ισχυρού κοινοβουλευτικού σώματος που δεν είχε προβλεφθεί εξ αρχής. Επίσης, μπόρεσε να ενσωματώσει, πολύ, να, να ενσωματώσει σωστά τον αριθμό των χωρών που συμμετέχουν. Πολύ μεγάλη αύξηση χωρών που συμμετέχουν στην Ένωση. Και εδώ και πάλι θα θυμάστε ότι υπήρχαν πολύ μεγάλοι φόβοι ότι μπορεί να αντιμετωπίζαμε την κατάρρευση ολόκληρου του συστήματος λόγω της ε, μεγάλης αύξησης του μεγέθους της Ένωσης. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη όπως είδαμε. Επίσης γνωρίζουμε παρόλα όσα ε, λέω ότι τα τελευταία 20 χρόνια υπήρξε ένα πρότυπο αλλά ταυτόχρονα αποτέλεσε και ένα αντικείμενο επικρίσεων, γιατί είχε να αντιμετωπίσει πολλές επικρίσεις από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ε, όχι μόνο όταν ε, θα έχετε διαπιστώσει στο Ευρωβαρόμετρο, αλλά και στις τελευταίες εθνικές εκλογές ότι ε, δέχεται επικρίσεις. Πρέπει να το δεχτούμε, να, να, να θυμηθούμε ότι είναι πρότυπο αλλά και σημείο πίεσης, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές απόπειρες να εφευρεθεί Κάτι ακόμα. Προσπάθειες οι οποίες δείχνουν αυξανόμενη απροθυμία από πλευρά των χωρών μελών να αφιερώσουν περαιτέρω, να, μάλλον να προσδώσουν περισσότερο αρμοδιότητα στην Ένωση. Και έτσι καταλήξαμε στο να έχουμε τη δομή πυλώνων στη συνθήκη του Μαστρίχτ. Έτσι εφευρέθη αυτό αυτό το μπαρόκικο δόμημα που είναι γνωστό ως ανοιχτό η μέθοδος ε, συνεργασίας, μέθοδος μάλλον ανοιχτής συνεργασίας και ε, έτσι έχουμε φτάσει στη σημερινή ένωση. Όπως τη γνωρίζουμε και αν κανείς τη μελετήσει θα διαπιστώσει πως πολλά ε, στοιχεία οφείλονται σε αυτή την απροθυμία να γίνει δεκτή η ευρωπαϊκή πειθαρχία και να δοθούν αρμοδιότητες στο κέντρο. Το θυμίζω γιατί νομίζω πως έχει σημαντικές επιπτώσεις για το μέλλον της, Ευρωπαϊκής, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Τούτου λεχθέντος, αυτό που μπορούμε νομίζω να διαπιστώσουμε από τις ευρωπαϊκές ε, αντιδράσεις στην οικονομική και νομισματική κρίση είναι ότι είτε μας αρέσει είτε όχι και δεν, είναι δεν ισχύει το ίδιο σε όλες τις πρωτεύουσε. η κοινοτική μέθοδος τυχαίνει να λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ως ένα ε, λειτουργικό σύστημα εξορισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει ότι παρότι έχουν γίνει διάφορες απόπειρες να εφευρεθούν εναλλακτικέ, δεν έχει ακόμα βρεθεί μια έγκυρη και λειτουργούσα ε, μέθοδος για την Ένωση. Τα στοιχεία στα οποία, τα οποία ανέφερα πριν από λίγο ε, απέδειξαν ότι δεν μπορέσαμε να φτάσουμε σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Και μάλιστα θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή για τη λειτουργία της ε, ε, ΟΝΕ οφείλονται την απροθυμία να δεχθούμε μεγαλύτερο βαθμό ευρωπαϊκής πειθαρχίας από εξ αρχής. Υπάρχουν βέβαια και εξωτερικοί παράγοντες, αλλά αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι εάν είχαμε δεχτεί έναν βαθμό ευρωπαϊκού ελέγχου και την πειθαρχία που, είναι, που εξυπακούεται, δεν θα βρισκόμασταν τώρα σε αυτή τη φάση. και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε παρά τη χλιαρή αντιμετώπιση της, αντιμε... της ανάθεσης και της ε, παραχώρησης αρμοδιοτήτων, τα κράτη-μέλη έχουν δεχθεί προωθηθεί σταδιακή κοινοτικοποίηση των όσων είναι πιο προσφυλή στην εθνική κυριαρχία όπως ε, ιστορικές υποθέσεις και δικαιοσύνη και όταν αντιμετώπισαν δύσκολες επιλογές σε σχέση με την κρίση χρέους οι απαντήσεις του ήταν ε, κλασικά κοκκινοτική μέθοδος, δηλαδή να δώσουν περισσότερες αρμοδιότητες, να χωρίσουν περισσότερες αρμοδιότητες στο κέντρο, στην Κομισιόν και στο δικαστήριο, το ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αξιοσημείωτο το ότι αυτό συνέβη παρά τους πολύ ισχυρούς αντίθετους πολιτικούς ανέμους. Τώρα, ποια είναι τα διδάγματα που θα έπρεπε κανείς να αποκομίσει από αυτό για το μέλλον της Οικονομικής και της Νομισματικής Ένωσης. Θα ξεκινήσω με δύο ε, προϋποθέσεις που κατά την ουσία εξηγούν τα υπόλοιπα που θα πω. Καταρχήν, αυτό για το οποίο συζητάμε σήμερα όσον αφορά τη μελλοντική δομή της ε, ΟΝΕ, βασικά είναι ένα μόνιμο πρόβλημα Οποτεδήποτε εξετάζουμε περαιτέρω ολοκλήρωση. Πόση εκχώρηση εξουσίας προς το κέντρο. Ποιο βαθμό πειθαρχία είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε. Και αυτό σημαίνει ότι η δική μας, ε, τουλάχιστον η δική μου άποψη είναι, και συμμερίζομαι τόσο από ο κύριο Μπροκ, να έχουμε υπόψη μας ότι η κοινοτική μέθοδος είναι κάτι πολύτιμο. Όχι οποιοδήποτε είδος πολιτικού, πολιτικής σκέψης, αλλά ως λειτουργική ε, σκέψη για το, όπως λένε και άλλοι, ε, σε άλλα πλαίσια, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση κατά τη γνώμη μου. Ένας από τους κινδύνους, και αυτό ήταν προφανές σήμερα το πρωί κατά τη συζήτηση, ε, είναι η υπερβολική διάλυση Δηλαδή, για να έχουμε στο πλευρό μας κυβερνήσεις που δεν δέχονται ένα συγκεκριμένο βαθμό πειθαρχία και εκχώρησης αρμοδιοτήτων, θα έτεινε κανείς να δεχτεί μια περιορισμένη πειθαρχία και όχι το επίπεδο που είναι απαραίτητο. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι, ε, θα ήταν λάθος, αλλά βέβαια και αναγνωρίζω ότι είναι πολιτική κρίση αυτή που εκφέρω τώρα. Επίσης σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι το θέμα της θεσμικής ε, σαφήνειας. Νωρίτερα αναφέρθηκα στο γεγονός ότι η κοινή γνώμη είναι μετριοπαθής κατά τη γνώμη μας, αλλά και κάπως τα έχει χάσει με τα όσα συμβαίνουν. Και ανησυχεί για τις εξελίξεις ε, σε σχέση με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στις χώρες μας. Θα ήταν λοιπόν πολύ σημαντικό όποια μεταρρύθμιση και να αποφασιστεί να γίνει απο... Ε, κατανοητή ξεκάθαρα και η χιονοστιβάδα μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει μέχρι στιγμή, οδήγησε, όπως είπαν και πολλοί ομιλητές, σε μια κατάσταση όπου όλο ένα και πιο δύσκολο είναι να κατανοήσει κανείς ποιος, ποιος ε, είναι ο επικεφαλής και, και Ποιο είναι αρμόδιο για αυτά που αποφασίζονται ή που δεν αποφασίζονται. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θεσμικό ζήτημα, ότι δηλαδή θα πρέπει να δομηθεί η σκέψη μας για αυτά τα θέματα. Έτσι λοιπόν έρχομαι σε κάποια πιο προσγειωμένα θέματα. Πώς μπορούμε εμείς να μεταρρυθμίσουμε την ΟΝΕ, διατηρώντας, μάλλον, έχοντας μάλλον όλα αυτά υπόψη, χωρίς δηλαδή να φτιάξουμε θεσμούς που μπορεί να δυσκεράνουν τη λειτουργία της Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα να ε, έχουμε και έναν επαρκή βαθμό σαφήνειας, θεσμικής σαφήνειας. Η προφανής απάντηση, η αρχή, θα ήταν να πούμε ότι ότι οι θεσμοί κοστίζουν χρήματα. Ας αποφύγουμε να δημιουργούμε νέους θεσμούς και νέους μηχανισμούς που μπορεί να επικαλύπτουν αυτά που ήδη υπάρχουν και να καταστήσουν όλα αυτά ακόμη πιο δυσνόητα για τους πολίτες. Και ας επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε μια εργαλειοθήκη πώς μπορούν τα υφιστάμενα θεσμικά όργανα να μπουν μέσα στη κυβέρνηση της μεταρρυθμισμένης ΟΝΕ. Όπως ακούσαμε το, σήμερα το πρωί, το πρόβλημα διαφέρει από τον ένα στον άλλο θεσμό. Μπορούμε ήδη να πούμε πως δεν φαίνεται να είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα σε σχέση, για παράδειγμα, με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γιατί έχει πολύ σημαντικό σε ελεγκτικές δραστηριότητες, περιορισμένες μεν, αλλά πολύ σημαντικές ε, μέσα στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο και δεν υπήρξε κανένα παράπονο για το γεγονός ότι ένας Βρετανός δικαστής θα μπορούσε να ε, δικάσει σε ένα δικαστήριο και μπορεί να έχει γνώμη να εκφέρει για την εφαρμογή του, του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Η Κομισιόν είναι πιο δύσκολο σώμα, γιατί δεν είναι πολιτικό. όργανο. Δεν είναι τόσο αντιπροσωπευτικό όργανο όσο είναι το κοινοβούλιο βεβαίως. Βεβαίως η συμμετοχή των χωρών της κάθε χώρας μέλους θεωρείται ως ένα σημαντικό και κεκτημένο. Αλλά ταυτόχρονα η ιδέα ότι η Κομισιόν θα μειωθεί, θα έχει λιγότερα μέλη από ό,τι τα μέλη της Ένωσης, είναι κάτι το οποίο φαίνεται να είναι δεκτό, να αποδεκτό από διάφορες ε, πρωτεύουσες. Αν σκεφτούμε την τελευταία έκθεση Βέστε Βέλε, Μα δεν είναι με αυτόν τον τρόπο φτιαγμένη αυτή τη στιγμή η Επιτροπή. Αυτό το χρησιμοποιώ ως πολιτική απόδειξη για να πω ότι η Κομισιόν δεν θεωρείται από όλους ως, ως αντιπροσωπευτικό σώμα και θα προχωρήσω λίγο περισσότερο. Και δεν ε, πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις συνθήκες μια επιτροπή πρέσβεων ε, που απλά θα ενημερώνει για τα συμφέροντα των χωρών τους. Αντιθέτως, οι επίτροποι δεν πρέπει να το κάνουν αυτό. Αφού λοιπόν όταν αποφασίζουμε τι και πρέπει να κάνουμε για την Κομισιό, να έχουμε στο μυαλό μας αυτή την αποστολή και ας δεχτούμε το γεγονός ότι μέσα στο Κομισιόν μπορεί να έχουμε εκπροσώπους χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης. Αυτό δεν είναι πρόβλημα είναι μάλλον ε, θέμα καλής πολιτικής. Το να πούμε δηλαδή ότι αναθέτουμε ευθύνε για την οικονομία και την Νομισματική Ένωση σε ένα μέλος της Επιτροπής που τυχαία είναι ε, και πολίτης της ε, Ευρωζώνης είναι, πολιτική, είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Τώρα έχουν υπάρξει έντονε εκκλήσει όπω αναμενόταν σήμερα το πρωί. υπέρ της συμμετοχής του Κοινοβουλίου στη μελλοντική λειτουργία της ΟΝΕ. Και αυτή δεν είναι νέα άποψη. Στη θυμάμαι ότι έχω ακούσει την ίδια έκκληση πριν από 15 χρόνια και παραπάνω στην διακυβερνητική διάσκεψη του Άμστερνταμ. Έχω ωστόσο αμφιβολίε γι' αυτό που δεν είναι βάσιμε νομικά, αλλά βασίζονται στα αυτά που βλέπω για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτό αυτό το σώμα, αλλά και η Ένωση ευρύτερα στις χώρες μας. Ναι, η συνθήκη αναφέρεται στους πολίτες ε, της Ένωσης γενικά. Και μπορεί, μπορεί κανείς να πει ότι οποιοδήποτε πολίτης ε, ε, ήταν το νόημα αυτής της συνθήκης, αλλά δεν ε, γίνεται αντιληπτό έτσι το κοινοβούλιο στις χώρες μας. Ξέρουν βέβαια ότι το κοινοβούλιο εκλέγεται σε κάθε μια σε κάθε μια από τις χώρες μας αλλά είτε μας αρέσει είτε όχι, θεωρούν τους ευρωβουλευτές ως εκπροσώπους μιας συγκεκριμένης ε, επικράτειας. Εγώ πιστεύω πως είναι καλό, γιατί ένα από τα βασικά προβλήματα της Ευρώπης είναι να θεσπίσει ισχυρούς δεσμούς, ισχυρούς δεσμούς, ισχυρότερους από ό,τι μέχρι τώρα, με τον εγχώρια πολιτική. Αν το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να επιχειρηματολογεί επί τη βάση του υπερεθνικού του χαρακτήρα, τότε τελικά το αποτέλεσμα θα είναι, φοβούμε, ότι ο κόσμος θα πει ναι, ναι, χρειαζόμαστε ένα βαθμό κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά δεν θα πρέπει να είναι το κοινοβούλιο προς χάρη του κοινοβουλίου, αλλά να είναι ένα κοινοβούλιο το οποίο να έχει ισχυρή σχέση με την χώρια ε, κατάσταση και πολιτική σκηνή. Κατά τη γνώμη μου, το Κοινοβούλιο αν επιμείνει σε κάτι τέτοιο θα βάλει μόνο του τρικλοποδιά στον εαυτό του. Δεν είναι λοιπόν προς το συμφέρον του Ευρωκοινοβουλίου να μείνει σε αυτή την ε, κλασική άποψη. Αλλά ξέρω πως υπάρχουν και πολύ ισχυρές αντίθετες απόψεις. Τελευταία παρατήρηση ότι το γερμανικό συνταγματικό δικαστήριο που συχνά αναφέρθηκε σήμερα το πρωί ανέφερε ότι η δημοκρατία είναι το δικαίωμα της ίσης εκπροσώπησης όλων των πολιτών. Αν θέλουμε, αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θέλουμε να πούμε πως ένα σώμα που αντιπροσωπεύει τις χώρες που δεν είναι στην Ευρωζώνη και έχει άποψη για αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για την Ευρωζώνη και να εφαρμοστούν ε, μόνο για την Ευρωζώνη, φοβούμαι πως αν ακολουθήσουμε κατά γράμμα τη λογική αυτή, δεν θα μπορέσουμε εύκολα να το δεχτούμε. Η συμβουλή μου λοιπόν προς το Κοινοβούλιο είναι να επιμείνετε για το τι είναι το πιο σημαντικό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει ισχυρός κοινοβουλευτικός έλεγχος για οποιοδήποτε μορφή διακυβέρνησης προκύψει για την Ευρωζώνη. Αν το τίμημα γι' αυτό είναι να υπάρξει ένα σύστημα κατά το οποίο από τη στιγμή που η Ευρώπη είναι διχασμένη στους ε, εντός και στους εκτός Ευρωζώνης και μόνο τα μέλη των χωρών εντός Ευρωζώνης συνδέονται με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, κατά τη γνώμη μου μπορεί να σταθεί αυτό συμβιβαστική λύση. Και ε, με αυτά θα κλείσω. Χωρίς μικρόφωνο ο Πρόεδρος, δυστυχώς. <laughs> Eh, Τώρα δίνω το λόγο στον καθηγητή Βέσελ που από το 1994 εργάζεται στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα αρχίσω στα γερμανικά, μη φοβάστε θα συνεχίσω αγγλικά όμως, γιατί ε, χρειάστηκε να γράψω το κείμενό μου στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχάς αλλά έχουν άμυκτα συναισθήματα στα αγγλικά. Δεν ξέρω μήπως ήταν κανένα δηλητηριασμένο δώρο αυτή η πρόσκληση, γιατί είναι ένα θέμα στο οποίο δεν έχω πραγματική απάντηση. Όπως είδαμε, η Διτεθνικά Κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είναι σε σύγκρουση μεταξύ τους ε, ε, για το ρόλο που πρέπει να παίξουν και αν υπάρξει κάποια μεικτή μορφή. Εγώ έχω τρεις αφετηρίες γι' αυτό. Πρώτον, δεν ξέρω αν είδατε το κείμενό μου, αναφέρθηκε και από τον κύριο Μανουηλίδη. Στην πρώτη μου σελίδα έχω μια γραφική παράσταση που είναι διδακτορικό μιας φοιτήτριά μου που πέρασε με πολύ καλό βαθμό γιατί είναι πάρα πολύ μεθοδική δουλειά ε, για να καταλάβει κανείς ποιος συμμετέχει πού, σε ποιο κύκλο λήψη αποφάσεων. Ποιος συμμετέχει με ποιο τρόπο και βλέπετε ήδη την περιπλοκότητα. Εμείς οι ίδιοι έχουμε τη ε, δυσκολία να ακολουθήσουμε και να παρακολουθήσουμε τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσει κανείς ε, οποιονδήποτε εκτός της Εθούσης ή εκτός άλλων ε, κύκλων εμπειρογνωμόνων της Ένωσης περί πρόκειται αυτό το νεφέλωμα. Από την άλλη, έχει αρχίσει από τη δεκαετία του 70 με το νομισματικό σύστημα και από ό,τι φαίνεται τα πράγματα λειτουργούν πάνω κάτω. Δεν υπάρχει και τεράστια επανάσταση. Ε, θα επανέλθω στο τέλος. Δηλαδή χρειαζόμαστε πραγματικά ριζικές αλλαγές. Και αν ναι, πώς και γιατί. Αυτή είναι η πρώτη εφετερία. Εφετερία δεύτερη αυτό το θέμα των, της πολυεπίπεδης κυβέρνησης ή των πολλών ταχυτήτων. Έτσι κι αλλιώς ακόμα περιπλέκει την κατάσταση. Άλλο είναι η μελέτη για το πολυεπίπεδο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ζήτησε και θα ε, έρθουμε σύντομα με τις απαντήσεις. Θα αναφερθώ στις ε, εμπειρικές ε, παρατηρήσεις και στις αναλύσεις. Το πολυεπίπεδο κοινοβούλιο ουσιαστικά δεν λειτουργεί και και απλή απάντηση γιατί δεν λειτουργεί. Και η τρίτη εφετηρία είναι ότι αυτό ακούστηκε στις ερωτήσεις ως πολιτικοί επιστήμονες πάντα σκεφτόμαστε την εξουσία. Έτσι, ε, κάπου εδώ κοντά είναι πάντα μακιαβέλη. Και η εξουσία δεν είναι μόνο η ομοιβία αλλά και το θέμα της νομιμότητας. Δηλαδή πώς τα κοινοβούλια ε, συνδέονται μεταξύ τους ε, με το συσχετισμό δυνάμεων. Τι είναι τα κοινοβούλια στη συνεργασία, είναι συμμαχία βουλευτών ή μήπως είναι σύγκρουση μεταξύ κοινοβουλίων. Και κοιτάζοντας αυτά που λέτε, ε, αγωνίστηκαν τα εθνικά κοινοβούλια και έχασαν κάποιες εξουσίες, άλλαξαν οι ε, οι συνθήκες με την κανονική ε, τακτική αλλαγή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε στη συντακτική συνέλευση, αλλά δεν συμμετείχε στην κύρωση. Και ποιο κυρώνει τα εθνικά κοινοβούλια. Όπω γίνεται και σε άλλε συνθήκε, πάντα τα εθνικά κοινοβούλια στι διακυβερνητικέ ε, κυρώνουν και όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα εκεί έχουμε ένα συσχετισμό δυνάμεων και ένα παιχνίδι εξουσία που μέχρι στιγμή είναι εξισορροπημένο προ τη μεριά των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, να σας αναφέρω λίγο τι ισχύει σήμερα, τι υπάρχει. Το γράφει ε, στο έγγραφό μου, ε, είναι η σπαζοκεφαλιά του Μοντεσκέ. δηλαδή πώς είναι αυτά τα πολλά επίπεδα και πολλές ταχύτητες. Υπάρχει ουσιαστική ισορροπία εξουσιών. Και δεν προβλημάτισε αυτό μόνο το Μοντεσκέ, αλλά είναι και ένα γενικότερο πρόβλημα και πολιτιστικό. Ξέρουμε το περίφημο ερώτημα. Α, ε, ε ξέρετε, στη Γερμανία λέμε ένα έκδοτο ότι έχεις για πινακίδες, η μία δείχνει Βερολίνο, η άλλη δείχνει Καλσρούι. Και ο κόσμος αναρωτιέται, αλλά ρωτάει, για πείτε μου, η κυβέρνηση δεν είναι ακόμα στο Βερολίνο, σωστά δεν το λέω. Ε, βλέπετε ότι ο κόσμος προβληματίζεται και ό,τι απόφαση παίρνει το δικαστήριο έχει μείζονε επιπτώσεις. Ε, και τι γίνεται ας πούμε με τα συνταγματικά ε, αιτήματα και τη ισορροπία των εξουσιών. Ξέρω ότι είναι πολλή δουλειά, έχουμε πολλές διδακτορικές διατριβές, αλλά τι γίνεται η Κόζα, κανείς δεν, δεν αναφέρθηκε, δεν άκουσα τουλάχιστον να αναφέρει κανείς την Κόζα σήμερα και δεν χρειάζεται να επεκταθώ, τα γνωρίζετε. Κοιτάξτε το πρωτόκολλο 1 για το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων και εκεί αναφέρεται κάτι για την Κόζακ που λέει «Α, ναι, θα μπορούσε να οργανωθεί η Κόζακ ε, η συνεργασία μόνη της». Ωραία. Ενδιαφέρον αυτό και ευχάριστο και μπορεί να ε, γνωμοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό χαριτωμένο είναι αλλά δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να λαμβάνονται υπόψη οι τη της ε, από κανέναν. Και ακούστηκε σήμερα το πρωί και το είπε και το δικαστήριο τη Καλσρούη ότι ε, αυτέ οι γνωμοδοτήσει τη ΚΟΖΑΚ δεν δεσμεύουν ούτε τα Εθνικά Κοινοβούλια ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι λίγοι οι συμμετέχοντες και δεν δεσμεύουν τα κοινοβούλια τους. Και αυτό είναι κατανοητό. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό το μείγμα έχει πάρα πολύ περιορισμένες δυνατότητες, αυτή η μεικτή δομή κοινοβουλίων δηλαδή. Ε, έχουμε το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, το άρθρο 13, ε, το, ε, πώς γίνονται τα κοινοβούλια εκεί, πώς συνδυάζουν οι διάφορες επιτροπές. Εγώ βάσει της παλιάς εμπειρίας λέω ότι δεν βγαίνουν πολλά και έρχομαι στη βασική ιδέα, την κεντρική ιδέα της ανάλυσης συζητούμε ε, την λογική λύση, την ορθολογική λύση, γιατί θα πρέπει η πολιτική και τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσουν σε μια τέτοια συνεδρίαση επιτροπής και να πάνε. Δεν, δεν είναι μόνο πρόβλημα ημερομηνία. Εντάξει, αυτό μπορούμε να το λύσουμε. Το θέμα είναι τι θα βγει από εκεί. Ωραία, μια ευχάριστη ανταλλαγή απόξε θα έχουμε. Γυρνάει ο καθένα σπίτι του και δεσμεύεται από το κόμμα του, από το κοινοβούλιο του, από το δικαστήριό του, ενδεχομένω το ίδιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει και πίεση των πολιτικών ομάδων. Οπότε γιατί να πάει κανεί σε ένα τέτοιο φόρουμ και αν πάει τι θα βγει από εκεί. Ωραία δήλωση, θα δημοσιευθεί κιόλα και Μοιάζεται. Ε, αδιαφορία πλήρης. Ξέρω ότι είναι πολύ ισχυρά αυτά που λέω, αλλά είναι βάση της εμπειρίας και αυτή είναι η προσέγγιση μου. Έρχομαι λοιπόν τώρα στις επιλογές. Αν αυτή είναι η λύση, μικτές δομές κοινοβουλευτική συνεργασίας λέμε δεν λειτουργούν γιατί δεν έχουν καμία εξουσία και δεν υπάρχει και κανένα κίνητρο για τους βουλευτές να συμμετέχουν. Ωραία, πώς μπορούμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Ε, το θέμα θα είναι ε, υπάρχει κανένας τρόπος αλλαγής των εξουσιών αυτής της μικτής συνέλευσης δομής των μικτών ε, ομάδων. Αυτό είναι βέβαια συνταγματικό θέμα και θεσμικό. Ο Ζισκάρη είχε προτείνει και στη συντακτική συνέλευση να γίνει ένα συμβούλιο λαών, το κογκρέσο, που πούμε το λένε οι Γάλλοι αυτό. Ε, ο πρόεδρος του Συμβουλίου να προεδρεύει. Ο κύριος Φαρόμπα είπε όχι. Δεν θέλει να το εγκλέγουν αυτοί και παρά μόνο οι ομόλογοι του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ε, να συζητάει την έκθεση του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση στην Ένωση. Ωραία. Ε, κάναμε συντακτική συνέλευση, μην το ξεχνάμε και αυτό, και νομίζω ότι ήταν αρκετά χρήσιμη και βοήθησε. Αλλά και πάλι, όπως είδαμε στη γαλλική και την ολλανδική περίπτωση, οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί δεν ήταν αρκετά ισχυροί για να πείσουν τους λαούς τους να δεχτούν το Σύνταγμα ή τη Συνθήκη. Αλλά η συντακτική συνέλευση μπορεί να είναι καλή για τροποποίηση των συνθήκων, όχι για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Ο Γιώ Λάινεν είπε επίση ότι μπορεί να έχουμε ενδεχομένω ένα μικρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα μικρότερο σχηματισμό, δηλαδή να συμμετέχουν μόνο οι 17-25 της Ευρωζώνης ή της Συμφωνίας του Συμβάνου θα μπορούσε να είναι αυτή η ενδιαφέρουσα λύση αλλά και πάλι νομικός δεν είμαι αλλά δεν βλέπω την νομική ε, διάσταση ε, και πώς θα, θα ευσταθεί αυτό σε νομική βάση ε, ή πρέπει και πάλι να αλλάξει συνθήκη. Αυτές είναι μερικές από τις επιλογές που ανοίγονται μπροστά μας. Και αν ξεκινήσουμε από την αφετηρία που σας λέγω, δηλαδή η σημασία να έχει κανείς νομική ισχύ, λύση δεν βλέπω. το λέω και στους συναδέλφους και τους φίλους που με γνωρίζουν. Πάντα έχω να κάνω προτάσεις, αλλά εδώ τι να κάνω, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Έχω κολλήσει λίγο. Αν αρχίσουμε από την ανάλυση ότι μόνο οι βουλευτές θα συμμετέχουν, αν υπάρχει εξουσία, η εξουσία είναι δύσκολη. Γιατί χρειάζεται αλλαγή και των συνθήκων, αλλά και τους κανονισμούς των Εθνικών Κοινοβουλίων. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε κολλήσει. Επανέρχομαι στο Μοντεσκέ βέβαια, έχουμε ε, ομοσπονδιακά συστήματα όπου υπάρχει ε, αυτή η συνοχή. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το κλασικό ομοσπονδιακό σύστημα Ηνωμένε Πολιτείε με ελέγχους και αντίβαρα. Τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχει μια ε, εγγενή σύγκρουση. Ε, κοιτάξτε την ιστορία των ΗΠΑ. Πολιτειών. Ε, ξέρετε ότι ο πρόεδρο συγκρούεται με τον Κογκρέσο, τα δύο σώματα του Κογκρέσου μεταξύ τους. Ε, είναι ένα οι συγκρούσει, οι οποίε δεν λύγονται, δεν, λύνονται με συνταγματικά μέσα, ούτε με, με ένδικα μέσα, αλλά με τρόπο που προβλέπει το Σύνταγμα. Κάπως έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε και εμείς, γιατί δεν βλέπω πολιτικά και συνταγματικά βιώσιμη λύση άλλη καμία εδώ έχουμε ένα μείζον κόστο που συνδέεται. Δηλαδή να μην λέμε τύχες Γιάννη τύχα πάντα, μια χαρά γαλά είμαστε. Ε, αλλά και γιατί να μπαίνουμε και στον κόπο. Γιατί αυτό που είπε ο Γιάννης ε, είναι σημαντικό και για τα Εθνικά Κοινοβούλια και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο καθένας μιλάει στο εθνικό πλαίσιο, έχει εθνικές απόψεις στο μυαλό του και πολλές φορές αυτά τα χαρακτηρίζω εγώ επαρχιώτικα. Είπατε ότι είμαι καθηγητής στην Κολονία, πηγαίνω έρχομαι και Βρυξέλλες και Βερολίνο συχνά και παντού ακούω τελείως διαφορετικές αντιλήψεις για το τι εστί η Ευρώπη. Ε, μια μικρή πόλη, μεσαία πόλη, έχει διαφορετική αντίληψη από ότι η Βρυξέλλες και ακόμα πιο διαφορετική έχει το Βερολίνο. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα για το μέλλον. Θα πρέπει να έχουμε πολύ πιο βαθιά ανταλλαγή απόψεων για να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, μια συναντήληψη. Αφού δεν έχουμε κοινή δράση, communauté d'action στα γαλλικά, να έχουμε τουλάχιστον communauté de vue, να έχουμε την ίδια άποψη ε, για ορισμένα πράγματα. Μπορεί ε, για να καταλαβαίνουμε γιατί άλλοι λειτουργούν με κάποιο τρόπο που θεωρούμε εμείς παράλογο. Να καταλαβαίνουμε ότι έχουν τη λογική τους και αυτή και όχι ότι είναι απλώς ηλίθιοι. Ας πούμε για το πώς δράει η Γερμανία, ε, διαβάζουμε, οι εκτός Γερμανίας θεωρούν ότι οι Γερμανοί είναι τελείως ανόητοι. Και τούμπαλιν, αυτό φρονούν οι Γερμανοί για άλλα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει καν κατανόηση, ε, όχι συνεννόηση, ούτε καν κατανόηση ε, για το τι πιστεύει ο καθένας και πώς βλέπει τα πράγματα. Πρόεδρε, εγώ δεν έχω μαγική λύση. Θέτω ερωτήματα κι εγώ. Ε, δεν ξέρω. Η εύκολη λύση να είναι οι μεικτές συνεδριάσεις δεν μου φαίνεται η πιο ενδεδειγμένη ε, ούτε στα Εθνικά Κοινοβούλια ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ας το προσπαθήσουμε, δεν λέω, αλλά δεν πιστεύω ότι θα αποδώσει ούτε θα ξεπεράσει το βασικό ε, χάσμα ε, μεταξύ ε, των συζητήσεων που γίνονται στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά, ευχαριστώ όλους όσους παρενέβησαν και ευχαριστώ και τους διερμηνείς που έμειναν στις θέσεις τους ακλόνητοι παρότι ξεπεράσαμε τα ωράρια. Ε, θα τα πούμε λοιπόν το απόγευμα, θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που έχουν προβλεφθεί για την τρίτη σύνοδο και έπειτα θα συζητήσουμε για τις πέντε αυτές παρεμβάσεις. Γεια σας.